Okay, colleagues. Γεια σας συνάδελφοι. Θα πρότεινα να αρχίσουμε. Καλωσορίζω όλους τους παρόντες. Καταρχάς κάποια διαδικαστικά. Σήμερα δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε διερμηνία από και προς όλες τις γλώσσες. Δεν έχουμε λοιπόν δανικά, φιλανδικά, λετονικά, μαλτέζικα και κροατικά, γιατί δεν υπάρχουν αρκετές καμπίνες σε αυτή την αίθουση. ζητώ συγγνώμη και ελπίζω να μπορείτε να ακούσετε κάποια άλλη γλώσσα. Έχουμε σήμερα λοιπόν τρεις ενότητες ε, στη Επιτροπή μας. Το πρώτο είναι τα προγράμματα παρακολούθησης των Ηνωμένων Πολιτειών και ε, ε, ο αντίκτυπός τους ε, στην ιδιωτική ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένε Πολιτείες. Η δεύτερη ενότητα αφορά το ρόλο της κοινοβουλευτικής εποπτείας των μυστικών υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο, ενώ η τρίτη ενότητα θα ασχοληθεί με τα ε, προγράμματα ηλεκτρονικής μαζικής παρακολούθησης της NSA και το ρόλο των εταιριών τηλεπικοινωνιών. Αρχίζουμε λοιπόν από τα προγράμματα παρακολούθησης των Ηνωμένων Πολιτειών και με πολύ μεγάλη χαρά καλωσορίζω ενώπιόν μας τον κύριο Jim Sensenbrenner, που κάθεται εξ ευωνίμων του Κλοντ Μωράη, είναι μέλο της Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, μέλο μέλος της Δικαστικών Υποθέσεων και, πιο σημαντικό για τη σημερινή μα συνεδρίαση, πρόεδρο της Υποεπιτροπής για το έγκλημα, την τρομοκρατία, την εσωτερική ασφάλεια και τι έρευνε. Και ένα από του δύο σπόνσορες για να το χαρακτηρίσω έτσι, ε, ενός νέου νομοσχεδίου που προτείνεται, το ε, Freedom Act, νόμος περί ελευθεριών, ε, διότι η κατάσταση έχει ξεφύγει με το νόμο Patriot Act έγινε μια ε, πρώτη επαφή της αντιπροσωπείας μας 29 Οκτωβρίου με τον κύριο Σένσεν Μπρένερ και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε σήμερα απόψε εδώ στις Βρυξέλλες για πολύ καιρό πραγματικά ε, είχαμε νιώσει μια απογοήτευση γιατί μόνο στην Ουάσιγκτον μπορούσαμε να τους βλέπουμε τους συνομιλητές μας και τους εταίρους Είναι πολύ σημαντικό να λέμε ότι ε, διατλαντική συνεργασία θα πρέπει να λαμβάνει η χώρα όχι μόνο σε επίπεδο κυβερνήσεων αλλά και σε επίπεδο εκλεγμένων εκπροσώπων όπως είναι ε, και τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένε Πολιτείες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι αυτός ο κοινοβουλευτικός πυλώνας, αν θέλετε, της διατλαντικής συνεργασίας. Τι έγινε, η NSA έχει υπερχίσει και παίζει και με τα φώτα εδώ. Ελπίζω λοιπόν να μην είναι μοναδική αυτή η ευκαιρία με την, έννοια της άπαξ ε, συνάντησή μας, αλλά να έχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα συνεργασία και συναντήσεις, διότι έχω την αίσθηση ότι ε, είναι πολλά τα θέματα που μας ενώνουν και μπορούμε να προβλέψουμε και ενδεχομένως μελλοντική συνεδρία σε επόμενη σε ένα εξάμεινο ή κάτι τέτοιο. Ε, θα ήθελα να δώσω λοιπόν το λόγο στο ε, κύριο Σέντζενμπρένερ για να μας παρουσιάσει την πρότασή του για το νόμο σχέδιο ε, Freedom Act μαζί με τον κύριο Πάτρικ Λέι την έχει ε, εκπονήσει. Ορισμένοι το γνωρίζετε από προηγούμενες επισκέψεις στην Ουάσιγκτον. Το Freedom Act είναι πολύ ενδιαφέρον για μας γιατί θα εμποδίσει την NSA να συλλέγει μαζικά ε, στοιχεία ε, των τηλεπικοινωνιών των Αμερικανών ε, τροποποιώντας τη διαβόητη ενότητα το τμήμα 215 του Patriot Act επίσης θα κάνει πολλές αλλαγές στη ΦΑΙΣΑ και στην διαγόμενη ε, μυστική δικαιοσύνη και μυστικές αποφάσεις δικαστηρίων. Εν πάση περιπτώσει αυτά εισαγωγικά θα ακούσουμε περισσότερα από τον ίδιο τον κύριο Σένσεν Μπρένερ. Θα μας παρουσιάσει την πρόταση λοιπόν για το νόμο Freedom Act. Θα ακολουθήσουν ερωταποκρίσεις. Πρώτα θα ρωτήσουν ε, ο εισηγητής Κισκιώδης και μετά τα υπόλοιπα μέλη. Κύριε Έγκστρομ, τι θέλετε διαδικαστικό. Ναι, θέλω να πω ότι μου είπαν οι βοηθοί μου τώρα ότι το web streaming δεν βγάζει ήχο. Μήπως θα μπορούσατε να το βελτιώσετε, να το διορθώσετε κύριε Πίρκερ, θέλετε διαδικαστικό, όχι. Ζητάτε το λόγο από τώρα και εσείς κυρία Ζήπελ, μάλιστα. Κύριε Σένσεμπέρνα, έχετε το λόγο. Very much, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόσκληση να σας ε, παρουσιάσω εδώ το νόμο. Ήμουν ε, πρόεδρος της Επιτροπής Δικαστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών όταν ε, ασκήθηκε η επίθεση της 10ης Σεπτεμβρίου. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε νέους μηχανισμούς και ευρύτερε εξουσίες για να αποτρέψουμε εκείνους που ήθελαν να μας βλάψουν, αλλά που δεν ήθελαμε θέλαμε να επιτρέψουμε αδιάκριτα την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας να κρυφοκοιτάει στη ζωή αθών πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Ως πρόεδρος λοιπόν Προσπάθησα με στενοχρονοδιάγραμμα να βρω την ισορροπία μεταξύ πολιτικών ελευθεριών και της εθνικής ασφάλειας στο πάτριο τάκτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, το τελικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε στην Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων Ομόφωνα και με υπερκομματική υποστήριξη. Πιστεύω ακράδαντα ότι το Patriot Act ε, θα σώσει ζωές, ε, βοηθώντας ε, τις μυστικές υπηρεσίες να εντοπίσουν και να αναχαιτήσουν δυνάμει τρομοκράτες. Αλλά δυστυχώς η NSA το τελευταίο καιρό εξασθένησε Έπληξε παρεμήνευση και αγνώριζε τι πολιτικέ ελευθερίε που προστατεύονται από το όνομα αυτό. Ο πρόεδρο Ρόναλτ Ρίγαν είπε: Πίστευε και ερεύνα. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου ε, και με ε, τι Ηνωμένε Πολιτείε ε, στα πρόθυρα του τη σημαντικότερη σύγκρουση μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, το Κογκρέσο διεύρυνε τις, εκτελεσ... τις εκτελεστικές εξουσίες για να προστατεύσει τον Αμερικανικό λαό. Αλλά δυστυχώς έγινε κατάχρηση των εξουσιών αυτών από την NSA. Ε, ε, αγνοήθηκαν οι εργοδός ε, εκπονηθήσεις διατάξεις των νομοθετών και η NSA περιχαρακώθηκε γύρω από ένα πυκνό σύννεφο μυστικότητας και διαφάνειας και έτσι δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε το κατά πόσο έλαβαν χώρα οι υποσχεθήσεις μεταρρυθμίσεις. Και μάλιστα η χιονοστιβάδα αποκαλύψεων ε, μου δημιουργήσε έκπληξη και αποτροπιασμό, όπως και σε πολλούς Αμερικανούς και ε, συμμάχους μας. Γι' αυτό και μαζί με τον ε, γερουσιαστή Πάτρικ Κλήχη, που είναι ο, ο πρόεδρος της ε, αντίστοιχης επιτροπής της Γερουσίας προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη της παγκόσμιας κοινότητας και να περιορίσουμε τις καταχρήσεις. Γι' αυτό θέλουμε ένα νέο νόμο με την ενίσχυση των δικαιωμάτων, το σταμάτημα των παρακολουθήσεων, την αδιάκριτη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση μέσω online, ε, παρακολούθηση online. Ε, θέλουμε λοιπόν να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των πολιτικών ελευθεριών και της ασφάλειας. Ο νόμος αυτός ήδη έχει προκαλέσει την ε, γενική υποστήριξη 100 ε, συγχορηγών και στο Κογκρέσο και σε πολλές ομάδες και ενώσεις πολιτικών ελευθεριών όπως την ACLU και την NRA. Επίσης μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Google, η Apple, η Facebook και η Microsoft έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους και σημαντικά διοικητικά συμβούλια εφημερίδων όπως το New York Times, Los Angeles Times, Milwaukee Journal Sentinel και Washington Times. Και παρά τις ε, αντίστοιχες προτάσεις των ε, μυστικών υπηρεσιών θα έχουμε πραγματικές ε, μεταρρυθμίσεις γιατί έχουμε ξεκινήσει με σφοδρή συζήτηση για το πώς συγκεντρώνονται οι πληροφορίες και από πού. Τον Οκτώβριο του, της 31 Οκτωβρίου με ψήφο 11 προς 4 Επιτροπή για τις Μυστικές Υπηρεσίες του ε, της Γερουσίας για πρώτη φορά στην ιστορία της ε, χώρας μας ε, ψήφισε το, την, το να, εξουσιοδετεί την αδιάκριτη κατασκοπία προς τον Αμερικανικό λαό. Εγώ πρεσβεύω διαφορετική προσέγγιση. Με το Freedom Act ε, και τα Patriot Act ε, θέλουμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία, να βρίσκουμε δεδομένα, αλλά όταν υπάρχουν ε, βάσιμες υπόνοιες ότι κάποιος έχει διασυνδέσει με την τρομοκρατία. Αλλά δεν επιτρέπεται πια η αδιάκριτη συλλογή δεδομένων και μάλιστα για αθώους ανθρώπους. Και μάλιστα άλλες μεταρρυθμίσεις για τον νόμο για την εποπτεία και την παρακολούθηση ξένων μυστικών υπηρεσιών θα αποτρέψουμε άλλες καταχρήσεις των νομοθετικών διατάξεων που δυστυχώς έχουν διαπραχθεί από τις μυστικές υπηρεσίες κατά των Αμερικανών και των ξένων. Όπως ε, είπε ο Λουίς Πράντα από το Αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο, το διάχυτο φως είναι το καλύτερο απολυμαντικό. Γι' αυτό θα πρέπει ε, να διευρύνουμε τη διαφάνεια και να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε τη λογοδοσία της NSA. Γιατί ε, ακόμη και οι σημαντικότερες ακόμη και σημαντικότεροι περιορισμοί μπορούν να καμφθούν. Γι' αυτό με τη διαφάνεια θα αποκαταστήσουμε την, ε, τον καλύτερο έλεγχο. έχουν, βέβαια το Κογκρέσο έχει περιορισμένη εξουσία να σταματήσει η παρακολούθηση ξένων ηγετών όπως της Άγγελας Μέρκελ. Ο πρόεδρος Ομπάμα είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για αυτή την παρακολούθηση, την παρέμβαση. Ε, ε, πιστεύω ότι το καλύτερο επιχείρημα για τη μεταρρύθμιση είναι όταν ε, ακούγεται το επιχείρημα ότι ο μόνος ε, άνθρωπος που μπορούσε να επιτρέψει τις καταχρήσεις δεν γνώριζε για αυτές. Αλλά ακόμη και όταν οι καταχρήσεις γίνονται πέραν των αρμοδιοτήτων του Κογκρέσου, δεν μπορούμε να υποτιμούμε τη συμβολική αξία μιας γνήσιας μεταρρύθμισης. Αν επιτύχουμε στο Freedom Act των ΗΠΑ, θα έχουμε την πρώτη ουσιαστική ε, πρωτοβουλία μετά την 10η Σεπτεμβρίου να περιορίσουμε την παρακολούθηση το σημαντικό μήνυμα είναι ότι οι αθώοι άνθρωποι θα πρέπει να τους μεταχειριζόμαστε σαν τρομοκράτες και το κράτος δικαίου δεν είναι ούτε πολύ ευέλικτο αλλά ούτε και πολύ επίκες. Θα πρέπει επίσης να ερμηνεύεται σωστά το Freedom Act. Οι παρελθούσες καταχρήσει δεν πρέπει να επαναληφθούν και να προστατεύονται οι πολιτικές ελευθερίες των Αμερικανών πολιτών. Γιατί τους τελευταίους μήνες είχαμε όλο και περισσότερες καταγγελίες και δημόσια κατακραυγή. Γι' αυτό με τον Πρόεδρο Λί θα προωθήσουμε αυτή τη σημαντική νομοθετική πρόταση ε, και στο Κογκρέσο για ψηφοφορία οι πολιτικές ελευθερίες ε, ε, εξασφαλίζονται εφόσον θα προσπαθήσουμε να τις προασπίσουμε. Και μαζί με τους συναδέλφους από το Κογκρέσο θα προωθήσουμε αυτή την νομοθεσία για να προσπίσουμε τα δικαιώματα των Αμερικανών και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στις μυστικές μας υπηρεσίες. Και όταν μιλώ για εμπιστοσύνη θα ήθελα να πω ότι αυτές οι αποκαλύψεις έχουν ε, βάλει ουσιαστικά την εμπιστοσύνη, έχουν λαβώσει την εμπιστοσύνη που δημιουργήθηκε από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ ε, Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Και η εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμάχων είναι πολύ σημαντική, γιατί σύμμαχες είναι οι χώρες μας και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα είμαστε κινητήριοι μοχλή τη παγκόσμια οικονομία. Θα πρέπει όμω ταυτόχρονα να είμαστε και υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών σε όλε τι δημοκρατικέ χώρε. Η διεθνή συνεργασία είναι πολύ σημαντική για να αναχαιτιστεί η τρομοκρατία. Αλλά και η εμπιστοσύνη θα πρέπει να είναι ακέραιη. Και ζητώ από τους φίλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συνεργαστούν ρεαλιστικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με ισορροπημένες προσπάθειες να προστατεύσουμε τα έθνη μας. Μόνο από κοινού θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη προστατεύοντας ταυτόχρονα τις πολιτικές ελευθερίες και στις δύο όχθες του Ατλαντικού. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και με πολύ χαρά θα απαντήσω και σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Σένσελ Μπρένερ. Ανοίγει λοιπόν η συζήτηση, ερωτήσεις. Μέχρι τις 4 η ώρα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Εκτός από τον εισηγητή και τους κοιόδης έχουν ζητήσει το λόγο και άλλοι δύο συνάδελφοι, συν δύο που βλέπω τώρα. Κλείνει ο κατάλογος. Um, I'm going to first... Προς το παρόν. Ε, θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Μωράες ένα δίλεπτο έκαστος, ερώτηση, απάντηση, ερώτηση, απάντηση, έτσι θα πάει. Ευχαριστώ ε, κύριε Γερουσιαστά που ήρθατε σήμερα και που μας υποδεχτήκατε και στην Ουάσιγκτον. Ήσασταν ε, μια σημαντική παρουσία λέγοντάς μας ότι η NSA θα μπορούσε να μας μιλήσει και να μας δώσει κάποιες με τις πληροφορίες που ζητάμε. Τώρα θα μπορούσατε να μας πείτε λεπτομερέστερα Πόσο νομίζετε ότι οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπουν οι ΗΠΑ θα είναι εφικτές και ρεαλιστικές και κατά πόσον πιστεύετε ότι θα υπάρξει διεθνής αντίκτυπος ιδίως στην Ευρώπη, ιδίως για τη μαζική συλλογή δεδομένων, την χίδιν συλλογή μάλλον. Θα μπορούσατε να περάσετε σε λίγες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Έπειτα, σε σχέση με τα αποδεκτικά στοιχεία που έχουμε λάβει ως τώρα, είναι προφανές ότι το νομικό πλαίσιο και το συνταγματικό σύστημα των ΗΠΑ το καθιστούν πολύ δυσχερέ να επεκταθεί η προστασία περιοδικού βίου και σε πολίτε εκτό Ευρωπαϊκή, εκτός ΗΠΑ. Τι στήριξη λοιπόν θα υπάρξει από το Freedom Act ώστε να μπορέσει να προστατευτεί και αυτό το μέρο των πολιτών που μπορεί να μείνει εκτός ΗΠΑ, των Ευρωπαίων, ώστε να εξομαλυνθούν οι σχέσει μας προ αυτό. Και μια τελευταία ερώτηση σχετικά. Οι συμφωνίε Ευρωπαϊκή Ένωση ΗΠΑ που ισχύουν ε, παρακολουθούνται από ε, την εκτελεστική εξουσία. Υπάρχουν ε, στο Κογκρέσο σκέψεις να ξανακαταστεί αυτό Εδώ ε, η Επιτροπή που ασχολείται με τα θέματα αυτά κοιτάζει τις ε, σχέσεις με τις, τις εξωτερικές μας σχέσεις. Το Κογκρέσο... Εδώ πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσον μπορεί να δεσμευτεί σε μια πορεία ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Θα είναι δύσκολο, σχεδόν αδύνατο να τον υποχρεώσουμε διότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει ερμηνεύσει το Σύνταγμά μας και τη συνταγματικό διαχωρισμό των εξουσιών ως προς την προστασία των Ευρωπαίων πολιτεών. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πράγματι η νομοθεσία σε ό,τι αφορά τη μαζική συλλογή δεδομένων δεν ορίζει κάτι με σαφήνεια, όμως επιτρέπει η μαζική συλλογή δεδομένων να πραγματοποιείται. Και αυτό αφορά και αυτήν την ε, πλευρά του Ατλαντικού, αλλά και την απέναντι. Θα χρειαστεί βεβαίω να υπάρχει διαρκής και εντατική εποπτεία. Και καλώ το συζητάμε το σήμερα αυτό, διότι για την ώρα είδαμε ότι η δικαστική και εκτελεστική εξουσία των ΗΠΑ, αυτό αυτά τα σκέλη της κυβέρνησης, δεν, δεν επιτήρησαν σωστά την NSA. Ε, αυτό το είδο λοιπόν η εποπτεία θα πρέπει να είναι λίγο πιο αυστηρή, αρκετά πιο αυστηρή και να φέρει και αλλαγέ να αλλάξει η πολιτική τη NSA όταν τεθεί σε ισχύ ο σχετικό νόμος. Καλώ, ευχαριστώ. Σκιώδη του ΕΛΚ ποιο είναι, απουσιάζει Δυστυχώ. Έχω γράψει τον εαυτό μου στο τέλο ε, του καταλόγου. Θα δώσω τότε το λόγο στον κύριο Άρμπεχ των Πρασίνων. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Σένσεν Μπρένερ που ήρθε μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ καλό μήνυμα ε, και μας ενθαρρύνει και μας βοηθάει να κάνουμε και τη δουλειά μας που είναι ε, ερευνητικής φύσεως για τις δραστηριότητες ε, κατά τα άλλα κατέρωθεν του Ατλαντικού, όχι μόνο στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και επίσης γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές κόκκινες γραμμές που έχουν ξεπεραστεί και στα κράτη-μέλη και στους θεσμούς των κρατών ε, των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο ας πούμε. Εσείς πώς βλέπετε τη διασύνδεση όλων αυτών, γιατί μιλάτε για το διαχωρισμό ως προς την εξωτερική πολιτική. Αυτό που μας απασχολεί εμάς όμως είναι ε, ένα θέμα εσωτερικής πολιτικής που έχει και διεθνείς επιπτώσεις ως προς διεθνείς σχέσεις. Πώς, ας πούμε, αξιολογείτε την αδιάκριτη συλλογή στοιχείων ε, Αμερικανών πολιτών ε, στην Ευρώπη και πώς ε, θα τερματιστεί αυτή η τήρηση αρχείου, αν θέλετε, αυτό το στοιχείο. Πώς ε, τα συζητά αυτά το Κογκρέσο. Κοιτάξτε, καταρχάς επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν θα υπάρχει χήμα μαζική συλλογή, ούτε αδιάκριτη τήρηση των στοιχείων αυτών. Δεν μιλάμε λοιπόν για το ίδιο πράγμα ακριβώς. Τώρα, αν θα υπάρξει μία επαόριστο διατήρηση των στοιχείων αυτών στην νομοθεσία Freedom Act, αυτό έχει να κάνει με το αν υπάρχουν υποψίες ε, ενοχής ή συμμετοχής σε τρομοκρατική δραστηριότητα. Ε, αυτό είναι θέμα των διοκτικών αρχών και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και ε, άλλων κρατικών υπηρεσιών. Εδώ περισσότερο μιλώ για τα κράτη-μέλη και όχι για την Επιτροπή θα πρέπει τα στοιχεία να διατηρούνται ε, εφόσον ε, υπάρχει στοχευμένη αντιτρομοκρατική έρευνα ε, επί συγκεκριμένων προσώπων. Διατηρούνται τα στοιχεία τους. Ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οτιδήποτε γίνεται θα πρέπει να είναι ενός, βάσει συνταγματικού πλαισίου ε, σε ό,τι μας αφορά ε, εντός του συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών και εδώ στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια των εκάστοτε συνταγμάτων αλλά και των συνθήκων που ορίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και διέπουν και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν συνταγματικές εγγύησεις. Εάν αυτές ε, παραβιάζονται ή ε, αγνοούνται, πράγμα που πιστεύω ότι έχει κάνει η NSA, ε, πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τώρα το χρονικό ορίζοντα, μέχρι πότε θα τηρούνται αυτά τα στοιχεία, πρέπει να σας πω ότι ούτε ο λευκός ήχος, ήχος ούτε η ηγεσία της γερουσίας ή της βολής αντιπροσώπων, ούτε οι υπηρεσίες πληροφοριών ικανοποιούνται ή χαίρονται με την νομοθεσία που προτείνουμε ο γερουσιαστής ε, λίγη και ε, εγώ. Ακόμα και ο πρόεδρος ε, Μπένερ της Βουλής των Αντιπροσώπων θέλουν να προωθηθεί αυτό και πότε θα γίνει η σύγκρουση αυτή όταν θα μας φέρουν το λογαριασμό οι μυστικές υπηρεσίες, τον προπολογισμό τους, θα προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε ε, τον προϋπολογισμό τους και πραγματικά μπορούμε να το κάνουμε και στη Βουλή και στη Γερουσία. Ή μπορούμε και να απορρίψουμε τον προϋπολογισμό τους. Οπότε η ε, απέναντι πλευρά θα κάνει ε, πολύ γρήγορα τα όσα πρέπει να κάνει. Εμείς ξέρουμε τι πρέπει να γίνει ε, και στην νομοθεσία και ο γερουσιαστής λέει που είναι από την αριστερή πτέρυγα και πολύ του ε, πολιτικού φάσματος και εγώ που είμαι από τη δεξιά και πολύ του πολιτικού φάσματος. Οι επόμενοι που έχουν ζητήσει το λόγο δεν είναι παρόντες. Εγώ θα είμαι τελευταία σκιώδηση συγγήτρια και μετά οι υπόλοιποι που ζήτησαν το λόγο. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που αναφερθήκατε στην αριστερά και στη δεξιά του πολιτικού φάσματο πάντα μας ε, παρηγορεί ότι μπορούμε πάντα να επιστρέφουμε κατέρωθεν στις κοινέ δημοκρατικές αξίες και χαίρομαι που υπάρχει ε, αυτή η προσέγγιση. Κατανοώ ότι ε, υπάρχει η μέρημνα της ασφάλειας στην Αμερική, αλλά πολύ συχνά είναι και πρόσχημα για ασυδοσία των υπηρεσιών ασφαλείας. Και πολλοί συνάδελφοι φαντάζομαι έχουν δει τι γίνεται με τις παρακολουθήσεις. Δηλαδή όταν ε, ακούτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Μέρκελ ή ε, κάποιον ε, άλλον ηγέτη. Αυτό πώς μπορεί να σας βοηθήσει στην αντιτρομοκρατική σας προσπάθεια. Πολύ συχνά στο παρελθόν η ασφάλεια γίνεται αντικείμενο κατάχρησης διαφόρων εξουσιών για λόγους πολιτικούς. Και τώρα νομίζω ανησυχούμε και οι δύο για αυτά τα ζητήματα, αντίστοιχα θέματα μαζικής ε, παρακολούθησης. Και η ρωσική κυβέρνηση χρησιμοποιεί κάτι αντίστοιχο, ένα πρόγραμμα ε, με πρόφαση ε, την τρομοκρατία και την ασφάλεια, αλλά μάλλον για ε, πολιτικούς σκοπούς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι αντίστοιχο με τον Κλώτ Μωράες. Εσείς βλέπετε καμιά πιθανότητα τελικά να συμπλησιαστούν τα εχέγγυα ασφαλιστικής δικλέδε και τα δικαιώματα ε, των αλλοδαπών πολιτών σε σχέση με τους Αμερικανούς. Έχω και άλλες ερωτήσεις. Νομίζω την άλλη εβδομάδα ε, στην Ουάσιγκτον θα γίνει μια συνάντηση. Η Επίτροπος Ρέντινγκ ε, θα συναντήσει τον Έρικ Χόλντερ, το Γενικό Εισαγγελέα και Υπουργό Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχω ιδέα τι θα συζητήσουν, ελπίζω να υπάρξει μια αναγνώριση ότι θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη μεταχείριση, είτε είσαι Αμερικανός πολίτης, είτε είσαι πολίτης τρίτης χώρας. Απαντώ εδώ σε αυτό που λέτε με διαφορετικό τρόπο. That's, Εντάξει, θετική απάντηση. Έχω δύο ακόμη σύντομε ερωτήσεις. Άκουσα προσεκτικά αυτά που είπατε. Οπότε το δικαστήριο αυτού του νόμου για την παρακολούθηση των ξένων μυστικών υπηρεσιών ε, μάλλον ε, είπατε ότι θα αφήσετε έναν περισσότερο ειδικό επόπτη από το να καταργήσετε αυτό το δικαστήριο ΦΙΣΑ, ΦΑΙΣΑ. Πώς θα ενισχύσετε τα εχέγγυα που προτείνετε και με ποιο τρόπο μπορούμε να συνεργαστούμε για να σας βοηθήσουμε να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες σας και ενδεχομένως ε, να έχουμε και μια διατηλαντική κοινή πρωτοβουλία για να αποτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι η ανταλλαγή μυστικών πληροφοριών είναι θεμελιώδου σημασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Γιατί μερικές πληροφορίες μπορούν να συγκεντρωθούν από εσά ε, και δεν γίνεται από εμά ε, ε, και σίγουρα η συγκέντρωση αυτών των στοιχείων είναι σημαντικό για να αναχαιτιστεί ή να αποσοβηθεί μια τρομοκρατική απόπειρα. Και αν είχαμε τέτοια καλή συνεργασία ή ανταλλαγή, θα είχαμε αποτρέψει και την 10η ε, Σεπτεμβρίου. Και τέτοιου είδου συνεργασία μεταξύ μυστικών υπηρεσιών γίνεται σχετικά εύρυθμα και μεταξύ των αστυνομικών αρχών και μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών. Αυτή η αγαστή συνεργασία θα πρέπει να συνεχιστεί μεν, αλλά υπό έλεγχο, υπό εποπτεία. Και αν δεν έχουμε πανομοιότυπα νομικά πλαίσια, τουλάχιστον έχουμε παρόμοια νομικά πλαίσια. Σε ό,τι αφορά το δικαστήριο ΦΑΙΣ αυτή τη παρακολούθηση ξένων μυστικών υπηρεσιών και του σχετικού νόμου, το Freedom Act προβλέπει πολλά πράγματα. Δεν έχει τον ειδικό επόπτη για την ιδιωτική σφαίρα, αλλά είχαμε ένα δικαστή που πρότεινε κάτι τέτοιο και μάλιστα συμμετείχε στο ε, δικαστήριο Φάσα γιατί μόνο ακούγαμε ε, τα σχόλια του Υπουργείου ε, Δικαιοσύνης και της NSA. Αλλά εμείς θέλουμε να ακούμε και τις δύο εμπλεκόμενε πλευρές προκειμένου να συγκεντρώσουμε τα διάφορα στοιχεία και να καταλήξουμε σε αποφάσεις. Και με τη σύσταση του δικαστηρίου ήταν αδύνατο κάτι τέτοιο. Αν έχουμε λοιπόν έναν ειδικό επόπτη για την ιδιωτική σφαίρα ή έναν ειδικό συνήγορο για την ιδιωτική σφαίρα θα καλύπταμε αυτό το κενό. Το πιο σημαντικό πάντως μεταρρυθμίσεις που προτείνουμε και για τη μεταρρύθμιση του δικαστηρίου της ΦΑΙΣΑ είναι ότι όταν αλλάζουμε πολιτικές δεν πρέπει, δεν πρέπει να, κατά, να, να δημοσιεύονται. Αλλά όταν μιλούμε για ένταλμα του δικαστηρίου ΦΑΙΣΑ για να ελεγχθούν τα επιχειρηματικά μητρώα κάποιων που, για τον οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι συμμετείχε σε μια τρομοκρατική απόπειρα, είναι λογικό να είναι εμπιστευτικές αυτές οι πληροφορίες. Γιατί σίγουρα αν γνωρίζει ο τρομοκράτης ότι έχει αποκαλυφθεί θα βρει άλλους τρόπους για να υλοποιήσει τους στόχους. Οπότε αν καταργηθεί το δικαστήριο αυτό για τον έλεγχο των ξένων μυστικών υπηρεσιών θα πρέπει να έχουμε κάτι αντίστοιχο. Ίσως το συνήγορο ε, του πολίτη για την ιδιωτική σφαίρα, Privacy Advocate. Έτσι θα είχαμε καλύτερη διαφάνεια και ίσως και μία αλλαγή στο δικαστήριο. Γιατί η επανερμηνία του Patriot Act έγινε από την NSA και το δικαστήριο κυρίως αυτή την πλευρά άκουγε. Έχουμε τώρα τον κύριο Πίρκερ, την κυρία Ζίβελ, Τόρβαλτς και τον κύριο Ρομέβα. Δεν ξέρω αν άλλο κάνει θέλει το λόγο για να ολοκληρώσω το κατάλογο. Ο κύριος Πίρκερ. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ζένζεν Μπρένερ, όχι μόνο που ήρθε στο κοινοβούλιο. Α, θα τα πω στη μητρική μου γλώσσα αν δεν σα πειράζει. Ε, σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Σένσενμπρένερ, όχι μόνο που ήρθατε, αλλά για την τόσο ειλικρινή και επικοδομητική συνομιλία που είχαμε στην Όσουγκτον πριν από λίγες μέρες. Ειλικρινής και ανοιχτή λέγω, γιατί είπατε ότι η συνεργασία προ όφελο αμοιβαία ασφάλεια είναι σημαντική γιατί τελικά και οι δύο υποφελούμεθα. Αλλά όλα αυτά βασίζονται στην εμπιστοσύνη και τελικά σε μια νομική βάση και νομοθετική οφείλει να βασίζεται. Ε, συχνά είπατε ότι χάθηκε η εμπιστοσύνη ακριβώ και σα παραθέτω τώρα, είπατε ότι η NSA είναι τελείω ασίδωτη, εκτός κάθε ελέγχου. Totally out of control και κάθε μέρα ε, αγνοεί τον νόμο. Ε, δηλαδή, ε, και εσείς ο ίδιος αναφερθήκατε με μεγάλη ειλικρίνεια σε αυτό που θέσαμε υπόψη και σας ευχαριστώ. Τώρα όμως, τι μελιγενέστε, τι συμπεράσματα θα βγάλετε από αυτά. Και η συγκεκριμένη ερώτηση, ποια είναι η νομοθετική βάση που κατά την άποψή σας αμελείται και αγνοείται από την NSA και για ποιο λόγο. Πώς εφτάσαμε εδώ να αγνοεί ε, και να αψηφεί αυτούς τους νόμους. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το μέλλον. Πώς θέλετε να επιτύχετε στι Ηνωμένες Πολιτείες, η NSA και άλλες μυστικές υπηρεσίες πραγματικά να ελέγχονται και ουσιαστικά να δρούν βάση του νόμου και υποέλεγχο και εποπτεία. Πάντα βεβαίως κατά της τρομοκρατίας και ε, εποφελία ε, της ασφάλειας και της εταιρικής σχέσης με την Ευρώπη. Και δεύτερη ερώτηση για το μέλλον. Αυτή η νέα νομοθετική ρύθμιση θα αφορά μόνο τους πολίτες ε, τους Αμερικανούς ε, ή και τους Ευρωπαίους που βλέπουν τα δεδομένα τους να κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά στις Ηνωμένε Πολιτείες και να τα επεξεργάζονται διάφοροι. Και μια τελευταία ερώτηση. Σε συνέχεια με το SWIFT και την ανταλλαγή δεδομένων αφορά τη Συμφωνία Πλαίσιων ε, Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για την ποινική δίωξη, δηλαδή ανταλλαγή πληροφοριών βάσει συμφωνίας για τις ποινικέ διώξεις. Αυτό πότε βλέπετε να γίνεται πραγματικότητα. Θα τα απαντήσω αντίστροφα για την προστασία των δεδομένων στην περίπτωση ποινική δική. Είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα στη συνάντησή μα με την Επίτροπο Ρέντινγκ και τον, και τον ε, Υπουργό Χόλντινγκ. Ελπίζουμε, δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει τελικώ μια συμφωνία, αλλά σίγουρα θα επιτευχθεί κάποια πρόοδο, ελπίζουμε. Έπειτα, σχέτω με το τι προβλέπει ο νόμο. Εάν ένα φορέα ή οργανισμό ξέρει ότι μπορεί να αγνοήσει την εποπτεία ή ότι δεν υπάρχει στην ουσία εποπτεία, ο οργανισμό θα φτάσει ως τα όρια των εξουσιών και θα τα υπερβεί. <clears throat> Αυτό έκανε η NSA και όσοι νομίζουμε ότι η NSA υπερεύει τα όρια που της είχαν αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Ε, ο, το Freedom Act πέρασε για να υπάρξει ακριβώς δυνατότητα ε, να υπάρξει καταγγελία εφόσον χρειαστεί. Γι' αυτό είναι σημαντική η εποπτεία της NSA από το Κογκρέσο, από το Λευκό Οίκο, από το το Δικαστήριο και ως προς τη βελτίωση της Αμερικανικής νομοθεσίας. Ιδιαίτερος ως προς την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών που επισκέπτονται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τελικά θα καταλήξουμε στην νομοθεσία που οι λέει τον και εγώ έχουμε προτείνει. Την έχει προτείνει και ο, ο κ. Φάινστάιν και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή για τις Μεστικές Υπηρεσίες με ε, ψηφοφορία 11 προς 4. Αυτό ουσιαστικά βέβαια επιτρέπει αυτό που έκανε η Νησέιος τώρα ε, για τη μαζική συλλογή δεδομένων και είναι τρομακτικό γιατί το ανώτατο δικαστήριο φαίνεται να επιτρέπει να γίνει το δικαστήριο της Φάιζα. πρέπει να υπάρξει όμως δικαστική εντολή και εάν ο νόμος αυτός περάσει θα, καταστεί το έργο της NSA νόμιμο. Επίσης για τους Ευρωπαίους που σκέφτονται τις ΗΠΑ επιτρέπεται 72 ώρες κράτηση ή έρευνα χωρίς να υπάρχει καν ε, η εντολή του Γενικού Σαγγελέα για να γίνει κάτι τέτοιο. Πολιτικός λοιπόν έλεγχος και επιβολή του νόμου από την πλευρά του Γενικού Σαγγελέα και του Υπουργού Δικαιοσύνη ή την επίβλεψη τελικά του Αμερικανού Προέδρου είναι κάτι που χρειάζεται. Δεν μπορεί να υπάρχει κράτηση 72 ωρών χωρί να γνωρίζει καν ο Γενικό Αγγελέα ότι συμβαίνει. Είναι τρομακτικό κατά την άποψή μου. Ευχαριστώ κυρία Σίπολ. Κυρία Ζίπελ, ευχαριστώ πολύ. Ε, θα τα πω και εγώ γερμανικά. Όταν επιτίθεται κάποιος σε μια χώρα, υφίσταται επίθεση μια χώρα, κάθε κυβέρνηση κάθεται και ε, προβληματίζεται για το πώς θα αντικρούσει αυτή την επίθεση. Και κατανοώ τα μέτρα ε, που υιοθετήθηκαν μετά την επίθεση της 11 η Σεπτεμβρίου. Από την άλλη όμως, στο μεταξύ έχουν πέρασει 12 χρόνια. Και, και εγώ δεν πρόκειται ποτέ να ισχυριστώ ότι δεν υπάρχει τρομοκρατία. Αλλάζουν τα πράγματα. Ποτέ μέσα σε αυτά τα 12 χρόνια δεν υπήρξε μια χρονική στιγμή όπου η κυβέρνηση των μέρων πολιτιών, το Κογκρέσο, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, να κάτσει να προβληματιστεί αν όλα αυτά τα μέτρα που είχαν αποφασιστεί τότε ε, είναι εύστοχα, είναι σκόπιμα, χρειάζονται ακόμα, ε, είναι ε, χρήσιμα ή όχι. Αναφερθήκατε στη γνωστή ρίση «καλός ο έλεγχος, καλύτερη, η εμπιστοσύνη, συγγνώμη, καλύτερος ο έλεγχος. Ε, όταν ε, μια υπηρεσία παίρνει περισσότερους οικονομικούς πόρους και εξουσίες, κινδυνεύει να αυτονομείται. Γιατί λοιπόν την τελευταία δωδεκαετία ουδέποτε κανείς δεν σκέφτηκε να κοιτάξει λίγο περισσότερο τι κάνει η NSA και άλλες ε, μυστικές υπηρεσίες για να δούμε κατά πόσο ευσταθούν αυτά τα μέτρα, έχουν περιοριστεί οι ελευθερίες ε, των πολιτών. Μήπως όλα αυτά είναι ατελέσφορα, έχουν νόημα γιατί είναι πολύ υψηλό και το κόστος και το προσωπικό πολύ πληθές που απασχολείται εκεί. Είπατε τώρα ότι θέλετε να επαναφέρετε την ισορροπία σε μερικά πράγματα, την ασφάλεια και τα δικαιώματα των πολιτών. Από την άλλη όμως ε, ανακύπτει για μένα το εξής ερώτημα όπως και στην Ευρώπη. Αν δεν είχε αποκαλύψει όλα αυτά ο κύριος Σνόουντεν, μάλλον όλα θα συνέχιζαν την λειτουργία τους όπως τώρα. Και ρωτώ, γιατί δεν ελέγχθηκαν μέχρι τώρα οι, νομε... οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Και επιπλέον, αν είναι σοβαρό αυτό που λέτε ότι μάλιστα οι μυστικές υπηρεσίες αυτονομήθηκαν και έκαναν πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν και δεν είναι εντάξει, μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε και όλα στη μεταχείριση θα πρέπει να επιφυλάξει οι ΗΠΑ προς τον κύριο Σνόουντεν σε σχέση με αυτή που του επιφυλάτουν αυτή τη στιγμή. Η ερώτηση, η απάντηση στην με τη της είναι όταν συνέταξα το Πάτριο Τάκτα ε, μίλησε για σταδιακή εξάλληψη σε τέσσερα χρόνια και δόθηκαν εκτεταμένες εξουσίες και στις αστυνομικές αρχές και στις μυστικές υπηρεσίες και προσθέθηκε μια διάταξη στη νέα ε, διάταξη για την, απομονωμένες περιπτώσεις τρομοκρατίας. Όταν όμως ε, ολοκληρώθηκε η τετραετία αυτή για τη σταδιακή εξάλληψη, εγώ ε, τήρησα την υπόσχεση που είχα δώσει στη χώρα και στους ψηφοφόρους μου ότι θα κάνω συγκεκριμένες ακροάσεις για τις επιπλέον αυτές εξουσίες, για να καταλήξω το συμπέρασμα αν θα έπρεπε να παραταθεί ο νόμος ή όχι και 14 από τις 17 εξουσίες ε, δεν ήταν επίμαχες και θα μείνουν ισόβιες. Το πιο σημαντικό ήταν η διάταξη που εμπόδιζε το FBI και τη CIA να ανταλλάξουν πληροφορίες μυστικές που ε, είχε συγκεντρώσει η Επιτροπή για, την, για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Ενάτου, γιατί έτσι έφτασαν και που έφτασαν οι τρομοκράτες. Επίσης είχαμε το τμήμα 215 που είναι και το πιο επίμαχο και αφιλεχόμενο και μάλιστα αυτό προσωρινά είχε παραταθεί και στις, την 1η Ιουνίου του 2015 θα εξαλειφθεί, θα καταργηθεί. Και είπα στο με του νόμου ότι αν ε, δεν ε, εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις που προτείνουμε τον κύριο Λίχ οι, νομικές, οι μυστικές υπηρεσίες ε, θα διδρέξει τον κίνδυνο να χάσουν τελείως το τμήμα 215 γιατί ακριβώς εξαιτία των προβληματικών διατάξεων είχαμε αυτές τις παρεκτροπές. Θα πρέπει λοιπόν οι παρακολουθήσεις να γίνονται στοχοθετημένα μόνο για όσους υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι αναμειγνύονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητε. Αυτό που συνέβη αν δείτε πώς η NSA, από εκεί που στοχοθετημένα παρακολουθούσε κάποιους που, για τους οποίους υπήρχαν βάσει υπόνοιες για τρομοκρατική ενέργεια, έχει φτάσει στα σημερινά έκτροπα, είναι ότι το 2006 έλαβε την άδεια που μιλούσε για relevant, δηλαδή ε, σχετικά με μια ε, τρομοκρατική επίθεση. Οπότε με τη χρήση του όρου relevant πολλοί θεωρούσαν ότι θα περιοριζόταν το πεδίο μιας έρευνας. Ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας έπεισαν το δικαστήριο Φάισα να διευρύνει, να υιοθετήσει διασταλτική ερμηνεία αυτού του όρου. Οπότε ε, έχουμε και μητρό τηλεφωνικών κλήσεων που ουσιαστικά επιτρέπει αναζήτηση δεδομένων, data mining, για υπόπτους τρομοκρατίας και οι εξωματούχοι της NSA σε δημόσιες ακροάσεις είπαν ότι μόνο σε μία περίπτωση από όλα αυτά τα στοιχεία κατάφεραν να, να ισχυριστούν ε, ότι με τη συγκέντρωση των στοιχείων κατάφεραν να χαιτήσουν μία τρομοκρατική ενέργεια. Ενώ είχαμε μία τεράστια επέμβαση στην ιδιωτική σφαίρα. Και η ερώτηση που δεν απαντήθηκε ποτέ ήταν ε, σε ό,τι αφορά την επανερμηνία του όρου relevant, θα μπορούσαν να σταματήσουν τις, ή να αναποσοβήσουν ε, τρομοκρατικές ενέργειες με άλλα μέσα. Εξαρτάται από το είδος της εποπτείας που εφαρμόζεται. Το δικαστήριο Φάισα και η Επιτροπή Μυστικών, η Επιτροπή Μυστικών Υπηρεσιών της Γερουσίας ε, είχαν ιδρυθεί το 1970, τη δεκαετία του 70 μετά από ε, καταχρήσεις που έγινε και τότε από τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Και τότε οι νεοσταθήσει υπηρεσίε ε, πρόκειτο να περιορίσουν ε, τα έκτροπα και τι καταχρήσει των μυστικών υπηρεσιών. Τελικά, αντί να αναχαιτήσουν τις υπηρεσίες, ουσιαστικά τις, τους έδωσαν ακόμη μια μεγαλύτερη όθηση σε, αυτές τις, σε αυτήν την ασίδωτη δραστηριότητα. Έτσι δημιουργήθηκε μια αντιπαράθεση μεταξύ της Επιτροπής Δικαστικών Υποθέσεων της Γερουσίας και της Επιτροπής της Αρμόδιας για τις Μυστικές Υπηρεσίες της Γερουσίας. Ο Γερουσιαστής Λέχη, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, ε, για τις δικαστικές υποθέσεις της Γερουσίας. Εγώ ήμουν το, ο αντίστοιχος πρόεδρος ε, του Κογκρέσου. Γνωρίζουμε ότι γίνονται κάποια, κάποια κατάχρηση της νομοθεσίας και έκτροπα και θέλουμε να σταματήσει αυτή η κατάσταση και φυσικά να αποφευθεί η επαράληψή της στο μέλλον. Ευχαριστώ. Επειδή και άλλοι συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο, έχω ακόμη τέσσερις ομιλητές θα ζητήσω από όλου να προσπαθήσουν να αυτοπιθαρχηθούν και να είστε σύντομοι. Κύριο Στόρβαλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Σάνσερμπρένερ. Ξέρουμε ποια ήταν η αμερικανική πολιτική του 90, της δεκαετίας του 90 Ξέρουμε ε, τι προσπάθειες κάνετε για να πετύχετε όσα λέτε. Αλλά είναι μεγάλη πρόκληση. Αν δείτε τον όγκο των δεδομένων που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή και τα συγκρίνετε με το τι συνέβαινε με την 11η Σεπτεμβρίου λόγου χάρη, έχει υπάρξει τεράστια αύξηση. Υπάρχει και πολύ κακός προγραμματισμός επίσης. Δεν είναι απλό να προστατεύσουν τα δεδομένα των πολιτών. Αμερικανών ή Ευρωπαίων. Όλα τα προγράμματα έχουν ε, πάντοτε κάποια παραθυράκια, κάποιες κερκόπορτες, είτε ηθελημένα είτε όχι. Και προφανώς θα είναι πολύ σκληρότερος ο αγώνας σας από τη δεκαετία του για να πετύχετε αυτά που λέτε. Αλλά πραγματικά θα ήθελα την άποψή σας. Πώς αυτός ο τεράστιος, αυτός ο απέρατος όγκος, πόσο μεγάλο πρόβλημα δημιουργεί. Κοιτάξτε για τον ε, κύριο και εμένα. Θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη για να περάσει η δική μας γραμμή και να πείσουμε τους, ε, τους, πούς ε, επικεφαλείς διότι πρέπει να πιστούν τα μέλη της Επιτροπής για τις Μυστικές Υπηρεσίες. Ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ήταν το γεγονός ότι η τροπολογία για, το, ε, για τη συλλογή δεδομένων από τα τέλη Ιουλίου δεν πέρασε μόνο για 7 ψήφους. Αυτό έδωσε ένα μήνυμα προς, τους, ε, προς την απέναντι πλευρά ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Αυτό το νομοσχέδιο όπως προτάθηκε εξετάστηκε μέσα σε 24 ε, μην, ε, ώρες, πριν από 3,5 μόλις μήνες και έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση. Το θέμα είναι ότι αφού με τόσο μικρή διαφορά δεν πέρασε αυτός ο νόμος, ο γενικός ε, διοικητής της NSA είπε ότι υπήρξε αυτοπαραβίαση του καταστατικού τους. Προφανώς όσοι εργάζονται για την NSA καταλαβαίνουν ότι ακόμη και το καταστατικό του δικού του οργανισμού μπορεί να, να παραβιαστεί. Όσο περισσότερο λοιπόν συζητιέται το θέμα, τόσο περισσότερο ευαισθητοποιείται το κόσμο και θα υπάρξει και μεγαλύτερη στήριξη. Το πραγματικό θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να περάσει βέβαια όμω ε, οι προτάσει μα. Και στη Βουλή και στη Γερουσία. Χαίρομαι που ο γερουσιαστή Λί, ένα από τα μέλη τη ε, Γερουσία, έχει περάσει αυτή τη γραμμή και το μήνυμα και προς την Προεδρία. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ρωμέβα. Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλος λόγος γίνεται για τις επιπτώσεις αυτής της κατάχρησης και παρέμβασης των νόμων από την NSA σε επίπεδο κυβερνητικό, διακυβερνητικό κτλ. Ε, η δική μου ερώτηση είναι σχετική. Ποια είναι η δική σας αίσθηση χρησιμοποιήθηκε αυτό για να ελεγχθούν οι αγανακτισμένοι, ε, το κίνημα κατάληψης της Wall Street, ε, Occupy Wall Street, κάποια μαζικά κινήματα καθόλου θεμητά και νόμιμα. Ε, μήπως ε, υπέστησαν αυτή την επίθεση ακριβώς εν ονόματι της τρομοκρατίας για να ελεγχθούν λοιπόν κάποια πολιτικά, ποια πολιτικά, κάποια κοινωνικά κινήματα χρησιμοποιούνται ε, τέτοιες ε, καταστάσεις από κυβερνήσεις. Έχετε την αίσθηση ότι χρησιμοποιήθηκε αυτό το στοιχείο για να ελεγχθούν αυτά τα κινήματα έτσι Ηνωμένε Πολιτείε και στην Ισπανία και στην Ευρώπη και στο μέλλον, ποια κατεύθυνση παίρνουν. Μπορώ να σας πω απαντώντα αυτό ότι σε ό,τι αφορά την εσωτερική πολιτική στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχω την ε, εντύπωση ότι είναι κάτι που αφορά κανέναν άλλον παρά μόνο τα κράτη-μέλη και την Ευρώπη. Υπάρχουν και οι συνθήκες ε, που διέπουν τη λειτουργία της Ένωσης και των Βρυξελών. Πάντως, οι αποτελεσματικές έρευνες κατά της τρομοκρατίας ε, εμπεριέχουν και το στοιχείο της ανταλλαγής ε, μυστικών πληροφοριών από τις υπηρεσίες. Και η νομοθεσία Freedom Act μπορεί να επαφέρει την ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ε, ελευθερία και τις πολιτικές ελευθερίες. Ε, στο Patriot Act, πριν την απόφαση του δικαστηρίου Φάιζα, ε, γιατί ο όρος relevant κατάλληλα ήταν υπερβολικός και μάλλον δεν περιόριζε τις εξουσίες αλλά τις διεύρυνε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να προσθέσω τι ευχαριστίε μου και εγώ στον κύριο Σενεσέ Μπέργκε που ήρθε να μα μιλήσει. Το εκτιμούμε ιδιαιτέρω. Αυτό που σκέφτηκα είναι ότι έχω την απορία. Είχατε την ευκαιρία ή θα υπάρξει ίσως ευκαιρία να συνομιλήσετε με πολιτικούς στο Λονδίνο από όλε τις πολιτικές πρατάξεις γιατί νομίζω ότι είστε το κατάλληλο άτομο για να μιλήσετε ιδίω στους συντηρητικού και του εκπροσωπούς του. Γιατί όπως τα γνωρίζετε, δεν έχει γίνει σοβαρή συζήτηση, είτε δημόσια, είτε ε, μεταξύ πολιτών, όπως ε, αυτά που αφορούν για τα θέματα που προκύπτουν από την Ουάσιγκτον. Ο Πρωθυπουργό μας σκέφτηκε και μίλησε ακόμη και για κατηγορίες κατά του, της Guardian που δημοσίευσε στοιχεία του Snowden Κάτι που θα ήταν ε, αδύνατο ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς. Ποια θα θέλατε λοιπόν να απαντήσετε σε αυτό το, αυτό το θέμα που σας θέτω ε, ως δέλεαρ για να δούμε ποιες είναι οι απόψεις, να αποπειραθείτε να δώσετε κάποιες απόψεις διότι πραγματικά δεν υπήρξε σοβαρή συζήτηση στο Λονδίνο και δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη συμφωνία για το θέμα αυτό μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, ούτε εξισορρόπηση των αναγκών, ε, ανταλλαγής δεδομένων τελικά. Κοιτάξτε, ε, δεν θα ε, τσιμπήσω ακριβώ το δόλωμά σα. Ε, για την εθνική κυβέρνηση ενό κράτου μέλου. Δεν ξέρω αν μπορώ να ασκήσω κριτική για το πώ χειρίζεται τι μυστικέ τη υπηρεσίε και την ανταλλαγή δεδομένων. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να παραμείνει υπόθεση εσωτερική. Και είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους βρίσκομαι εδώ σήμερα και έχω δεχτεί την πρόσκλησή σας. Γιατί υπάρχουν δείγματα ότι η μαζική συλλογή δεδομένων είχε αντίκτυπο και στην Ευρώπη. Ιδιαίτερο σε ορισμένε χώρες. Είναι πάντοτε χαρά μου να μιλώ για τα λεπτά όρια μεταξύ ασφάλειας και ελευθεριών των πολιτών μεν. Από την άλλη όμως αυτό που είχα προτείνει και ζήτησα και τώρα προτείνω ξανά είναι να υπάρξει ένας ε, νόμος γενικός για την προστασία δεδομένων που να αφορά όλο τον πολιτισμένο κόσμο διότι δεν θα δουλέψει ε, αλλιώς ε, λόγω των ε, μεγάλων διαφορών των συνταγματικών και νομοθετικών λεπτομεριών που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Τελευταίο ομιλητή ο κύριο Άγκστρομ. Ευχαριστώ. Αναφέρατε ότι η NSA είπε κάποια στιγμή ότι η εποπτεία επέτρεψε μόνο την αποφυγή μιας μόνο τρομοκρατικής ε, απειλής. Σε αυτή τη μία περίπτωση υπήρξε καμιά καταδίκη, διότι Ξέρουμε όλοι ότι είναι σοβαρά το, αδίκημα η προετοιμασία τρομοκρατικού χτυπήματος, έτσι. Ε, υπήρξε καμιά καταδίκη. Τι έγιναν αυτοί οι ύποπτοι που εντοπίστηκαν χάρη στη δράση της NSA. Κοιτάξτε, η απάντηση είναι ότι καταδίκη υπήρξε, αλλά ως προς την χρηματοδότηση. Χρηματοδότηση όσων ε, σχεδιάζονταν και όχι ως προς ίδια την επίθεση. Εάν μου επιτρέπετε να πάω ένα βήμα παραπέρα, η διαφορά μεταξύ τρομοκρατία και οποιοδήποτε, και οποιοδήποτε εγκληματική ενέργεια σημαίνει ότι αν ένα έγκλημα, οι διοκτικέ αρχέ μπαίνουν σε διαδικασία αντίδραση. Δηλαδή να εντοπίσουν το δολοφόνο, να συγκεντρώσουν τα αποδεκτικά στοιχεία, να μιλήσουν με του μάρτυρε, να προσπαθήσουν να αποδείξουν τι συμβαίνει με την υπόθεση, να συγκεντρώσουν στοιχεία και να την περάσουν στον εισαγγελέα ή τον ανακριτή για να πάει στο δικαστήριο. Αλλά στην περίπτωση τη τρομοκρατία πρέπει κανείς να είναι πιο πολύ ενεργός παρά να αντιδρά. Διότι είναι πολλά αυτά που διακυβεύονται. Ε, είναι περίπου 3.000 ναι, οι ζωές που χάθηκαν την 11η Σεπτεμβρίου. Ε, αυτοί που ε, βρίσκονταν στα αεροπλάνα είναι αυτοί που έχασαν τη ζωή τους στη Δυτική Πενσιλβάνια και όσοι ήταν στα κτίρια. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει με μια αθλητική διοργάνωση. Δεκάδε χιλιάδε άνθρωποι που μπορεί να απειλούνται οι ζωέ του. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσουμε την ε, δράση πρωτού γίνει η επίθεση. Γι' αυτό ε, ο βασικό υπεύθυνο για την νομοθεσία αυτή, στην οποία έχω συμμετάσχει και εγώ ω προ το σχεδιασμό τη, πρέπει να έχουμε πόσο θα χρειαστεί και τη συγκέντρωση πληροφοριών και την ε, παρακολούθηση και την εποπτεία. Αλλά πρέπει να γίνεται αυτό μέσα σε ένα πλαίσιο συνταγματικό πρέπει να γίνεται βάσει κάποιου νόμου, οποιοδήποτε αν είναι αυτός ο νόμος και όπου ισχύει, εκεί όπου η δράση μπορεί να πραγματοποιηθεί. Η τρομοκρατική επίθεση στη Γερμανία, μάλλον η τρομοκρατική οι τρομοκράτε στη Γερμανία σχεδίαζαν χτύπημα στι Ηνωμένε Πολιτείε. Εντοπίστηκαν στη Γερμανία. Αυτό θα έπρεπε να κριθεί με βάση αυστηρά το γερμανικό δίκαιο. Είναι και θέμα εδαφικότητας ε, του αμερικανικού δικαίου. Όμως τώρα αυτοί οι συνομότες είτε είναι Γερμανοί πολίτες είτε πολίτες μιας άλλης χώρας και εφόσον εκδοθούν στις ΗΠΑ θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα αποδεκτικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί βάσει του γερμανικού δικαίου και να τους εκδικάσουμε. Ή ακόμη και αν δεν, έχουν, ε, δεν έχει διακοπεί δράση τους να ε, προσπαθήσουμε να, να, να ανακόψουμε την πορεία τους. Σας ευχαριστώ. Η τελευταία σας παρατήρηση ε, δημιουργεί ένα ερώτημα, γιατί η εξοδαφικότητα η εξοδικία δημιουργεί πρόβλημα γιατί δεν, ε, αποτελεί, δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία ενός ε, τρομοκράτη στο, στην Αμερικανική επικράτεια. Απλώς χρειάζεται πρόσβαση των δεδομένων του είτε στην Αμερικανική επικράτεια ή οπουδήποτε αλλού. Υπάρχει ένα ουσιαστική δηλαδή εξοδαφικότητα όπου και αν ε, σχεδιάζει κανείς τρομοκρατική ενέργεια οπουδήποτε στον κόσμο, ακόμη και στην Γερμανία. Μας έχει απομείνει ε, ελάχιστος χρόνος, αν θέλετε να υποβάλλετε κάποια συμπληρωματική ερώτηση. Μία τελευταία ερώτηση, συναφής, είναι συναφής προς την προηγούμενη, σε ό,τι αφορά το νόμο για την παρακολούθηση αλλοδαπών μυστικών υπηρεσιών, ΦΑΙΣΑ και εφαρμογή του νόμου αυτού σε προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών. Εκεί δεν υπάρχει καμία δυνατότητα προσφυγής ενδίκων μέσων ούτε καν των Αμερικανών πολιτών προς το Ανώτερο Δικαστήριο. Έχετε κάποιο σχέδιο για τη μεταρρύθμιση και αυτού του δικαστηρίου. Σε ό,τι αφορά το νόμο Φάισα, ε, ένας Αμερικανός πολίτης δεν ξέρει αν το δικαστήριο έχει ε, εκδώσει εντολή επιτρέποντας ε, αστυνομικές υπηρεσίες ή υπηρεσία μυστικών υπηρεσιών έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα. Τώρα, αν έχει ε, κατηγορηθεί αυτός η αποκάλυψη ποινικη διαδικασια ποινικη οποτε η αποκαλυψη αυτων των πληροφοριών στους συνηγόρους του για να προετοιμαστεί η υπεράσπιση, αν δεν είχε συγκεντρωθεί νόμιμα αυτές ε, οι πληροφορίες, αυτό είναι ένα επιχείρημα που μπορεί να επηρεάσει το δικαστήριο. Υπάρχει όμως διαφορά μεταξύ των υπηκών κατοίκων των Ηνωμένων Πολιτειών και των υπολείπων. Ε, υπάρχει διαφορετικά στη μεταχείριση και αν ναι, πώς αντιμετωπίζετε αυτή τη διακριτική μεταχείριση μεταξύ Αμερικανών και λοιπόν πολιτών. Επανερχόμαστε και πάλι στην συνάντηση που θα έχουν την επόμενη εβδομάδα η Επίτροπος Ρέντι με τον Αμερικανό Υπουργό Δικαιοσύνης. Εκεί θα δούμε τι νομικές συμφωνίες θα γίνουν ή τι διευθετήσεις. Το καλύτερο παράδειγμα θα είναι ένας ε, Αμερικανός πολίτης να μπει σε ένα κατάλογο για απαγόρευση πτήσης στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, παρόλο που δεν έχει καμία σχέση με την νομοκρατία. Συνέβη αυτό σε Αμερικανός πολίτες, ακόμη και στον γερουσιαστή Κέννεντι. Γιατί κάποιος με παρόμοιο όνομα είχε ε, συσχετιστεί με τον Ήρα στην Βόρεια Ιρλανδία και ε, κανονικά δεν, δεν να επανέλθει στην, στον κατάλογο για να το επιτραπεί η πτήση. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπρένερ για την παρουσία σας εδώ, Σέσεν Μπρένερ, ε, και για την παρουσία σας και για την προθυμία σας να απαντήσετε σε τόσες ερωτήσεις και ελπίζω να μπορούμε να υπολογίζουμε σε εσά και στην προσήλωσή σας και τη δέσμευσή σας για τη συνέχιση του διαλόγου, γιατί πραγματικά πολλά σημεία θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον. Και παρακαλώ λίγη ησυχία ακόμη. Είπατε κύριε Βουλευτά, κύριε Γερουσιαστά, ότι θα ήταν δυνατό ακόμη και ένα παγκόσμιο νομοθετικό σύστημα για την ιδιωτική σφαίρα. Γιατί έχουμε διαφορετικές ένομες τάξεις, αλλά πρεσβεύουμε τις ίδιες αρχές. Ε, βέβαια, εμείς θέλουμε ε, αναλογικότητα και αναγκαιότητα που θα πρέπει να συνδυαστούν. Και φυσικά η προάσπιση των πολιτικών ελευθεριών είναι ένα κοινό μας μέλημα και σίγουρα αποτελεί προϋπόθεση για τις επιτυχείς συμφωνίες και την αίσια έκβαση και των εμπορικών μας συμφωνιών. Θα πρότεινα λοιπόν μια νέα συνάντηση κάπου την Άνοιξη για να συνεχίσουμε την αγαστή μας συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Um, Ωραία. Περνάμε στο δεύτερο πάνελ τώρα. Ο ρόλος ε, της κοινοβουλευτικής εποπτείας στις μυστικές υπηρεσίες, ε, εθνικές μυστικές υπηρεσίες σε μια εποχή μαζικής παρακολούθησης. Θα έχουμε δύο μιλητές. Πρώτα τον κύριο Πίτερ Έριξον που είναι πρόεδρος της Επιτροπής για το Σύνταγμα στην Σουηδική Βουλή, το Ρίξτακ. Και ο δεύτερος ομιλητής μας είναι ο κύριος Βαντέλδεν, πρόεδρος της ε, ε, Ολλανδικής Ανεξάρτητης Επιτροπής Επανεξέτασης των, υπηρεσιών, των Μυστικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Ασφάλειας. Okay, colleagues, we continue with the second... Συνάδελφοι, να, ξεκινήσουμε με το δεύτερο, να συνεχίσουμε με το δεύτερο πάνελ. Όσοι συζητούν σε πηγαδάκια, αν θέλουν να πάνε τα πηγαδάκια έξω. Κύριε Άλμπερτ. Ωραία. Καλωσορίζουμε τον κύριο Έριξον και τον κύριο Φαντέλντεν. Θα προσκαλέσω και τους δύο κυρίους να μας κάνουν μια σύντομη παρουσίαση. Δεκάλεπτη ο καθένας και μετά θα έχουμε Συζήτηση. Διαδικαστικό, κύριε Πυρκά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους της Σουηδικής Αντιπροσωπείας έχω μια ερώτηση, διότι δεν υπάρχει αρκετή σαφήνεια να το κάνουμε. Μου, τέθηκε να... μου ζητήθηκε να θέσω το ερώτημα αυτή εξ αρχή, πριν αρχίσει η συζήτηση του πάνελ. Στη Σουηδία, η Επιτροπή για τις διαγματικές υποθέσεις δεν είναι αρμόδια στο Σουηδικό Κοινοβούλιο για το θέμα που σήμερα συζητούμε, δηλαδή για την προστασία των δεδομένων και τη δράση των μυστικών υπηρεσιών. Το ερώτημα λοιπόν τη Σουηδική Αντιπροσωπείας είναι γιατί προσκλήθηκε ο κύριος Έριξον. Ο κύριος Έριξον είναι εδώ ο μιλητή που εκπροσωπεί την Επιτροπή του Σουηδικού Κοινοβουλίου, τις οποία προεδρεύει, διότι δεν είναι η αρμόδια επιτροπή στο συγκεκριμένο τομέα. Υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση για την οποία έχει προσκληθεί συγκεκριμένα ο κύριος Έριξον, πρόεδρος. Νομίζω η απάντηση ε, αναφέρεται στα email που λάβατε κι εσείς, το λάβαμε όλοι πριν από την έναρξη αυτής της συναντρίασης, αν καλά κατάλαβα, είναι δύο συναρμόδιες επιτροπές στο Σχετικό Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά, αυτή είναι η μία από τις δύο, και νομίζω ότι το αίτημα για να αποσταλεί ο μιλητής έγινε από τους επισημότερους κοινοβουλευτικούς διάβλους, ο κύριος Έριξον προτάθηκε λοιπόν από το Σχετικό Κοινοβούλιο το ίδιο. Δεν βλέπω να υπάρχει εδώ κάποιο ζήτημα. Εάν λοιπόν ξεκαθαρίστηκε το θέμα, να δώσω το λόγο στον κύριο Έριξον. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Θα ξεκινήσω απαντώντας κι εγώ στην ε, ερώτησή σας. Ε, την πρόσκληση αφετή την έλαβα από την κυρία Κοράτσα Μπίλτ και την κυρία Όλσον. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ είναι σύζυγος του Σουηδού Υπουργού Εξωτερικών. Και είναι τρεις οι επιτροπές μας στο στην Σουηδική Βουλή, που είναι ταυτόχρονα αρμόδιες για τα θέματα αυτά από τρεις διαφορετικές σκοπιές. Αλλά η Επιτροπή που περισσότερο ασχολείται με τα θέματα αυτά είναι η Επιτροπή Άμυνας. Διότι προφανώς αφορά πολλά ζητήματα της αμυντικής πολιτικής και υπάρχει αυτή τη στιγμή και μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα. Αλλά και η Επιτροπή Δικαιοσύνης. Η, Επιτροπή για τις Συνταγματικές Υποθέσεις έχει αρμοδιότητες για τις ελευθερίες των πολιτών. Λόγω χάρη για τα θέματα ακεραιότητας, όπως τα ονομάζουμε. Γι' αυτό και η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων είναι είναι συν-αρμόδια, εν μέρη αρμόδια για τα θέματα αυτά. Έχετε λοιπόν ε, εν μέρη δίκιο, αλλά ίσως όχι απολύτως δίκιο. Ελπίζω να ε, μου επιτρέψετε να περάσω στα σουηδικά στη μετρική μου γλώσσα κατά την ομιλία μου. Μετά ίσως να έχουμε το διάλογο στα αγγλικά όταν περάσουμε σε ερωταπαντήσεις αλλά είναι κάπως τεχνικό το ζήτημα και θα προτιμούσα να μιλήσω σουηδικά για να μην κάνω και σοβαρά λάθη. Η κατάσταση στη Σουηδία για θέματα που αφορούν τις μυστικές υπηρεσίες και την υποπτία τους ή την υποπτία του διαδικτύου ε, έχουν οργανωθεί ως εξής. Το 2008 για το 2009 είχαμε μια πολύ εντατική συζήτηση για τα θέματα αυτά, διότι η Σουηδική κυβέρνηση υπέβαλε ένα νομοσχέδιο για να ρυθμίσει τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι μυστικές υπηρεσίες. Κάτι που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν διέπεται από νομοθεσία. Έτσι ξεκίνησε μια σοβαρή συζήτηση με πολλές επικρίσεις κατά το νομοσχεδίο από μεγάλο αριθμό οργανώσεων και οργανισμών και εκτός κοινοβουλίου και ε, εντός. Ε, τα επικριτικά σχόλια αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό το κατά πόσον είναι δέον να παρακολουθούνται οι συνομιλίες πολιτών στη Σουηδία. Ε, συνομιλίες ανθρώπων που δεν ήταν ύποπτοι για κάτι. Πέθηκαν λοιπόν θέματα προστασίας εδώ του ιδιωτικού βίου και του κατά πόσον οι Σουηδοί θα μπορούσαν να είναι όλοι αντικείμενο παρακολούθησης των συνομιλιών τους. Πολλοί ήταν αυτοί μέλη της κυβέρνησης συγκεκριμένα που εξέφρασαν επικριτικά σχόλια και μέλη του συνασπισμού που κυβερνά τη χώρα και πολλοί βουλευτές που δεν μπορούσαν να δεχτούν σε καμία περίπτωση την πρόταση της κυβέρνηση. Αυτό μεταξύ άλλων οδήγησε σε αναθεώρηση της πρότασης, ε, τροπολογίες και αναθεώρησή της. Πολλές αλλαγές έγιναν και το νομοσχέδιο εγκρίθηκε να το διατρέξω σύντομα για να σας πω τα βασικά του στοιχεία. Τι εργαλεία δηλαδή θεσπίστηκαν και τι ακριβώς εγκρίθηκε για να επιστρέψω μετά στην τωρινή ε, συζήτηση για τα θέματα αυτά στη χώρα μου. Υπάρχει κρατική αρχή, η FIA, η οποία είναι υπεύθυνη για τα σήματα ε, που παρακολουθούνται τις μυστικές υπηρεσίες βάσει της ειδικής νομοθεσίας. Πέραν αυτού του φορέα, είναι και άλλες οι αρχές που κάνουν ε, ελέγχους και παρακολούθηση των θεμάτων αυτών. Η βασική ο βασικός έλεγχος γίνεται από το αρμόδιο δικαστήριο για τα θέματα των μυστικών υπηρεσιών που πρέπει να δώσουν την έγκρισή τους, αλλά υπάρχει και ένας τρίτος φορέας. Η Επιτροπή για τα θέματα άμυνας και μυστικών υπηρεσιών της Σουηδίας, η οποία ε, σε καθημερινή βάση παρακολουθεί, εποπτεύει τις δραστηριότητες αυτές και βεβαιώνεται ότι η FIA ακολουθεί τις συστάσεις του αρμόδιου δικαστηρίου. Οποιαδήποτε έγκριση δοθεί από οποιαδήποτε φορέα έχει εξάμενη διάρκεια και μετά επανεξετάζεται. Και το δικαστήριο αποφασίζει κατά πόσον εθνική αμυντική, η Εθνική Αμυντική Επιτροπή πρέπει να θέσει συγκεκριμένου όρου για την ε, συνέχιση μιας ε, διαδικασίας ή όχι. Ο βασικός κανόνας είναι ότι εάν ο πομπός και ο παραλήπτης βρίσκονται και οι δύο στη Σουηδία, η παρακολούθηση δεν επιτρέπεται. Όμως, ένα μεγάλο μέρος των στοιχείων που ενδιαφέρουν τον Εθνικό Ραδιοφωνικό ε, Φορέα έχει να κάνει με επικοινωνίες που περνούν από τη Σουηδία, από και προς τρίτες χώρες. Είναι μεγάλος ο όγκος των πληροφοριών που μπορεί να εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Χωρίς να ισχύουν αναγκαστικά οι ίδιοι νομικοί περιορισμοί. Τώρα, η Επιτροπή για τα θέματα άμυνας και μυστικών υπηρεσιών δεν καθορίζει μόνο τους όρους διενέργειας τέτοιων διαδικασιών, αλλά και την ε, υποχρέωση υποβολής εκθέσεων ή το κατά πόσο υπάρχουν παραβιάσεις του ιδιωτικού βίου από τις μυστικέ υπηρεσίες. Υπάρχει όμω και άλλη μια αρχή, ένα φορέας που ε, ασχολείται με την ε, εποπτεία του έργου της FIA ένα φορέας ο οποίο ε, κοιτάζει με μεγάλη προσοχή τα ζητήματα ε, ιδιωτικού βίου. Η αρχή για τα προσωπικά δεδομένα. Αυτή είναι πραγματικά η αρχή, ο φορέα, που ασχολείσαι με θέματα του ιδιωτικού βίου, της προστασίας των δεδομένων ε, στο διαδίκτυο και το τι είδου άδεια πρέπει να δίνεται στι διαφορετικέ αρχέ ή του φορεί για να παρακολουθούν τα προσωπικά δεδομένα. Εάν όμως τώρα επιστρέψουμε στο σήμερα και το τι γίνεται αυτή τη στιγμή, υπάρχει αναβρασμός στο Σουηδικό Κοινοβούλιο. Την περασμένη Παρασκευή έγινε μια γενική συζήτηση για το συσχετισμό μεταξύ της ε, NSA και της Σουηδικής FIA. Κατά πρώτον, να πω ότι τα θέματα που συζητούνται αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο ε, καυτά όσο ήταν το 2008 και 2009 πλέον. Ε, τουλάχιστον δεν γίνονται αντιληπτά έτσι. Αυτό που οι Σουηδοί θεωρούν ως πρόβλημα είναι ότι έχουμε αδύναμο, αδύναμη κοινοβουλευτική εποπτεία ως προς τα ζητήματα αυτά. Και πολλές ε, επικρίσεις ακούστηκαν για τα διάφορα παραθυράκια της νομοθεσίας που επιτρέπουν την ε, παρακολούθηση Σουηδών πολιτών στη Σουηδία. Υπάρχει λοιπόν ανασφάλεια, γενικευμένη ανασφάλεια στη Σουηδία για τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και το ποια είναι η κατεύθυνση στην οποία θα έπρεπε να οδεύσουμε. Ε, Ποιε θα ήταν οι καλύτερες... Ε, μέθοδοι για να αποφευθεί κατασκοπία ε, κατά ε, Σουηδών και Ευρωπαίων πολιτών. Αυτές οι ανησυχίες ακούγονται κυρίως γιατί δεν είναι ισχυρή κοινοβουλευτική αποπτία και κοινοβουλευτικός έλεγχος. Μία φορά το χρόνο η, Βουλή, η Σουηδική Βουλή υποχρεούται να εξετάζει τον όγκο των σημάτων που έχουν αξιοποιηθεί από, και έχουν μελετηθεί από την FIA βάσει της νομοθεσίας. Αλλά πάνω απ' όλα στη Σουηδία έχουμε μακρά ιστορία παρακολούθησης και συγκέντρωσης στοιχείων μέσω σημάτων από τις μυστικές υπηρεσίες με πολύ υψηλές τεχνικές γνώσεις και πολύ ισχυρό κλάδο ως προς αυτό. Οι ε, σουηδικές αρχές που είναι υπεύθυνε για την άμυνα και τις μυστικές υπηρεσίες θεωρούν ότι για την άμυνα της χώρας είναι πολύ σημαντικές οι υπηρεσίες αυτές. Και η κυβέρνηση δίνει μεγάλη αξία στις πληροφορίες που συγκεντρώνονται και μπορεί να ε, χρησιμοποιηθούν. Θεωρείται άκρος σημαντικό το θέμα αυτό. Είναι ένα ζήτημα προτεραιότητας. Αυτό ε, εξηγεί εν μέρη γιατί η κυβέρνηση είναι πάντοτε τόσο προσεκτική και γιατί δεν ε, επικρίνει εύκολα τις δραστηριότητες που έχουν ε, λάβει χώρα στις ΗΠΑ. Εγώ, ως μέλος του Κοινοβουλίου, είμαι μέλος της αντιπολίτευσης. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το νέο νόμο για τα ε, σήματα που συγκεντρώνονται τις μασικές υπηρεσίες. Θεωρούμε ότι τίθενται θέματα ιδιωτικού βίου εδώ. και πιστεύουμε ότι τα θέματα αυτά έχουν ε, παραμεληθεί, δεν ε, καλύφθηκαν ως προτεραιότητα μέσω του νόμου δεν ήταν επαρκέ το επίπεδο προστασία των δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων του νόμου που εγκρίθηκε. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο νόμος αυτός πρέπει να αναθεωρηθεί και να γίνει μια νέα πρόταση που να λαμβάνει υπόψη τα θέματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, των προσωπικών ελευθεριών και του ιδιωτικού βίου. Θα πρέπει να βελτιωθεί επίσης η κοινοβουλευτική εποπτεία και ο έλεγχος και να πω εδώ ότι στις συζητήσεις στο Σουηδικό Κοινοβούλιο, ακόμη και οι σοσιαλδημοκράτε τη της Βουλής πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη πλαισίωση ακόμη και της ε, εταιρική ή βιομηχανική κατασκοπία, κυρίως από τρίτε χώρε. Όλα αυτά βεβαίως ε, πυροδοτούνται από τι συζητήσει σε σχέση με την NSA. Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου είναι λιγότερο σαφής και λιγότερο καλή μάλλον όταν προσπαθεί να συγκεντρώσει στήριξη για να υπάρξει ένα θεωρήση αυτής της νομοθεσίας. Βέβαια όσο το νωρίτερο δράσουμε τόσο καλύτερα πριν από το 2010 υπήρχε μια κοινή πλατφόρμα για τους πράσινους, τους αλληλδημοκράτες και τους χριστιανοδημοκράτες για να ζητήσουν αναθεώρηση του νομοσχεδίου από το προτινόμενο ε, και να προωθηθούν τα θέματα ιδιωτικού βίου. Δυστυχώ οι Δημοκράτες αποχώρησαν από αυτό το κίνημα και τελικά ο νόμο αυτό εγκρίθηκε και είναι αυτό που σήμερα δεν μα ικανοποιεί. Θα θέλαμε να γίνουν έστω και μικρέ αλλαγέ στο νόμο, αλλά η πλήρη αναθεώρησή του αρχίζει να γίνεται απίθανη ω προοπτική. Νομίζω ε, σε μια πρώτη φάση αρκούν αυτά, ε, αλλά είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Πάντως, να πω ότι δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Άμυνας, οπότε δεν έχω τέτοια πείρα για να σας απαντήσω σε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. Ε, Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε το πρώτο γύρο ερωταπαντήσεων. Ο κύριο Μωράς, ο εισηγητής μας πρώτα και ο κατόπιν οι σκιώδης εισηγητές. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό εδώ είναι, μετά τα πρώτα σχόλια που ακούσαμε από εσά, είναι ότι προσπαθούμε στην έρευνα αυτή να επιχειρήσουμε κάτι το ανέφικτο ουσιαστικά σε τόσο λίγο χρόνο, γιατί θα πρέπει να έχουμε την έκθεσή μας για το Φεβρουάριο και κάνουμε μια απογραφή των ε, βασικών ε, επίμαχων σημείων και ένα απολογισμό της κατάστασης των μυστικών υπηρεσιών στα κράτη-μέλη. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, σήμερα ε, μιλούμε για την κατάσταση στη Σουηδία και τις κάτω χώρες. Ουσιαστικά παίρνουμε στιγμιότυπα της κατάστασης των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε εξορισμού δεν αποκλείεται να είναι μια τέλεια απογραφή της κατάστασης και σας προσκαλέσαμε ως πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων όχι για να μας δώσετε μια κομματική προσέγγιση αλλά για να μας πείτε κατά πόσο κρίνετε ότι αυτός, αυτή η κοινοβουλευτική εποπτεία ε, είναι αποτελεσματική ή κατά πόσο χρήζει τροποποίησης. Ρωτήσαμε παρόμοιες ερωτήσεις ε, και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ίδιο θα κάνουμε και στις κατοχώρες. Ε, ε, αναφέρθηκαν ε, κατηγορίες για, παρακολούθηση ή για συνεργασία με Δανία, Φιλανδία και ανταλλαγή δεδομένων, προσωπικών δεδομένων. Εσείς ασκήσετε επικρίσεις στο νομικό πλαίσιο. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν και με το νομικό πλαίσιο, υπάρχει πρόβλημα και με την πρακτική. Έχει δυνατότητα η Σουηδική Βουλή να τροποποιήσει την κατάσταση, θα γίνουν μεταρρυθμίσεις Φαντάζομαι και άλλοι συνάδελφοι θα εκφέρουν τη γνώμη. Ποιες είναι οι εξουσίες ε, που έχει η Σουηδική Βουλή ε, και ποια πιστεύετε την είναι η λύση. Νομοθετική αλλαγή, αλλαγή στην έμπρακτη εφαρμογή. Γιατί στην έρευνα αυτή ε, ουσιαστικά κάνουμε μια σύντομη απογραφή της κατάστασης στα κράτη-μέλη. Πείτε μας, ποια είναι η πορεία που πιστεύετε θα πρέπει να ακολουθήσουν οι μεταρρυθμίσεις στη Σουηδία. Κυρία Έριξον, έχετε το λόγο. Μπορούμε να καταστήσουμε πιο αυστηρό το έλεγχο από πολλές απόψεις. Και το δικαστήριο ουσιαστικά δίνει την άδεια σε αυτόν τον οργανισμό για τη συλλογή πληροφοριών από το ηλεκτρονικό φάσμα και πιστεύω ότι η Σουηδική Βουλή θα μπορούσε να ασκήσει καλύτερο έλεγχο στο τι συμβαίνει στους διάφορους οργανισμούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Γιατί ούτε και η Επιτροπή Άμυνας της Σουηδικής Βουλής δεν φαίνεται να έχει έλεγχο της κατάστασης. Οπότε σίγουρα ε, η κατάσταση χρήση βελτίωσης και μάλιστα σημαντικής βελτίωσης. αλλά α, ρυθμίσεις υπάρχουν και διατάξεις κυρίως για την παρακολούθηση Σουηδών στη Σουηδία. Σε ό,τι αφορά την κατασκοπία σε άλλες χώρες η ανταλλαγή δεδομένων, κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να γίνουν κάποιες συμφωνίες. Θα πρότεινα λοιπόν να προσπαθήσουμε οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνήσουν μεταξύ τους ότι δεν θα κατασκοπεύουν η μία την άλλη. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό. Μία συμφωνία αποφυγής αμοιβέ κατασκοπίας. Θα πρέπει να δούμε όμως ποια θα πρέπει να είναι η βάση μιας τέτοιας παρακολούθησης. Επίσης το επόμενο βήμα θα είναι μια συμφωνία μεταξύ των χωρών μελών για αποφύγη κατασκοπίας μεταξύ τους και μετά να πάμε στις ΗΠΑ και να πούμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό συμφωνήσαμε. Να αποφύγουμε μαζική παρακολούθηση των πολιτών, των εταιριών, των πολιτικών και να αποφύγουμε κατασκοπία μεταξύ μας. Και ζητούμε και από εσάς τις Ηνωμένε Πολιτείε να υπογράψετε μαζί μας αντίστοιχη συμφωνία. Είναι θέμα ακεραιότητας πολιτικής. Δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστική μια τέτοια συμφωνία, αλλά θεωρώ ότι αν μη τι άλλο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα, θα πρέπει μεταξύ μας να είμαστε ε, ειλικρινείς και ρεαλιστές. Μιλούμε για κοινή άμυνα μερικές φορές. Αν δεν καταφέρουμε όμως ε, πριν από την κοινή άμυνα να ε, διαθετήσουμε τέτοια θέματα, τότε τα κοινή άμυνα είναι χαζομάρα. Καλά, ας, διαγράψουμε το τελευταίο σχόλιο περί χαζομάρες από τα πρακτικά. Εμείς μπορούμε να διαγράφουμε ό,τι θέλουμε, αλλά σίγουρα η NSA θα το έχει καταγράψει. Ας αφήστε δε που με, μεταδίδεται και από το διαδίκτυο. Γίνεται κοινοβουλευτικό έλεγχος μερικές φορές και πίσω από τις ε, οθόνες. Ε, φαίνεται ότι από τις οθόνες κάνετε παρακολούθηση του ΕΛΚ, γιατί στην αίθουσα δεν βρίσκεται κανένας ε, βουλευτής του ΕΛΚ. Κύριε Όλμπριχτ, παρακαλώ και από εδώ και πέρα χρονοφίδου γιατί, γιατί μένουμε λίγο πίσω όσο περνάει η ώρα. Κύριο Άρμπρεχτ, ναι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο και να εστιάσω σε μερικέ ερωτήσει που μα ενδιαφέρουν έτσι, συγκεκριμένα και οι απόψεις σας. Για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, γνωρίζετε να ενέχονται καθόλου σοηδοί βουλευτές σε μια έρευνα ε, στην οποία συνεργάζονται τα διάφορα κοινοβούλια ως προς τις μυστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ασφαλείας τους. Δηλαδή συμβαίνει τίποτα, υπάρχει συνεργασία μεταξύ διαφορών κοινοβουλίων, υπάρχει κάποιο είδους θεσμική συνεργασία για τον έλεγχο. Και ένα ερώτημα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έχετε ακούσει ποτέ τι είναι το INTSEN. Έχει ε, κανένα συνάδελφό σας ακούσει τι είναι το INTSEN και τι κάνουν και σε ποια νομική βάση. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε καταφατικά. Γιατί φαντάζομαι ότι ξέρω από τώρα την απάντηση. Και ένα τελευταίο, πολύ καλό ε, που σας έχουμε εδώ, γιατί ασχολείστε με συνταγματικά θέματα. Και ε, όταν απευθυνόμαστε στα κράτη-μέλη μας λένε ότι είναι συνταγματικό αυτό το θέμα. Και μιλήστε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα κράτη-μέλη που κατασκοπεύουν το ένα το άλλο. Εσείς λοιπόν ως βουλευτής και μέλος της Συνταγματικής Επιτροπής πώς αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα. Από ό,τι φαίνεται οι νόμοι άλλων κρατών μελών εφαρμόζονται στη δική σας επικράτεια. Π.χ. Ε, ε, ε, όταν η GCHQ επιτίθεται στο διαδίκτυο στη βελγική Belgacom ή στη Google ή στη Yahoo δεν ξέρω αν στη Σουηδία υπάρχει τέτοια υπόθεση, αλλά γνωρίζω ότι ισχύει στη Φιλανδία. Με αυτή την ετεροδικία λοιπόν εσείς πώς το βλέπετε και πώς μπορούν οι βουλευτές σας να το ελέγξουν. Ευχαριστώ. Μπορείτε να είστε εξίσου σύντομος. Some of the questions is no. Ε, ε, η απάντηση σε μερικά από τα ερωτήματα είναι αρνητική, Είναι απλό όχι και σύντομη. Αλλά για το τελευταίο Ένα από τα πράγματα που θέλω να τονίσω είναι ότι θα πρέπει πολύ περισσότερο να προστατεύουμε τις εταιρείες από κυβερνό επιθέσεις ε, από το διαδικτυακό ε, έγκλημα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί πόροι και χρηματικοί και ανθρώπινοι και γενικότεροι που αφιερώνονται εκεί. Και αν θέλουμε ευρωπαϊκές εταιρείες να είναι ανταγωνιστικές θα πρέπει να τις προστατεύουμε καλύτερα από τέτοιου είδους επιθέσεις στο μέλλον πιστεύω. Okay, thank you. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Οι άλλοι δύο σκιώδεις συντηρητικοί και γκουε απουσιάζουν. Οπότε ερχόμαστε σε μένα. Δύο ερωτήσεις. Αναφερθήκατε σε μια ε, της συμφωνίας περί μη κατασκόπευσης, no spy agreement. Αυτό λίγο με προβληματίζει. Είτε είναι νόμιμη κατασκοπία, οπότε δεν χρειάζεται συμφωνία, είτε είναι παράνομη, οπότε γιατί να το συμφωνήσουμε. Τι θα συμφωνήσουμε, δηλαδή ποια θα είναι η προσθέμενη αξία. Δεν θα σου πει μια χώρα ότι σε κατασκοπεύει, εκτός αν την καρφώσει κάποιος. με εξέπληξε αυτό που αναφέρατε για τον ασθενή κοινοβουλευτικό έλεγχο στη Σουηδία. Γιατί πιστεύω ότι ένα από τα πράγματα που μάθαμε σε προηγούμενες συνεδριάσεις ήταν ότι η Σουηδία διαπρέπει στο δίκτυο της τηλεπικοινωνίας και σε όλη αυτή την ιστορία κατασκοπίας και τα δίκτυα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένου Βασιλείου. Δηλαδή ο ισχυρός κοινοβουλευτικός έλεγχος και εποπτεία πιστεύω ότι είναι ακόμα σημαντικότερη στη Σουηδία από ότι σε πολλές χώρες της Ένωσης. Ναι, δίκιο έχετε. Αλλά θα τα συζητήσαμε περί κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αλλά όταν ο νόμος αυτός πέρασε πριν από λίγα χρόνια, αυτά ε, προβλέφθηκαν. Ο νόμος τώρα ήδη εφαρμόζεται εδώ και κάποια χρόνια. Αλλά πιστεύω Οπωσδήποτε ότι πρέπει να ενισχύσουμε το σκέλος του κοινοβουλευτικού ελέγχου για να γίνει το νομικό πλαίσιο ε, αποτελεσματικό όπως αρχικά είχε συλληφθεί στο σχεδιασμό του. Όμως αυτό παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα στη Σουηδία. Έχουμε εκλογές του χρόνου και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα από τα θέματα που θα αποσχολήσουν την προεκλογική περίοδο. Το θέμα βέβαια είναι αν θα γίνει ε, νόμιμο κάτι τέτοιο στη Σουηδία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι. Ε, υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο χοντρικά σε όλες τις χώρες και από τη στιγμή που έρχεσαν οι διεθνείς διαπραγματεύσεις και συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαίων, τέλος πάντων σε άλλα επίπεδα, από τη στιγμή που θα υπάρξει μια συμφωνία σε τέτοια επίπεδα, δεν θα είναι νόμιμη κατασκοπία. Πρόεδρος, Ευχαριστούμε ο κύριος και ο κύριος Κύριε κύριος πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ευκαιρία να μιλήσω και εγώ τη μετρική μου γλώσσα και είναι και ένα θέμα που αφορά τις σχέσεις μεταξύ Σουηδίας και Φιλανδίας αυτό που συζητάμε. το 39 οι Σουηδοί έλεγαν ότι αυτό που είναι σημαντικό για τη Φιλανδία ή που είναι θέμα για τη Φιλανδία, το ίδιο είναι και για τη Σουηδία. Έκτοτε τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά και πλέον φαίνεται ότι ό,τι συμβαίνει στις βαλτικές χώρες είναι αυτό που είναι σημαντικό για την ε, Σουηδία. Έκτοτε έχουμε δει να υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια για το τι γίνεται στις ΗΠΑ μεν, αλλά λιγότερο για το τι μπορεί να κάνει η Σουηδία κατά των γειτονικών της χωρών. Εκεί θα μπορούσαμε να δούμε αν υπάρχουν επικρίσεις ή όχι. Κοιτάξτε, το δίκτυο των, της καλωδιακής και των καλωδίων περνάει από τη Σουηδία για τις χώρες της Βαλτικής. Είναι αλήθεια αυτό. Όχι μόνο από τη Φιλανδία, αλλά, μόνο προς τη Φιλανδία μόνο, αλλά και προς τις υπόλοιπες χώρες της Βαλτικής. Άρα είναι εύστοχη η παρατήρηση που κάνετε. Αλλά εδώ όντω έχουμε να κάνουμε με ζητήματα στρατηγικής σημασίας για τη Σουηδία. Εάν σκεφτούμε σοβαρά την ε, πιθανότητα επίτευξη συμφωνιών μεταξύ Σουηδίας, Φιλανδίας και χωρών της Βαλτικής και σε ευρωπαϊκό επίπεδο βέβαια για το τι επιτρέπεται να ερευνούμε και να είναι αντικείμενο συγκέντρωση πληροφοριών σε αυτό το δίκτυο καλωδίων τότε κατά πόσο θα, θα προκύψει και ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Αλλά προ στιγμή το νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει κανένα περιορισμό για τον οργανισμό συγκέντρωση στοιχείων από το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα και το τι μπορεί να κάνει. Ευχαριστούμε. Κύριο Σάγκστρομ, τελευταίο ομιλητή από το γύρο αυτό των ερωταπαντήσεων. Σα ευχαριστώ. Και εγώ θα αξιοποιήσω τη δυνατότητα που έχουμε να μιλήσουμε σου Θα ήθελα πρώτα να επιβεβαιώσω αυτά που είπατε στην αρχή. Δηλαδή, ότι όταν πέρασε το σχετικό νομοσχέδιο για τον οργανισμό FRA στη Σουηδία έγινε σφοδρή συζήτηση και εντός και εκτός Σουηδίας. Τώρα μπορώ να επιβεβαιώσω ότι όντως είχαμε εκτεταμένη συζήτηση και οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών είναι εξοικειωμένοι με το θέμα της Σουηδίας γιατί αναφέρθηκε πολλές φορές σε ακροάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οχτώ αρχές, αν δεν κάνω λάθος, οχτώ φορείς έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν ε, παρακολούθηση από τον αρμόδιο οργανισμό για τη συλλογή πληροφοριών. Έχουμε ε, τη στρατιωτικές υπηρεσίες, ε, τις υπηρεσίες ασφάλειας, αστυνομία, και η τρίτη ομάδα φορέων είναι κάποια πολιτική, κάποιοι πολιτικοί θεσμοί, η κυβέρνηση, Υπουργικό Συμβούλιο, το Υπουργείο Εξωτερικών συγκεκριμένα. Τώρα, η ερώτησή μου προς εσάς που είστε και πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Αν δείτε τα αιτήματα που βάλλονται στον FRA, ποιο τμήμα αυτών των αιτημάτων είναι από, από στρατιωτικές αρχές, ε, ποιο ποσοστό από, από αστυνομικές και ποιο από πολιτικούς φορείς. Λυπούμε, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση. Όχι γιατί είμαι μυστικοπαθής ε, ή γιατί δεν μπορώ να αποκαλύψω τέτοια στοιχεία, αλλά γιατί δεν γνωρίζω την απάντηση στην ερώτηση που υποβάλλατε. Ωραία, ήσασταν ειλικρινέστατος. Οπότε ολοκληρώνουμε αυτό το γύρο και περνάμε στον επόμενο μας καλεσμένο, τον κύριο Φαντέλντεν, που είναι πρόεδρος της ε, ε, Ολλανδικής Ανεξάρτητης Επιτροπής ε, για τις Μυστικές Υπηρεσίες, που έχει τα αρχικά CTIVD στις κάτω χώρες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ θα εκμεταλλευτώ και εγώ την ευκαιρία που μου δίλετε, τουλάχιστον να αρχίσω στα Ολλανδικά. Θα πω και δύο λόγια στα Αγγλικά, μην ανησυχείτε. Έχω ε, διατελέσει ε, ε, δικαστής πολλά χρόνια και άλλο είναι το δίκαιο στα εγχειρίδια και άλλο το δίκαιο στην πράξη. Law in the books και law in action και το έμπρακτο είναι πολύ πιο σημαντικό. Θα κάνω ένα βήμα πίσω, δεν θα αρχίσω με την εποπτεία ή την επιτήρηση αλλά θέλω να τονίσω ότι πρόκειται για τις ίδιες τις υπηρεσίες, αυτές καθ' αυτές. Στην ε, ε, Ολλανδία είναι δύο, είναι η Γενική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το ένα είναι General και το άλλο είναι Defense, ε, που πάντα ε, ξέρουν ότι θα πρέπει να τηρούν τον νόμο και κάθε φορά που ε, παραβαίνουν το νόμο ε, και μάλλον κάθε φορά που δρούν θα πρέπει να έχουν ε, υπόψη τους την επικουρικότητα, την αναλογικότητα και την αποτελεσματικότητα. Και πάντα γίνονται απαραίτητοι έλεγχοι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προχωρούν σταδιακά. Όταν κάνουν καλά τη δουλειά τους οι μυστικές υπηρεσίες και υπηρεσίε υπηρεσίες πληροφοριών, στο Ολλανδικό σύστημα θέλουν ε, την έγκριση είτε του Υπουργείου ε, Εσωτερικών είτε ε, του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης με υποστήριξη στελεχών που είναι και νομικοί πολλές φορές και μελετούν πάρα πολύ τα αιτήματα και μόνο τότε και μόνο τότε μπορούν να προχωρέσουν σε μια δράση όπως είναι παρακολουθήσει υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, παγιδεύσεις κτλ τότε και μόνο τότε τέλος έρχεται η εποπτεία και η επιτήρηση που σε αυτή την περίπτωση στην Ολλανδία διεξάγεται από την Επιτροπή που συμμετέχω που είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή, όχι κοινοβουλευτική, ούτε πολιτικά διορίζεται, ούτε πολιτικά είναι στρατευμένη, είναι τελείως ανεξάρτητη Επιτροπή Επιτήρησης Υπηρεσιών Πληροφοριών και Ασφαλείας. Έχει απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες των ε, υπηρεσιών. Μπορούμε, έχουμε γραφεία, μπορούμε να κάνουμε login ε, στα συστήματά τους, έχουμε τις ίδιες αρμοδιότητες με τους διευθυντές τους, μπορούμε να παρακολουθούμε και εμείς τα πάντα. Βέβαια μπορούμε να βλέπουμε τα πάντα, αλλά δεν μπορούμε να ανοίγουμε τα πάντα, ε, να, τα, να παρακολουθούμε στην ουσία τους. Ε, γιατί αυτή έχουν ε, εκατοντάδες ε, στελέχη υπαλλήλους και υπηρεσιακούς. Εμείς έχουμε έξι υπαλλήλους και μερικούς εκτάκτους. Πάντως μπορούμε ε, να ελέγχουμε τις υπηρεσίες, κάνουμε εκθέσεις, όλες οι εκθέσεις πηγαίνουν στους αρμόδιους υπουργούς και από εκείνους μετά διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο. Είναι δημόσιες οι εκθέσεις μας αυτές και φροντίζουμε κάθε φορά όταν έχει πάει κάτι στραβά, όταν είναι κάτι παράνομο στις υπηρεσίες να ε, αναφέρεται στις δημόσιες εκθέσεις. Δεν μπορούμε πάντα να μπαίνουμε στην ουσία γιατί υπάρχει πρόβλημα απορρίτου και εμπιστευτικότητας. Πάντως αναφέρουμε ότι κάτι πήγε στραβά. Αυτό το λέμε. Ε, από εκεί και πέρα χρειάζεται και σχεδόν πάντα χρειάζεται ε, κάνουμε και απόρριτες εκθέσεις εκτός από τη δημόσια έκθεση όπου περιγράφουμε λεπτομερώς τι αποκαλύψαμε δεν ε, ε, κρατάμε τίποτα μυστικό και είναι υποχρεωμένες οι υπηρεσίες να λογοδοτούν. Και είναι υποχρεωμένοι να απαντούν στις ερωτήσεις μας και οι υπάλληλοι. Και όλα αυτά τα γράφουμε σε μια έκθεση, η οποία επίσης διαβιβάζεται στους αρμοδίους υπουργούς και από εκείνους στο κοινοβούλιο, αλλά δεν είναι δημόσια, δεν διαβιβάζεται σε όλους τους βουλευτές και αυτό είναι ένα καθόδες ερώτημα πάντα στην Ολλανδική Βολή, αλλά στην αρμόδια υπηρεσία που είναι ξεχωριστή, ε, που είναι η πρόεδροι των πολιτικών ομάδων ε, του, της Κάτω Βουλής ε, και είναι μια ειδική επιτροπή για τις μυστικές υπηρεσίες. Δηλαδή δεν κρατάμε τίποτα κρυφό ή απόρριτο από το Κοινοβούλιο, απλώς δεν έχουν πρόσβαση όλοι οι βουλευτές αυτό. δεν είναι, είναι διαπιστευμένοι. Συγγνώμη, διαβαθμισμένοι. Δέκα ετών είναι αυτή η νομοθεσία και γίνεται μεγάλος λόγος μήπως θα πρέπει να ενισχυθεί η θέση της Επιτροπής μας. Εμείς έχουμε ένα συμβουλευτικό ρόλο και στα έξι χρόνια που συμμετέχω σε αυτή την Επιτροπή διαφωνήσαμε μόνο σε ίσονες ε, περιπτώσεις, ε, όχι σπουδές ε, που θεώρησε ο υπουργό ότι η συμβουλή που του δώσαμε δεν ήταν σωστή και δεν έπρεπε να την ακολουθήσει. Είναι μικρή δηλαδή η σημασία των ενδεχομένων προβλημάτων. Δεν ξέρω αν χρειάζεται αναθεώρηση ολόκληρη τη νομοθεσία. Εγώ περιμένω να ακούσω ε, τι θα βγει, θα ενισχυθεί μάλλον η ε, επιτροπή αυτή και ο ρόλος της θα γίνει περισσότερο δεσμευτικός και όχι συμβουλευτικός. Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες, στην Ολλανδία ξέρετε ότι γίνεται μια πολύ έντονη συζήτηση για τις μαζικές παρακολουθήσεις και υποκλοπές μετά από το σκάνδαλο NSA και γίνεται μια προσπάθεια από τη Βουλή με εξεταστική επιτροπή Τώρα είναι πολύ νωρίς, δυστυχώς ε, αρχές Δεκεμβρίου θα έχουμε ολοκληρώσει την έρευνά μας και αρχές Ιανουαρίου θα διαβιβαστούν όλα αυτά στην Ολλανδική Βουλή και θα πούμε τι ανακαλύψαμε ή τι δεν ανακαλύψαμε και τι μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε. Γίνεται αυτή η συζήτηση στην Ολλανδία πραγματικά και το σημαντικό είναι ότι μέχρι τώρα μπορούν να Ε, παρακολουθούν ε, ότι δεν ε, συνδέεται με καλώδια. Ότι, μπορούν να παρακολουθούν ότι είναι κύματα, α πούμε, και κυκλοφορεί στον αέρα. Αλλά στα μεταξύ περισσότερε ανταλλαγέ πληροφοριών και συνεννοήσει και επικοινωνίε γίνονται με καλώδια και πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσουν αυτή τη δυνατότητα οι υπηρεσίε. Μπορεί αυτό να σα φαίνεται ιδιαίτερα επεμβατικό ε, αλλά προσωπικά θεωρώ ότι Εντάξει, μπορεί κανείς να παρακολουθεί μαζικά, μετά πρέπει να επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες. Ε, ε οι πληροφορίες αυτές ε, έχουν να κάνουν με στοχευμένα νούμερα, τηλεφωνικά, ε, συνδιαλέξεις, διευθύνσεις ε, αυτό είναι μια αρμοδιότητα που δίνεται από τους αρμόδιους υπουργούς ε, στις υπηρεσίες. Δεν γίνεται αδιάκριτα. Υπάρχει διακριτική ευκαιρία, υπάρχει έλεγχος και αρκετά καλός, αλλά τώρα έχει αργήσει η συζήτηση και για την οτροπία που επικρατεί στις μυστικές υπηρεσίες. Σήμερα υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες και είναι ενδιαφέρον για διεθνή συνεργασία και για την επιτήρηση και την υποπτήρα, ε, είναι μικρές αυτές. Κάθε δύο χρόνια γίνεται μια διάσκεψη μιας ε, επιτροπής ε, που επιτηρεί τις μυστικές υπηρεσίες. Οι αγγλοσαξονικές χώρες συμμετέχουν εκεί και το Βέλγιο και οι κατοχώρες, αλλά κάθε χώρα ελέγχει το δικό της σύστημα και μόνο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε ανταλλαγές. Συζητούμε γενικά και αόριστα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταλλάξουμε πληροφορίες με τις Ηνωμένε Πολιτείε το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν μας λένε τι κάνουν στις υπηρεσίες τους. Το ίδιο ισχύει και για μένα, δεν μπορώ να απαντήσω σε όποιο με ρωτάει για τις υπηρεσίε ε, ε, Και πόσο μάλλον για δράση υπηρεσιών άλλων κρατών. Σταματώ εδώ και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Μωράς. Ευχαριστώ. Όπως είπα και προηγουμένως τον κύριο Έριξον, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις και να κάνουμε μια σύντομη υπογραφή της κατάστασης ε, των μυστικών υπηρεσιών στις επιμέρους χώρες μέλη, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν κάποια προβλήματα. Μας κάνατε μια επισκόπηση της κατάστασης κάτω χώρες και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Αλλά πρόσφατα σε μια συνέντευξη μιλήσατε για ένα νέο σύστημα, είναι ένα νέο λογισμικό που ετοιμάζεται ή τουλάχιστον αυτό αναφέρθηκε, αυτό κατάλαβα από τη συνέντευξη που δώσατε. Μπορείτε να μας ε, διευκρινίσετε αυτό το θέμα, γιατί ίσως δοθούν περισσότερες ε, ε, ευκαιρίες έτσι, στις μυστικές υπηρεσίες. Αν συμβεί κάτι αυτό, υπάρχει μια τέτοια αναβάθμιση, πώς εσείς ε, θα καλύψετε το έδαφος, γιατί... Η συμφωνία για τα εννέα μάτια Είπαμε και αυτό ακούστηκε στις αρχικές αποκαλύψεις για την NSA και τις κατηγορίες για μασικές παρακολουθήσεις. Και μάλιστα αναφέρθηκε και ανάμειξη κοινοτικών χωρών. Ποια ήταν η δική σας εντύπωση, γιατί και εσείς συμμετέχετε στη Συμφωνία των Εννέα Ματιών, οπότε μας ενδιαφέρει και η θέση της Επιτροπής σας με τα τις αποκαλύψεις που έγιναν για την NSA. Κύριε Βαντέλταν, αυτό το νέο σύστημα που ίσως ε, τεθεί σε εφαρμογή στο μέλλον δεν είναι ακόμη σίγουρο πώς θα λειτουργήσει. Και αυτό του άλλους δεν μας αφορά, δεν αφορά την Επιτροπή μας, αφορά μόνο το Υπουργείο και τις υπηρεσίες. Εμείς απλώς θα κάνουμε μια υποπτία, θα σκίσουμε μια υποπτία στο έργο τους. Φαίνεται ότι είναι καταπληκτικό το σύστημα, αυτό ισχυρίζεται τουλάχιστον η Αρμόδη. Εμείς θα τηρήσουμε τον νόμο και τις νομικές δυνατότητες που προσφέρει. Αυτό είναι και το δικό μας Σε Ό,τι αφορά τα εννέα μάτια, θα ακούσετε τον Υπουργό Εσωτερικού που είπε ότι δεν μπορώ να σας πω αν αν έχει προσυπογράψει την οδηγία για τα εννέα μάτια. Μπορεί και να συμμετέχει και η Ελλαδία στην συμφωνία αυτή, μπορεί και όχι όμως σε ό,τι αφορά την NSA, πριν από μια-δυο εβδομάδες έδωσα μια διάλεξη ε, και συμμετείχε και ο Κιθ Αλεξάνδερ. Ήμουν μόνος με ένα κόμπι μέλος ε, της Επιτροπής. Ένα κύριος είχε 10-12 ε, ανθρώπους επιτελείου και μας είπε δεν μας ενδιαφέρουν οι κατοχώρες γιατί εσείς δεν έχετε καμία πληροφορία. Αυτό το ε, έγινε πριν μάθουμε πόσες υποκλοπές είχα γίνει στο μεταξύ. Και παρόλα αυτά ήταν ένα πολύ μικρό ποσοστό το συνολικό αριθμό των υποκλοπών που είχαν γίνει και της λαθροσύνδεσης του tapping. Τώρα, αν είναι πραγματικά σοβαρή κατάσταση, τι διαστάσεις έχει, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Δεν θα αναφέρω πια τους απόντες, ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς ευχαριστώ που ήρθατε. Ε, η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξή. Είδατε τα έγγραφα που αποκάλυψε ο κύριος Νόντεν. Διότι αυτά αποδεικνύουν αναντήρητα αυτά που λέμε. Ε, Άρα θα περίμενα να γνωρίζετε το περιεχόμενο, δεν αντιφάσκεται στις απαντήσεις σας με το περιεχόμενο τουλάχιστον των εγγράφων που εμείς ε, γνωρίζουμε. Για τις πρώτες με τώρα που είχα θέσει και στον κύριο Έριξον δηλαδή, για να επανέλθω σε αυτές. Ως Επιτροπή πώς ε, συζητάτε το θέμα ότι υπάρχουν ε, κατάφορες παραδιάσεις στην επικράτεια του δικού σας κράτους από κυβερνό επιθέσεις της NSA ή της GCHQ ασχολείστε με αυτά, κάνετε κάποια έρευνα. Αυτά είναι θέματα που μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε. Τι κάνουν οι βουλευτές στη χώρα σας γι' αυτά. Και έπειτα γνωρίζετε αν υπάρχει κάποια συνεργασία μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων για θέματα εποπτείας της, των δράσεων των μυστικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. Γνωρίζετε την Ίνσεν. Τι κάνουν, ποια είναι η βάση του έργου τους. Και επίσης άκουσα ότι υπάρχει κάποιος στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα που είπε στον τύπο ότι τόσες παγιδεύσεις που κάνουμε δεν ξέρουμε τι να τις πρωτοκάνουμε. Άρα ε, υπάρχει εντατικοποίηση της συλλογής, συλλογής δεδομένων και πληροφοριών αυτή τη στιγμή. Τι κάνουν γι' αυτό οι βουλευτές. Να αρχίσω από το τέλος. Υπάρχει αυστηρή διάκριση στο σύστημα της Ολλανδίας. Για τις ποινικέ ε, διαδικασίες και τις ε, αστικές διαδικασίες τις διαδικασίες ασφαλείας. Ε, συμφωνώ μαζί σα ότι είναι υπέρμετρες οι παγιδεύσεις που γίνονται και οι υποκλοπές, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται σε ποινικέ υποθέσεις. Τώρα για τα έγγραφα που έχουν δημοσιευτεί με τον Αλεξάνδερ. Αυτό που είχα πει ήταν ότι δεν ξέραμε ως τότε τι γίνεται με τον ε, Σνόντεν. Δεν μπορούσα να απαντήσω κιόλας γιατί τότε δεν είχα καμία σχέση με το τι γίνεται στην Ολλανδία. Δημοσιεύτηκαν μια εβδομάδα μετά. Ε, αν τα γνώριζαμε από πριν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αυτά μπορώ να σας απαντήσω προς τη μήνυ. If Πρόεδρος, θέλετε να προσθέσει κάτι. Έχετε δέκα δεύτερα και μικρόφωνο. Την ίντσετ δεν την έχετε ακουστά. Ούτε για τη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια ξέρετε τίποτα. Μα πρέπει να περιμένετε την έκθεση. Την εκπονούμε αυτό το καιρό. Δεν μπορώ να σας πω από τώρα τι θα γράφει η έκθεση, γιατί πρώτα πρέπει να αναφέρουμε στο κοινοβούλιο μας. Thank you. Okay. Don't, uh, I give... ε, ναι, ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον εαυτό μου, ως και όδη των φιλελευθέρων, πριν πάμε στα άλλα μέλη, να τα πω και ολλανδικά στη μητρική μου που δεν το πράττω συχνά εδώ στο Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα είπατε ότι υπάρχει αναλογικότητα, η σκοπιμότητα και η επικορικότητα. Γνωρίζουμε ότι είναι παγκόσμιο πρωταθλητής στις παρακολουθήσει και στις υποκλοπές τηλεφώνων η Ολλανδία. Τα θεωρείτε όλα αυτά αναλογικά. Και είπατε ότι όταν είναι δυσανάλογα ε, αυτά που γίνονται ε, αφορούν ποινικέ υποθέσεις. Μα τα τελευταία χρόνια αυτή η διαχωριστική γραμμή μεταξύ μυστικών υπηρεσιών και ε, ποινικών υποθέσεων έχει διαταραχθεί, ιδιαίτερα και ως προς την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Είπε ο Μωράες και διάβασα κι εγώ με τρόμο με έκπληξη εν πάση περιπτώσει στον τύπο αυτά που είπατε το Υπουργείο Αμήνης ε, αγοράζει παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό που απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει. Και μας λέτε ότι ποντάρουμε στην οτροπία των μυστικών υπηρεσιών για να υπάρχει μια αυτοπιθαρχία. Ποια αυτοπιθαρχία. Μπορώ να φανταστώ ε, τι θα γίνει. Αυτό δεν σας ανησυχεί. Και μια άλλη ερώτηση, τρίτη και προτελευταία κατά τη δική σας αίσθηση η εποπτεία και επιτήρηση των μυστικών υπηρεσιών στην Ολλανδία πηγαίνει καλά και λειτουργεί. Γιατί έχω την αίσθηση εγώ ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλιώς θα είχαμε αποφύγει αυτό που αποκάλυψε τώρα ο κύριος Σνόουντεν. Γιατί σας κάνει να πιστεύετε ότι στην Ολλανδία λειτουργούν καλά τα πράγματα ενώ δεν λειτουργούν καλά σε κοντά πολιτείες. Και ε, τώρα για τη μαζική ε, παρακολούθηση, τι είναι σκόπιμο, τι είναι ε, χρήσιμο και τι όχι. Υπάρχει αυτό το λεγόμενο chilling effect. Δικηγόροι, δημοσιογράφοι, whistleblowers, ακόμα και πολιτικοί ε, θεωρούν ε, ότι μπορούν να τους παρακολουθούν. Οπότε δεν μπορούν να εκφράζονται και να επικοινωνούν ελεύθερα, δημοκρατικά, ακριβώς επειδή υπάρχει όλη αυτή η άχρηστη παρακολούθηση και το φακέλωμα το μαζικό. Δεν κινδυνεύει το κράτος δικαίου και η δημοκρατία από όλα αυτά. Η άσκοπη παρακολούθηση και οι υποκλοπές οι δυσανάλογες είναι μεγάλος κίνδυνος μεν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ε, ότι γίνεται ε, σύγχυση, τουλάχιστον στην Ολλανδία, μεταξύ των ποινικών υποθέσεων και των ε, υπηρεσιών ε, πληροφοριών. Δεν υπάρχει υπέρμετρη και ανόητη και υπερβολική παρακολούθηση. Εγώ το ξέρω γιατί βλέπω όλες τις παρακολουθήσεις, τις τηλεφωνικές παγιδεύσεις, τους κοριούς, σε πάση περιπτώσει. Μπορούμε να κάνουμε έλεγχο εκεί, υπάρχει δυνατότητα τεχνική ε, και όταν βλέπουμε ότι παρακολουθούνται κάποιος μακρον ή ε, οι συνακροάσεις αφορούν διάφορα άσχετα πράγματα, τα θέτουμε υπόψη των υπουργών και είναι σε πάρα πολύ περιορισμένη κλίμακα μπορώ να σας πω. Κάτι ε, για το ε, λογισμικό αυτό, το spyware, ε, αν αγοράστηκε ή όχι, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην αγορά ενός συστήματος και στη χρήση του. Και μπορεί να είναι και μια κακή αγορά, κακή προμήθεια που κόστισε μερικά εκατομμύρια ευρώ. Απλώς το έχουν εκεί και το έχουν έτοιμο, αν αλλάξει ο νόμος μήπως το χρησιμοποιήσουν. Ε, αν αλλάξει η νομοθεσία θα δούμε. Σε περίπτωση ε, που δεν το επιτρέψει ο νόμος, μην θα φροντίσουμε να μην χρησιμοποιηθεί. Να το ε, αποτρέψουμε ή θα το γράψουμε. Τώρα αν η επιτήρηση η εποπτεία λειτουργεί, τι να σας πω. Εγώ μπορώ να σας πω για τη χώρα μου. κάθε χώρα μπορεί να κοιτάξει μόνο το δικό της σύστημα. Το τι κάνουν οι Αμερικανοί ή άλλες χώρες γύρω από την Ολλανδία ή στην επικράτεια της Ολλανδίας δεν το βλέπουμε εμείς. Εμείς δεν έχουμε υποπτία σε αυτό. Αλλά αφή στιγμή περιέλθει σε γνώση αυτό των μυστικών μας υπηρεσιών, δηλαδή ότι κάποιες άλλες χώρες κατασκοπεύουν χωρίς να έχουν ενημερώσει την Ολλανδική υπηρεσία, λαμβάνονται μέτρα. Είτε είναι αμερικανικές, βελγικές, φιλανδικές μυστικές υπηρεσίες, δεν μας ενδιαφέρει. Υπήρξαν και παραδείγματα και αποσύρθηκε και η υπηρεσία που έκανε διάφορα πράγματα που δεν συνάδουν με τον τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας των μυστικών υπηρεσιών. Αυτό θα ίσχυε και αν είχαν μπει στο SWIFT οι Αμερικανοί ή οι Βρετανοί. Ναι, αν γίνει κάτι τέτοιο και αποκαλυφθεί, βεβαίω. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί από τους servers βρίσκονται αλλού, <laughs> πανταχού της γης. Δηλαδή ένα σερβερ που κάποιος νομίζει ότι βρίσκεται στην Ολλανδία, βρίσκεται σε ένα τελείως διαφορετικό μέρος δεν αφορά την Ολλανδία αυτό το πράγμα, αλλά αν συμβαίνει κάτι στις κάτω χώρες θα πρέπει να υπάρχει και απόδειξη ότι παραβιάστηκε ένας νόμος ή υπήρξε μια άλλη ε, παράνομη δραστηριότητα. Η κυρία Ζίπελ, η κυρία Σαρχεντίνη, άλλος κανείς, αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις, έχω σχετικά σύντομες και απλές. Είπατε ότι ε, γράφετε τακτικά εκθέσεις για τις δραστηριότητες των ε, ε, υπηρεσιών. Η Επιτροπή σας συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν έρθει κάποιος και σας πει πρέπει να ασχοληθούμε με την τάδε περίπτωση. Και επίσης κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ερευνών που κάνουμε ακούσαμε επανειλημμένα ότι δεν μπορείτε να ε, ότι μάλλον δεν γίνονται συνακροάσεις για τα πάντα, ούτε παρακολουθούν όλες τις συνδιαλέξεις, αλλά ότι υπάρχουν λέξεις κλειδιά. Και ποιος το ορίζει αυτό. Μπορείτε να το πείτε αυτό για την Ολλανδία και αρκεί να υπάρχει στην επικοινωνία μία λέξη κλειδί για να με παρακολουθήσουν, για να υπάρχει συνακρόαση ή είναι συνδυασμός διαφόρων λέξεων ή παρακολουθούνται και συμπεριφορές και ήθη και έθιμα και συνήθειες. Και πόσες είναι αυτές οι λέξεις κλειδιά σήμερα στις οποίες βασίζεται η συνακρόαση και παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Α, να τα πω Ολλανδικά τώρα που άρχισα. Υπάρχει τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών. Αυτό ε, συμβαίνει παγίως με άλλες υπηρεσίες περισσότερο, πιο συχνά με άλλες λιγότερο και οι Ολλανδικές υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να έχουν τακτική ε, ανταλλαγή πληροφοριών ε, μαζί μας για να δούμε αν υπάρχουν πρότυπα που τηρούν κάποιες υπηρεσίες, αλλιώς δεν μπορούν να συνεργαστούν μαζί τους. Τώρα, ε, οι λέξεις κλειδιά στις οποίες αναφερθήκατε Υπάρχουν διάφορες λίστες, κατάλογοι ολόκληροι. Δεν τους γράφουμε εμείς, τους βλέπουμε, μπορούμε να βάλουμε σχόλια, μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν έχει νόημα και να σβηστεί αυτή η λέξη. Επιπλέον αυτοί οι κατάλογοι ε, πολύ συστηματικά και πολύ τακτικά ε, υφίστανται επεξεργασία, κάθε αναδίμηνο. Αλλιώς ε, ασχολούμαστε με άσκοπα πράγματα. Ε, έχουμε όντως τακτική συνεργασία ε, και στις εκθέσεις λέμε ότι πολλές από αυτές τις λέξεις κλειδιά παρά είναι γενικές και ε, αόριστες και θα πρέπει να είναι πιο εστιασμένη παρακολούθηση. Ευχαριστώ κυρία Σαρχεντίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Φαντέλντεν, θα ήθελα να μπω ε, λίγο στην συνέντευξη που δώσατε στην εφημερίδα Volkskrant το Σαββατοκυριακό, το είπε και ο κύριος Μωράης και η πρόεδρος, όπου λέτε ότι οι Ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών θέλουν να αγοράσουν ένα νέο σύστημα ε, κατασκοπίας, δεν παραθέτω επιλέξει, ερμηνεύω αυτά που είπατε, που ακόμα είναι άχρηστα σε μεγάλο βαθμό, αλλά είπατε ότι ο νόμος είναι ε, ξεπερασμένος και είπατε ότι η αγορά ενός συστήματος δεν σημαίνει κατά ανάγκη ε, και τη χρήση τους. Ναι, αυτό ισχύει και για το φύρα, το τρένο υψηλή ταχύτητας που πήγε στραβά στην Ολλανδία, η υπερταχή αυτή, ή το ε, JSF, ε, το καινούριο καταδιοκτικό πολεμικό αεροσκάφος, περίεργη είναι αυτή η παρατήρηση ότι άλλο είναι να αγοράζει ένα σύστημα και άλλο να το χρησιμοποιείς. Ε, τότε γιατί το αγοράζεις και γιατί θεωρείτε ότι είναι απαρχιωμένη η νομοθεσία και για ποιο λόγο οι ολλαδικές μυστικές υπηρεσίες να πάνε να αγοράσουν αυτό το λογισμικό ε, ποντάροντας στην αλλαγή του νόμου. Και κάτι άλλο, σας άκουσα να ε, δίνετε μια κρίση και μια αξιολόγηση για τις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούνται, αν είναι πολύ αόριστες ή πολύ ε, γενικές και δεν έχει νόημα η παρακολούθηση. Στην αρχή του έτους ε, βγήκε μια έκθεση δική σας για την ε, άκρα αριστερά ή για τον αριστερό εξτρεμισμό. Εσείς θεωρείτε ότι είναι σκόπιμο να παρακολουθούνται αυτοί οι άνθρωποι και για ποιο λόγο. Ε, ευχαριστώ για την ομοθεσία γιατί πιστεύω ότι είναι ξεπερασμένη. Αυτό έχει να κάνει ε, με τις καλωδιακές σημείες επικοινωνίες. Αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται στην Ολλανδία ότι μπορούν να παρακολουθούν σε μεγάλο βαθμό ε, τις επικοινωνίες που γίνονται με ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Έχει αλλάξει όμως τώρα η κατάσταση και το 90% είναι καλωδιακή. Αυτό είναι το θέμα και είναι περίεργη η κατάσταση να μην ε, ρυθμίζεται δια νόμου. Και στο παρελθόν, στο ποινικό δίκαιο πριν από 40 χρόνια, η αστυνομία μπορούσε να παρακολουθεί τα τηλέφωνα, αλλά όχι τα τέλεξ. Ε, οπότε καταλαβαίνετε ότι πολλοί ε, μιλούσαν στο τηλέφωνο και λέγανε «Λοιπόν, πάω στο τέλεξ τώρα να σου πω τα υπόλοιπα» και η αστυνομία δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τα τέλεξ. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Ε, και η Επιτροπή μου πραγματικά θα γνωμοδοτήσει για να επεκταθεί το σύστημα και στις καλωδιακές επικοινωνίες. Να μην γίνεται διάκριση μεταξύ ε, κυμάτων ηλεκτρομαγνητικών ας πούμε και καλωδίων γιατί μπορούν σήμερα να παρακολουθούν ό,τι κυκλοφορεί στον αέρα και όχι ό,τι μεταδίδεται με καλώδια. Ε, τώρα, για το αν είναι άσκοπο, άχρηστο κάτι ή αν έχει νόημα, μπορεί να έχω την προσωπική μου άποψη, αλλά αυτό δεν αφορά την Επιτροπή μου. Εμείς κοιτούμε ε, αποκλειστικά ε, το νόμιμο και όχι το σκόπιμο. Δεν μας απασχολεί κάτι τέτοιο προς Θεού δεν μας έχουν συστήσει γι' αυτό και δεν ασχολούμαστε καθόλου με τη σκοπιμότητα παρά μόνο με την νομιμότητα μιας δράσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φαντέλτεν. Ε, πραγματικά αυτό που είπατε για το τέλεξ το είχα πει και εγώ σε μια συζήτηση με κάποιους ασκούμενους και με ρώτησε ένας ασκούμενος τέλεξ τι είναι αυτό. <laughs> You know, in the future someone will say, what's a smartphone? Σε λίγο στο μέλλον μπορεί κάποιος να μας ρωτήσει smartphone, τι είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε και αυτό το τμήμα της δημόσιας ακρόσης, μόνο με 7 λεπτή καθυστέρηση, γι' αυτό και προχωρώ κάθεκτα στο τελευταίο τμήμα, προσκαλώντας την κυρία Μπέλ, τον κύριο Λούντμπλατ και τον κύριο Άλαντ από τη Microsoft, τη Google και το Facebook για το τελευταίο τμήμα της δημόσιας ακρόσης. Okay, colleagues, we continue. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε και περνάμε στο τρίτο τμήμα της ακρόασης. Καλωσορίζω τους εκπροσώπους ε, της Microsoft, της Google και του Facebook. Η, με την Apple συναντηθήκαμε στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα και η Apple μας έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής 6 Νοεμβρίου. Προσκαλέσαμε και τη Yahoo και την Amazon, αλλά αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στην ε, δημόσια κράση, ε, στέρνοντας επιστολές ε, στις οποίες αιτιολογούν αυτή την άρνηση και αν δεν κάνω λάθος έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής μας. Είναι περίτω να σας πω γιατί έχουμε καλέσει και εκπροσώπους του κλάδου, των εταιριών ε, πληροφοριών και τεχνολογιών των πληροφοριών. Θα ήθελα να ζητήσω από τους καλεσμένους μας να κάνουν σύντομες εισαγωγικέ ε, ομιλίες, το πολύ δεκάλεπτο ο καθένας. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Μπέλτς και μετά στον κύριο Λούντπλαντ και στον κύριο Άλαν. Κυρία Μπέλτς, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην σημερινή ακρόαση και εκτιμώ ιδιαίτερα στην ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω στο, στην Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι ο διάλογος είναι ο καλύτερος τρόπος ε, για να προχωρήσει η συζήτηση και να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της εθνικής ασφάλειας και της ιδιωτικής σφαίρας και της ιδιωτικής ζωής στον ψηφιακό κόσμο η ισορροπία αυτή και η ανέβρεσή τη είναι απαραίτητη. Γι' αυτό και χρειάζονται μερικέ μεταρρυθμίσει μερικέ φορέ. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρία θέματα. τι πρακτικέ τη Microsoft, σε ό,τι αφορά τις αιτήσει ε, παροχής δεδομένων από διάφορες κυβερνήσεις. Δεύτερον, ε, η εξασφάλιση των δεδομένων των πελατών και η προστασία ε, των δεδομένων των πελατών από ανεπιθύμητη πρόσβαση. Και τρίτον, τι μπορεί να κάνει η Microsoft ώστε να εξασφαλίσει η προστασία των δεδομένων των πελατών της παντού στον κόσμο. Πριν μιλήσουμε λοιπόν για τις πρακτικές και το πώς ανταποκρινόμαστε στις αιτήσει δημοσίων αρχών στις ΗΠΑ, ΗΠΑ και αλλού για δεδομένων. Θα ήθελα να σα πω δύο λόγια για το ρόλο που παίζει η Microsoft ε, ω εταιρεία ε, και τι υπηρεσίε και τα προϊόντα τη. Ε, ο όγκος και η περιπλοκή των πληροφοριών και των δεδομένων που συγκεντρώνουμε είναι μεγάλο και γι' αυτό υπάρχει μια σύγχυση είναι προς το κοινό μας συμφέρον να κατανοήσουμε καλά τα πραγματικά περιστατικά για να μπορέσουμε να βρούμε και τις σωστές λύσεις. Η Microsoft λοιπόν είναι γνωστό ότι προσφέρει μεγάλο φάσμα υπηρεσιών, ε, συσκευών και λογισμικά στα Windows και Office ε, δίνουμε διάφορες ε, λύσεις, αλλά και στο cloud, στην εφοή υπολογιστική. Έχουμε Xbox, Apple, Mobile Technologies, συστήματα αναζήτησης, online ε, tools και έχουμε και συσκευές. Και επίσης ε, το Νοέμβριο του 2011 ε, αγοράσαμε και το Skype που βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης. Κατά την προσφορά των υπηρεσιών μας στους πελάτες μας, όπως το Hotmail ή το Office 365, έχουμε, χειριζόμαστε και τις αιτήσει των κυβερνήσεων και προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις υποδομές των διακομιστών μας ε, έναντι ανεπιθύμητων προσβάσεων. Έχουμε δημόσιους ε, providers, ε, παρόχους υπηρεσιών, δεν έχουμε τα δικά μας δίκτυα, προκειμένου να προστατεύσουμε τα δεδομένα των πελατών μας και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς έχουμε διάφορες λύσεις προστασίας για να αποφεύγονται οι παρεμβολές. Και μάλιστα χρειάζονται άδειες για τη χρήση των υπηρεσιών ε, από τους παρόχους και οι πάροχοι υπηρεσιών ελέγχουν την πρόσβαση στα δεδομένα. Εμείς βοηθούμε τους πελάτες μας να προστατευτούν ε, έναντι ανεπιθύμητων ε, παρεμβάσεων και κυβερνοεπιθέσεων. Τώρα, πώς ε, χειριζόμαστε αιτήσει για πρόσβαση σε δεδομένα. Η Microsoft ε, δίνει στοιχεία δεδομένων ε, πελατών μόνο σε συγκεκριμένους φορείς μετά από έλεγχο και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες με εξαίρεση συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου το Αμερικανικό Δίκαιο αποδεί, αποκλείει την χορήγηση τέτοιων στοιχείων. Η Microsoft δεν δίνει σε καμία κυβέρνηση στον κόσμο άμεση ή έμεση πρόσβαση σε δεδομένα πελατών ούτε δίνουμε τεχνικές ε, λεπτομέρειες σε κυβερνήσεις ε, ώστε να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα ε, πελατών. Οπότε δεν έχουμε κερκόπορτες στα προϊόντα μας, στις υπηρεσίες μας και ούτε δίνουμε κωδικούς κρυπτογράφηση σε κυβέρνηση. Δεν τους βοηθούμε να σπάσουν τέτοιους κωδικούς. Τώρα, όταν λαμβάνουμε ένα αίτημα από μια κυβέρνηση, ποια είναι η διαδικασία. Καταρχήν, δεν επιτρέπεται να επιβεβαιώσουμε ποιες μυστικές υπηρεσίες μας έχουν απονείμει τέτοιες αιτήσει. Ε, τηρούμε τον νόμο, δεν μπορούμε να σας δώσουμε τέτοια στοιχεία. Αλλά μπορώ να σας εξηγήσω με λεπτομέρεια πώς ε, ε, χειριζόμαστε τέτοιες αιτήσει από μυστικές υπηρεσίες ή αστυνομικέ αρχές. Όταν λαμβάνουμε μια τέτοια αίτηση, έχουμε μια ομάδα συμμόρφωσης που εξετάζει αυτή την αίτηση προκειμένου να, είναι, να δούμε αν είναι παραδεκτή και απορρίπτουμε αυτές που δεν είναι νομότυπες. Και παραλαμβάνω μόνο για συγκεκριμένα δεδομένα που αναφέρονται στο, στο αίτημα. Η Microsoft, Microsoft μόνο συγκεντρώνει και μετά δίνει τα στοιχεία δεν δίνουμε εμείς πρόσβαση ε, σε έναν διακομιστή για να εξετάσει ε, ο φορές που το ζητάει τα στοιχεία. Εμείς κάνουμε την έρευνα και ε, χορηγούμε τα συγκεκριμένα δεδομένα. Επίσης δημοσιεύονται πληροφορίες σε σχέση με αιτήσει που δόθηκαν και για πρώτη φορά περιλάβαμε το συνολικό όγκο ετοιμάτων της εθνικής ασφάλειας που περιλαμβάνουν και κάποιες ε, βιντάλματα για βίζα και δεν μπορούμε να ε, ε, τις μάλλον δεν, έχουμε, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε να έχουμε λάβει και από τη φύσα τέτοιες αιτήσει. Και μάλιστα τον 31 Δεκεμβρίου του 2012 είχαμε λάβει μέχρι 6 με χιλιάδες εντάλματα κλητεύσεις ε, ποινικού χαρακτήρα για 31.000 ε, ε, λογαριασμούς από κυβερνητικούς φορείς των Ηνωμένων Πολιτειών, από, τοπικές, από τοπικούς φορείς, φορείς πολιτιών ή και κυβερνητικούς φορείς. Αυτά βρίσκονται και στα συγκεντρωτικά στοιχεία που χορηγούμε σε ό,τι αφορά τα αιτήματα αστυνομικών αρχών, απορρίπτουμε αιτήματα εφόσον έχουμε μια νομική βάση για τέτοια απόρριψη. Για παράδειγμα, κατά το πρώτο εξάμεινο του 2013 απορρίψαμε 911 τέτοιε αιτήσει, δηλαδή 2,4% των συνολικών αιτήσεων εξαιτία τη μη εκπλήρωση των νομικών ε, ε, προϋποθέσεων. Το, στο 90% των περιπτώσεων τα στοιχεία που ζητούσαν δεν τα είχαμε, άρα δεν μπορούσαμε να δώσουμε τίποτα. Επίσης, ε, απαντούμε για συγκεκριμένους ε, λογαριασμούς και όχι, δεν προσφέρουμε αδιάκριτη πρόσβαση στα δεδομένα. Επίσης, ε, καταγράφουμε τα αιτήματα και αποκαλύπτουμε στοιχεία μόνο, για τα, μόνο εφόσον αναφέρονται στο συγκεκριμένο ένταλμα ή το αίτημα. Ε, και οι εθνικοί φορείς θα πρέπει να τηρούν τις, τους κανόνες για την υποβολή τέτοιων αιτήσεων με βάση ποινικές διαδικασίες. Εμείς φροντίζουμε να είμαστε διαφανείς, να, να συμμορφωνόμαστε με τον νόμο και να επεξεργαζόμαστε νομότυπα όλες αυτές τις αιτήσει. Τώρα δεύτερον, πώς εξασφαλίζουμε την προστασία των δεδομένων των πελατών. Κάνουμε διάφορες προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων, τεχνικά μέτρα, υλικά μέτρα. Ένα που αναφέρθηκε στη συζήτηση είναι η, η κρυπτογράφηση, ε, η κωδικοποίηση. Ε, επίσης, ε, παράταση των κωδίκων έγκρισης και γενικώ υψηλό βαθμός κωδικοποίησης. Επίσης, έχουμε ε, λάβει πολλέ πληροφορίες από τα μέσα μαζική ενημέρωση, Γι' αυτό και προσπαθούμε να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας και να δούμε αν χρειάζονται κάποιες τεχνικές ε, προσαρμογέ για να βελτιώσουμε την ασφάλεια των δεδομένων των πελατών μας και των καταναλωτών. Τρίτον, τι κάνουμε ώστε να φροντίσουμε τα δεδομένα των ε, πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ασφαλή παντού στον κόσμο. Βέβαια δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο. Είναι πολύ σημαντικό όμως να βρούμε λύσεις ώστε τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών όπως είναι η ιδιωτική σφαίρα να ε, τύχουν προστασίας και στον ψηφιακό κόσμο οι κυβερνήσει πρέπει να προστατεύουν την ασφάλεια των πολιτών του και τη εθνική του ασφάλεια και φυσικά θα πρέπει ταυτόχρονα να καταπολεμούν το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Πώ θα βρούμε την ισορροπία σε αυτέ τι πολιτικέ λύσει με βάση δημοκρατικέ και νομοποιημένε διαδικασίε. Όλε οι κυβερνήσει ζητούν σήμερα πρόσβαση σε δεδομένα. Πρέπει να βρούμε λύσει ώστε να περιοριστούν οι παρεμβάσει στην ιδιωτική σφαίρα, λαμβάνοντα όμω το σφαιρικό χαρακτήρα και τον γενικευμένο χαρακτήρα που έχει το διαδίκτυο. Γι' αυτό και οι λύσει θα πρέπει να είναι παγκόσμιε. Επίση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο σημαντικό αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια παρέμβαση στο ανοιχτό και δωρεάν διαδίκτυο. Η Microsoft ε, καλωσορίζει την ε, πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να βρει λύσει για την κατάσταση αυτή. Και ω πολυεθνική εταιρεία ε, συμμορφωνόμαστε με την νομοθεσία σε πολλέ χώρε είδαμε ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον των κυβερνήσεων για πρόσβαση στα δεδομένα και προσπάθεια να, να προστατευτεί κατά της άρνησης αποκάλυψης τέτοιων δεδομένων. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να αποφύγουμε τον αντίκτυπο αυτής της αυξανόμενης αίτησης και να αποφύγουμε κυρίως την αρνητική επιρροή προς πολίτες και την προστασία της ιδιωτικής του σφαίρας. Χρειαζόμαστε οικουμενικούς κανόνες και αρχές που θα διέπουν την πρόσβαση σε δεδομένα των πελατών μας. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν και να καταλήξουν σε συμφωνίες για τους εφαρμοστέους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να εξασφαλίζουν σεβασμό της ιδιωτικής σφαίρας στο χρηστών από όλες τις χώρες, όπου και αν βρίσκονται οι χρήστε από όπου και αν κατάγονται, λαμβάνοντα υπόψη τον παγκόσμιο χαρακτήρα των προϊόντων και των υπηρεσιών. Επίση, η συζήτηση θα πρέπει να είναι ανοιχτή, ώστε να μπορεί και το κοινό να καταλαβαίνει την έννοια που έχει και το, το σκοπό που έχει η πρόσβαση τη κυβέρνηση σε προσωπικά δεδομένα. Επίση θα πρέπει να, δίνονται περισσότερε πληροφορίε για τα αιτήματα των υπηρεσιών ασφαλεία και των μυστικών υπηρεσιών. Επίση ενθαρρύνουμε το Αμερικανικό Κογκρέσο να ε, εγκρίνει τον σχετικό νόμο και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος είχατε καλεσμένο ένα μέλος του Κογκρέσου που είπε ότι και εμείς υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία, την νομοθετική πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται. Θέλουμε και αναγνωρίζουμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά και μεταρρυθμίσει στο σύστημα. Η εμπιστοσύνη θα αποκατασταθεί όταν ε, αλλάξουν οι κυβερνήσεις τον τρόπο πρόσβαση στα δεδομένα η κρυπτογράφηση, η κωδικοποίηση είναι μία λύση, αλλά προϋποθέτει και εύστοχα μέτρα πολιτικής και λογικά μέτρα πολιτικής. Επίσης, το θέμα της ε, εδαφικής εφαρμογής είναι σημαντική αρχή του δικαίου. Επίσης, χρειάζονται κάποιες συμφωνίες νομικής αρρωγής, αλλά μερικές χώρες ήδη έχουν βρει τρόπους για να παρακάμψουν αυτές τις συμφωνίες. Γι' αυτό και ζητούμε καλύτερη επεξεργασία των συμφανιστών προκειμένου να εξασφαλιστεί αναβάθμιση της συνεργασίας αντί να εξωθούνται οι χώρες σε παράκαμψη της νομοθεσίας. Επίσης, υποστηρίζουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τον σεβασμό του ιδιωτικού βίου και πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε κατοχήρωση των αρχών αυτών και στις ΗΠΑ. Θέλουμε προστασία της ιδιωτικής σφαίρας και καλό θα ήταν να έχουμε ένα συνεπές ε, οικουμενικό πλαίσιο. Έχουμε ε, επίσης μια αντίστοιχη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του κυβερνοχώρου και μια άλλη διεθνή συμφωνία. Έχουμε δηλαδή ήδη διεθνείς συμφωνίες που μπορούν να αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω συζήτηση. Η Microsoft ε, έχει αναλάβει δέσμευση για το σεβασμό της ιδιωτικής σφαίρας ε, και της ελευθερίας έκφρασης. Γι' αυτό και προσβλέπουμε σε συνέχιση του, διαλόγου προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο. Σας ευχαριστώ. Ξέχασα να πω ότι η κυρία Μπέλτς είναι αντιπρόεδρος ε, για τα νομικά και εταιρικά θέματα στη Microsoft για την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Αφρική. Δεύτερος ομιλητής είναι ο κ. Λούντμπλακ, που είναι διευθυντής ε, απίθυνος για δημόσια πολιτική και σχέση με τις κυβέρνηση της Google. Και μετά έχουμε τον κύριο Ρίτσαρ Τάλλαν, που είναι διευθυντή δημόσια πολιτική για την περιοχή Ευρώπη, Μικρασία, ε, Μέση Ανατολή και Αφρική για το Facebook. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσω εδώ σήμερα. Λέγομαι Λούντλαμ και είμαι υπεύθυνο για την κυβερνητική πολιτική και τις σχέσεις ε, για την Google που έχει την στην ε, Ιρλανδία. Εδώ να σας πω ότι ο γενικός διευθυντής της Google αρνείται ε, με κάθε τρόπο τις κατηγορίες ότι συνεργάστηκε με την Αμερικανική κυβέρνηση. Δεν δώσαμε πρόσβαση στις υπηρεσίες της Google στην Αμερικανική κυβέρνηση, ούτε απευθείας ούτε εμέσως με το λεγόμενο Dropbox. Η Google δεν συμμετείχε σε κανένα πρόγραμμα για την εθνική ασφάλεια που απαιτεί να αποκαλυφθούν στοιχεία στην Αμερικανική κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλη και να, δίνοντας πρόσβαση στα συστήματά της, καθώς και τα δίκτυα στα οποία ε, ενεργοποιείται. Ε, μάλιστα ε, προκαλεί ε, όντω όργη το πώς μπόρεσε η κυβέρνηση από οπτικέ ίνες να αντλήσει τα στοιχεία τα οποία άντλησε. Ε, αυτό έχει σοκάρει ολόκληρη την κοινωνία του ίντερνετ και των πληροφοριών και απαιτείται μεταρρύθμιση του συστήματος εποπτείας της συγκέντρωσης προσωπικών δεδομένων. Το να υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασία για μα είναι προτεραιότητα. Η Google θέλει να υπερβεί τα σημερινά όρια προστασία ε, και το κάνει αυτό ήδη με ε, πολλού τρόπους. Όταν υπάρχει κάποια υποψία για την χρήση ενός λογαριασμού μέσω του login, αμέσως ειδοποιεί το χρήστη μέσω email. Επίσης, η Google έχει μια επαλήθευση του κατόχου λογαριασμού σε δύο στάδια, προκειμένου να υπάρχει ένας ενιαίος κωδικός για την χρήση μιας, ενός λογαριασμού πέραν του login και του username. Ένα παράδειγμα από πολλές προσπάθειες που κάνουμε για την ασφάλεια ε, είναι αυτό. Επίσης, για την ε, κρυπτογράφηση των στοιχείων των ε, χρηστών, η Google έχει συγκεκριμένε μεθόδους που είναι ένα σύστημα υπεράσπισης από κάθε είδους κυβερνοεπίθεση, είτε κυβερνητική είτε όχι. Επίσης, η σύνδεση στο Gmail γίνεται με το σύστημα 10 10 και έχει ξεκινήσει να λειτουργεί το σύστημα αυτό από το 2004. Επίση, η αναζήτηση στο διαδίκτυο το 2011 είναι και αυτή κρυπτογραφημένη και ο Eric Roth, ε, ε, υπεύθυνο για τα θέματα ασφαλεία τη Google, ζήτησε στην Washington Post πρόσφατα ότι κρυπτογραφημένη είναι και η μετακίνηση δεδομένων μεταξύ των κέντρων τη Google. Ήδη κάτι ε, που είχε ανακοινωθεί από τον Ιανουάριο του 2011. Ωστόσο, το να δίνεται να προβλέπετε διεξοδική κρυπτογράφηση δεν αρκεί αυτό. Το διαδίκτυο είναι ένα μέρος όπου υπάρχει διαρκής αγώνας δρόμου. Οι επιθέσεις είναι όλο και περισσότερο εξελιγμένες. Έτσι η Google ερευνά και κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι μπροστά από όσους προσπαθούν να επιτεθούν ε, στην προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών της. Κάνει λοιπόν σοβαρές προσπάθειες για να αποφύγει την ε, επίθεση από ιούς. Το 2006 ένα προηγμένο σύστημα που ονομάζεται Safe Bouncing ε, προβλέφθηκε για να αποφεύγονται είδους επιθέσεις στο διαδίκτυο όταν κανείς χρησιμοποιεί Google. Πολλοί πρόβλεψαν το σύστημα μαζί με την Google για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και επίση προειδοποιούνται οι χρήστε όταν πρόκειται να επισκεφθούν έναν ιστότοπο που μπορεί να μην είναι ασφαλή. Το ίδιο λοιπόν και για τι προσπάθειε κυβερνήσεων που προσπαθούν να συλλέξουν πληροφορίε ή να παρακολουθήσουν την συμπεριφορά χρηστών. 10.000 οι καθημερινώ ε, εντυπίζονται από την Google και ένα δι ε, ε, χρηστών προειδοποιείται για την ύπαρξη των ιών. Η Google προσφέρει πόρου για του webmaster που θέλουν επίση να αφήσουν τους ιστοτόπους τους ελεύθερους από ιούς. Ακόμη και η ε, ομάδα εργασίας για τα ζητήματα των ιών ή των ε, ε, παραβιάσεων είναι κάτι που εξασφαλίζει τους δείκτες παγκοσμίω. Επίσης σε λίγα λεπτά θα θέλω να εξηγήσω πως η Google ασχολείται με τα αιτήματα οποιασδήποτε κυβέρνησης για να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα της. Η νομική ομάδα της Google αναζητά εξετάζει την κάθε περίπτωση, ανά περίπτωση ακριβώ, και ε, με τρόπο ανεξάρτητο, διαφανή και ανοιχτό. Εάν τα αιτήματα είναι μεγάλου εύρου, δεν τα δέχεται η ομάδα και βεβαίω τα εξετάζει εξονυχιστικά. Από του οργανισμού για την Εθνική Ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, λόγου χάρη, να σα πω τι έχουμε κάνει ω τώρα. Ε, ε Προσφύγαμε στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ για, ζητώντας μια δήλωση που να προστατεύει τα δικαιώματα των χρηστών. Η δήλωση αυτή δεν μα δόθηκε, Τουλάχιστον θέλησαμε να οργανώσουμε μια διερθωμένη συζήτηση για να γνωρίζουν και οι χρήστε που μπορούν να προστατευτούν από παράνομε δράσει των κυβερνήσεων για ανάγκε των διεκτικών αρχών ή των μυστικών υπηρεσιών για παράνομου σκοπού. Και ήθελα να συζητήσω λίγο το θέμα τη διαφάνεια για να κλείσω, λέγοντα ότι το νομικό πλαίσιο που αυτή τη στιγμή υπάρχει για τι κυβερνητικέ αιτήσει ε, για τα δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών είναι κάτι που μα ενδιαφέρει και ε, ε, ναι, συνηγορούσαμε υπέρ τη διαφάνεια ε, στη χρήση των ε, την εξέταση μάλλον των ετοιμάτων των κυβερνήσεων για τη χρήση των δεδομένων ε, των χρηστών της Google. Η υποβολή εκθέσεων αναχώρα δείχνει τι ε, αιτήματα των κυβερνήσεων υπήρχαν και η Google είναι η πρώτη εταιρεία που χρησιμοποίησε ένα τέτοιο εργαλείο από το 2010. Ε, Επίση, μετά τι αποκαλύψει αυτού του καλοκαιριού, η Google ζήτησε να δημοσιευθούν στατιστικά στοιχεία για αιτήματα ή αιτήσει που έγιναν βάσει των θεμάτων εθνικής ε, ασφαλείας ή εθνικού δικαίου. Η διαφάνεια στη δικασία είναι απαραίτητη. Κανεί δεν μπορεί να δει για την ώρα τι έχει ζητήσει μια κυβέρνηση ή τελικά τι προσήλθε στο δικαστήριο. Η διαφάνεια όμω είναι μόνο το πρώτο βήμα. Οι συμφωνίε όπω ε, οι συνθήκε για την αμοιβαία αρρωγή ή ότι καλύπτονται τα νομικά πρότυπα ή ένα συγκεκριμένο και συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο για οποιαδήποτε νομική έρευνα και στοιχεία που συλλέγονται από το διαδίκτυο είναι κάτι που αφορά όλε τι χώρε, όχι μόνο αυτέ στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα τη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για την συνεργασία των διοικητικών αρχών. Αλλά περισσότερα μπορεί να γίνουν για να βελτιωθεί η όλη διαδικασία όπω σήμερα προβλέπετε. Έχουμε σκεφτεί τι μεταρρύθμιση θα χρειαζόταν εδώ και χρόνια και ευχαρίστω να συζητήσουμε με την Επιτροπή σα για τέτοια ζητήματα. Σα ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σα. Ε, και στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε τόσο συνεπτικός ο τελευταίος ομιλητή θα είναι ο κύριος Άλλαν, ε, που εκπροσωπεί το Facebook. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να είμαι και εγώ συνοπτικό όπως ο Νίκολας και για να ε, διευκολύνω τις διερμηνίες θα αφήσω το πρώτο τρισέλιδο της παρουσίασής μου και θα ξεκινήσω στο τέρμα της σελίδα 3 για την ε, αίτηση και τις αιτήσει υποβολής δεδομένων για να σας δείξω πόσο είμαστε αποτελεσματικοί. Ποιες είναι οι πολιτικές του Facebook για την αποκάλυψη στοιχείων του Facebook ε, και εδώ θα γίνω λίγο ε, ε έχει καθορισμένες διαδικασίες για να βοηθά τις ε, αρχέ αρχές ανά τον κόσμο ή τις κυβερνητικές αρχές που ζητούν ε, δεδομένα. Αυτές οι κατευθυντήρες γραμμές είναι δημοσιευμένες στον ιστοτοπό μας και οι αρχές της Ευρώπης ή από τον υπόλοιπο κόσμο μπορούν να απευθύνουν αιτήματα για την αποκάλυψη των δεδομένων απευθείας στο Facebook μέσω του, μέσω του συστήματος που προβλέπεται και στη σελίδα www.facebook.com records το σύστημα των επιγραμμικών αιτήσεων ακόμη μέσω Facebook ή ταχυδρομικά προς την Facebook Island. Για να είναι κατανοητές αυτές οι πρακτικές, ε, το Facebook ε, δίνει, προσφέρει κατάρτιση και ε, εκπαίδευση για αστυνομικού σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να γνωρίζουν τι ισχύει για το διαδίκτυο και την ασφάλεια των παιδιών. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα των κυβερνήσεων και το Facebook τα εξετάζει πολύ ε, αυστηρά, προκειμένου να υπάρχει υψηλή νομική προστασία. Η κάθε αίτηση εξετάζεται ξενοχιστικά, προκειμένου να δούμε κατά πόσο ανταποκρίνεται στο νομικό πλαίσιο, σε αυστηρά πρότυπα και με λεπτομερή περιγραφή των αναγκών που υπάρχουν για να υποβληθεί το αίτημα αυτό. Έτσι, όταν υπάρχουν ανεπάρκειες ή πλημελήματα το Facebook δεν δέχεται τις επίσης και έχει περιορίσει πάρα πολύ την κατηγορία αιτημάτων που μπορεί να αποδεχτεί. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα μπορεί να δοθούν πολύ περιορισμένα στοιχεία για ένα λογαριασμό, όπως τα βασικά στοιχεία του μέλους. Επίσης, ε, εφόσον υπάρχει επικείμενος κίνδυνος θανάτου ή σωματικής βλάβης, το Facebook μπορεί να απαντήσει πολύ άμεσα σε αιτήματα, σε περιπτώσεις απαγωγής λόγου χάρη, προκειμένου να εντοπιστεί ένα παιδί που έχει απαχθεί. Ε, υπάρχει υπεύθυνο ε, για την προστασία των δεδομένων στα κεντρικά της Ιρλανδίας και ο οποίος υποβάλλει εκθέσεις ε, συστηματικά. Σύμφωνα με την έκθεση του Σεπτεμβρίου 2012, ο υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων είδε ότι ε, καλύπτονται όλα τα πρότυπα για την προστασία των δεδομένων μέσω από την πολιτική του Facebook, το οποίο αποτιμά ορθώς τις, τα αιτήματα για την αποκάλυψη πληροφοριών και όταν απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες πληροφορίε ή δεν υπάρχει επαρκή αιτιολόγηση, οι αιτήσει απορρίπτονται. Βέβαια, του τελευταίου μήνε υπήρξε πολύ μεγάλη προβολή στα μέσα μαζική ενημέρωση και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα κυβερνητικά αιτήματα προ του επιγραμμικού ε, προμηθευτέ ε, υπηρεσιών για το κατά πόσον ε, υποβλήθηκαν αιτήματα για αποκάλυψη στοιχείων. Πολλέ φορέ όμω ο τρόπο που αυτά αποβλήθηκαν στα μέσα μαζική ενημέρωση ήταν ανακριβή και παραπλανητικό. Το Facebook λοιπόν έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα. Ο Μάρκ Τζοκεμπέρκ που είναι ο ιδρυτή του Facebook και ο ε, γενικό ε, διευθυντή είπε ότι δεν μπορεί να υπάρχει άμεση ή ανεμπόδιστη πρόσβαση από οποιαδήποτε κυβέρνηση στα δεδομένα του Facebook. Διότι το Facebook δεν είναι ούτε υπήρξε ποτέ μέρος προγράμματος για να παράσχει στην Αμερικανική οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση άμεση πρόσβαση στη, στα στοιχεία των μελών. Ουδέποτε υπήρξε κάποια ε, γενική αίτηση ή δικαστική εντολή για να αποκαλυφθούν σε κυβερνητικό φορέα στοιχεία ή μεταδεδομένα. Ε, ε, χοντρικά ε, σε μεγάλο όγκο. Ε, Ιδάλλω θα είχαμε αντισταθεί. Έπειτα το Facebook έχει αποκαλύψει τον όγκο των πληροφοριών που οι κυβερνητικές, που οι κυβερνητικοί φορείς έχουν δεχτεί. Υπάρχει συγκεκριμένη, υπάρχουν συγκεκριμένε διαπραγματεύσει με την Αμερικανική κυβέρνηση και βεβαίω ε, καμία άλλη εταιρεία δεν έχει κάνει κάτι ανάλογο στο παρελθόν, ενημερώνοντα για τα αιτήματα τη Αμερικανική κυβέρνηση για σκοπού εθνική ασφαλεία ω τώρα. Α, για του ε, έξι μήνε που τελειώνουν την 31η Δεκεμβρίου 2012, ε, οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, οποιοδήποτε φορέας που έχει υποβάλει αιτήματα ε, για στοιχεία από το Facebook ήταν γύρω στις 9 με 10 Τα αιτήματα αυτά είχαν να κάνουν από την περίπτωση ενός τοπικού σερίφη που αναζητούσε ένα παιδί που είχε εξαφανιστεί μέχρι την διερεύνηση μιας μιας κλοπής ή κάποιον που, ε, ομοσπονδιακό αστυνομικό που έψαχνε στοιχεία για μια τρομοκρατική απειλή μελετήθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο 18-19.000 λογαριασμοί χρηστών. Τον Αύγουστο αποκαλύψαμε στοιχεία ε, στην Αμερικανική κυβέρνηση με την συνολική έκθεση για τις κυβερνητικές αιτήσει. Εκεί καταγράφηκαν τα στοιχεία που δόθηκαν σε οποιαδήποτε κυβέρνηση ανά τον κόσμο μέχρι το πρώτο εξάμεινο του 2013. Η έκθεση αυτή καταγράφει όλες τις αμερικανικές αιτήσει, 11 με 12 που ζητούσαν πληροφορίες για περίπου 20 έως 21.000 λογαριασμούς. Να σημειώσουμε ότι ο αμερικανικός αυτό αριθμός περιλαμβάνει όλες τις αιτήσει που έγιναν και εκ μέρους τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, μέσω τη συνθήκη ε, για την αμοιβή νομική αρρωγή. Ε, μέσω λοιπόν αυτή τη διαδικασία τη νομική αρρωγή, αίτηση υποβλήθηκε στο Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνη από ομόλογο Υπουργείο Συνεργαζόμενη Χώρα και εξετάστηκε ε, από ε, το Αμερικανικό Δικαστήριο σε ένα πρόκειτο για εγχώριο, εσωτερικό αίτημα των ΗΠΑ. Ε, βλέπετε πόσο πλαισιωμένη είναι όλη η διαδικασία. Στη συνέχεια υπήρξε μια συγκεκριμένη έκθεση για κάθε ευρωπαϊκό αίτημα και οι αιτήσει που ήρθαν προ εμά από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα έφτασαν στι 8.500 για την ίδια περίοδο, ενώ αφορούσαν περίπου 10.000 λογαριασμού. Με περισσότερου από 1,2 δισεκατομμύρια χρήστε ενεργού καθημερινά, οι εκθέσει αυτέ δείχνουν ότι είναι ένα απειροελάχιστο κλάσμα των συνόλου των χρηστών του Facebook, αυτό που καλύφθηκε από κυβερνητικά κίνητα την περασμένη χρονιά. Αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί να μας δώσει μια σχετική εικόνα, ε, σχετικοποιημένη εικόνα για το τι αριθμητικά στοιχεία συζητάμε και για το πόσο υπερβολικέ παραπλανητικέ είναι οι δηλώσει που γίνονται στον τύπο για τη δράση του Facebook. Επίση, όπω και άλλοι στον κλάδο, το Facebook πιέζεται την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να γίνει ακόμη διαφανέστερη σε σχέση με τα αιτήματα που υποβάλλει. Το Σεπτέμβριο το Facebook προσέφυγε ε, στο ε, δικαστήριο FISA, Φάιζα τη Washington για ε, την αποκάλυψη, για θέμα αποκάλυψης στοιχείων σε σχέση με θέματα εθνικής ασφαλείας και για το πόσο τέτοια θέματα μπορεί να χειρίζεται. Ε, οι λογαριασμοί και ο συνολικός αριθμός ε, έπρεπε να γίνουν αντικείμενο οριοθέτησης, το ίδιο και οι συναλλαγέ ή οι πληροφορίε για τα μέλη. Πιστεύουμε όμω ότι για τη διαφάνεια πρέπει να γίνουν περισσότερα γιατί είναι κρίσιμο το θέμα αυτό. Ε, τον Οκτώβριο μαζί με άλλου προμηθευτέ ε, το Facebook ζήτησε να πλαισιωθούν οι κυβερνητικέ δράσει εποπτεία και παρακολούθηση προκειμένου να υπάρχουν και μηχανισμοί λογοδοσία και εποπτεία για τι περιπτώσει αυτέ. Μαζί με άλλε εταιρείε όπω ε, μα είπε και ο ε, κύριο Σένσεμπρένερ σήμερα Καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να προστατευτούμε καλύτερα και να πλαισιωθούν τα αιτήματα αυτά. Στο Facebook λοιπόν θα συζητούμε, θα συνεχίσουμε να ζητούμε από όλε τι κυβερνήσει να είναι όσο το δυνατόν διαφανέστερε γίνεται στα αιτήματα που υποβάλλουν. Ελπίζουμε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύστημα σε διεθνέ επίπεδο, καθώ πρόσβαση στα δεδομένα του διαδικτύου ζητούνται όλο και περισσότερο. Πιστεύουμε ότι έχουμε ένα ρόλο να διαδραματίσουμε εδώ, ώστε να υπάρχει ένα ε, γενικό κλίμα εμπιστοσύνη στο πώ οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ε, το διαδίκτυο και πώ βεβαίω οι κυβερνήσει μπορούν μπορούν να ασκήσουν τι εξουσίε του και από τον ευαίσθητο χώρο. Ελπίζουμε το Ευρωκοινοβούλιο να μα δώσει την ειδική του γνώση ώστε να λύσουμε τέτοια περίπλοκα ζητήματα και με στη διάθεσή σα για να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτημα έχετε και να σα διευκολύνω στην όλη διαδικασία. Um, okay, having listened to these three... Ευχαριστώ. Ακούσαμε τι τρει εισαγωγέ και τώρα ε, ανοίγει η συζήτηση, ε, ερωτήσει, απαντήσεις, ε, ε, συγητής, δύο σκιώδης και άλλοι δύο, άλλο κανεί, ναι, η κυρία Λάτσφορντς. και τρεις ε, άλλοι και εγώ τελευταία στον κατάλογο. Λοιπόν, προτείνω την εξής διαδικασία. Είτε να απευθύνετε το ερώτημά σας σε ένα συγκεκριμένο ομιλητή μας ή θα ζητήσω και από τους τρεις να απαντήσουν με την ίδια σειρά. Ο κύριος Μωράες. Ευχαριστώ Σοφή. Με τόσες προφορίες που πήραμε Είχαμε και την Apple στην Ουάσιγκτον και τώρα τις τρεις μεγάλες εταιρείες ε, και στις ιστοσελίδες. Ε, αυτό που ακούμε ε, είναι μια απάντηση στις βασικές κατηγορίες και ισχυρισμούς. Να υπενθυμίσουμε και πάλι ποιες ήταν οι βασικές κατηγορίες και ισχυρισμοί αυτοί. Γιατί υπάρχει μια άρνηση αναπόφευκτη προφανώς, αλλά να σας πω ε, ε, και πάλι μερικά πράγματα και να κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Δεν θα πάρουν και πάρα πολύ το λόγο. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να ρωτήσω ειδικά ε, την κυρία Μπέλτς για τη Microsoft και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Τα εξής. Μερικά από τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρατε, για να μην χαθούν για τα πρακτικά. Η Microsoft κάνει κρυπτογράφηση στα, ε, μεταξύ των ε, κέντρων δεδομένων. Γιατί η Google είπε ότι δεν κάνει. Η Microsoft προβαίνει σε τέτοια κρυπτογράφηση. Αν όχι, προτίθεται να το κάνει. Ε, ή να το απαγορεύσει σε αντίθεση με την Google. Επίσης, στη δήλωσή σας Ε, πολύ γρήγορα ε, αντιπαρήλθατε το γεγονός της νομοθεσίας και είπατε ότι συμφωνείτε με τον κύριο Σένσενμπρένερ. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω γιατί μέχρι τώρα από ό,τι ακούμε το 90% της παραγωγής ε, του Prism βασίζεται στη Yahoo, στη Google και στη Microsoft. Δηλαδή στο email, στο Skype, στο Hotmail έχετε αφήσει την πρόσβαση. Πώς υπάρχει δυνατότητα αυτών των υποκλοπών ε, και των ε, επικοινωνιών. Πώς αντιδράτε εσείς αυτές τις αιτιάσεις. Γιατί έτσι λίγο νομίζω ε, τις αντιπαρήλθατε πάρα πολύ εύκολα. Πώς αντιδράτε σε αυτές τις κατηγορίες. Ότι χρησιμοποιούνται διαδικασίες δώσατε πρόσβαση στην NSA με, τρόπο και διαδικασίες πουλ και πους. Εσείς μιλήσατε για εντάλματα και κλητεύσεις, αλλά δεν σας κατηγορούν γι' αυτό. Σας κατηγορούν ότι μαζικά δίνετε ε, hidden στοιχεία, αυτό, bulk data. Ε, πώς απαντάτε σε αυτό. Ε, για τον κύριο Λούντμπλαντ. Ε, μιλήσατε για την εμπιστοσύνη των χρηστών, για τις μεταρρυθμίσεις, αλλά στις 30 Οκτωβρίου και πάλι στην Ουάσιγκτον ρωτήσαμε τι γίνεται με την πρόσβαση ε, από σερβερ σε σερβερ και τις κατηγορίες που σας απευθύνουν. Δεν θέλω να τις επαναλάβω, αλλά έτσι, για να ακούσουμε την άποψή σας για να γραφεί και στα πρακτικά. Πώς απαντάτε σε όλα αυτά. Τα είπατε στην παρέμβασή σας ε, και πάλι για το Facebook. Μίλησατε για το Mark Zuckerberg και ε, την άρνηση. Είχε όμως πρόσβαση, ε, είχε την άδεια συνεργασίας με υπηρεσίες της Αμερικανικής κυβέρνησης. Το το διαψεύδεται δεν σημαίνει ότι δεν συνέβη κιόλα. Και μέχρι τώρα από τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψουμε ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο με την NSA. Ευχαριστώ. Θα ζητήσω από τους ομιλητές μας να απαντήσουν. Παρακαλώ δύο λεπτά έκαστο στο πολύ, αλλιώς δεν θα προλάβουμε μέχρι τις 6.30. Η κυρία Μπέλτς. Θα προσπαθήσω. Καταρχάς, με το πρίσμα και τη δυνατότητα παρακολούθησης. Το μόνο που μπορώ να επιβεβαιώσω είναι αυτό που επιβεβαιώνει και η αρχή της Microsoft, η διεύθυνση, η διοίκηση. Δεν ξέρουμε τι είναι το πρίσμα, δεν έχουμε χρησιμοποιήσει, δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα, ούτε δίνουμε πρόσβαση χωρίς έλεγχο. Κοίταξε όλο το οικοσύστημα, υπάρχει ε, τρόπος να φτάσει κανείς του σερβερ και της Microsoft και στα δεδομένα και έχουμε κοινό συμφέρον να μάθουμε πώς έγινε αυτό. Το δεύτερο, απαντώ και στην τρίτη ερώτηση, η άμεση πρόσβαση, την ανέφερα και στην εισαγωγική μου ε, παρουσίαση, δεν δίνουμε άμεση πρόσβαση ε, στους σερβερ. δεν έχουμε το σύστημα push, έχουμε το pull. Το μόνο που μπορώ να σας πω για την ε, κρυπτογράφηση. Η Microsoft προσφέρει πολλές υπηρεσίες, ένα φάσμα δεν μπορώ να σας εξηγήσω τι κάνουμε παντού με τα διάφορα συστήματα και τις υπηρεσίες, ούτε πώς τις κρυπτογραφούμε. Γενικά, αυτό που θα μπορούσα να σας πω σήμερα είναι ότι η μεταφορά των δεδομένων από σερβερ σε σερβα δεν είναι κρυπτογραφημένη. Γι' αυτό ε, αναθεωρούμε το σύστημα ασφαλείας για να μην υπάρχει δυνατότητα υποκλοπών από την εσωτερική μας ενημέρωση. Ευχαριστώ κύριε Νούμπλα. Thank you. Ευχαριστώ. Σε τη φορά της καταγγελίας στη Washington Post, εμείς όπως όλα τα συστήματα στην κοινωνία των πληροφοριών ε, είμαστε ε, συνεχώς ε, ε, σε, ελέγχουμε τα συστήματά μας και τον τρόπο αντίδρασης. Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε την κρυπτογράφηση όλων των συνδέσεων και όλων των δικτύων για προστασία. Βέβαια είναι μια διαδικασία να εξελίξει, δεν μπορούμε ποτέ να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια και αναζητούμε συνεχώς μέσα και μεθόδους για να εξασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια των δικτύων μας. Ο κύριος Άλαν, σε ό,τι αφορά το υλικό που δημοσιεύθηκε, και εμείς μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα αυτά και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, ούτε το γεγονός ότι... Ε, δουλεύει κανείς σε μια επιχείρηση τη δικιά μας σημαίνει ότι γνωρίζει περισσότερα για, τη, για τα κυβερνητικά γρανάζια. Εδώ μιλούμε για το εσωτερικό σύστημα και την μεθοδολογία του NSA. Αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε εμείς είναι όταν υποβάλλεται από ένα τέτοιο φορέα ένα αίτημα για πρόσβαση σε δεδομένα. Αυτά τα σας, σας τα διευκρινίσαμε. Είπαμε ότι μπορούμε να δημοσιεύσουμε όσο περισσότερες πληροφορίες μπορούμε για τις αιτήσει αυτές και είπαμε ότι οι αιτήσει είναι στοχοθετημένες, στοχευμένες, ε, ε, δεν ε, ζητούν μαζική ε, πρόσβαση, ούτε άμεση πρόσβαση σε δεδομένα και επίσης στηρίζονται σε μια νόμιμη νομότυπη διαδικασία. Δεν συμβαίνει τίποτε άλλο ύποπτο. Γιατί μετά από τα στοιχεία που κυκλοφόρησαν προσπαθούμε και εμείς ως εταιρεία να είμαστε όσο πιο σαφείς γίνεται. Αυτές είναι οι μόνες αιτήσει που λάβαμε και δεν υπάρχει τίποτα που να λαμβάνει χώρα κρυπτό. Ο κύριος Όλμπρεχτ. Άλμπρεχτ, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ που ήρθατε. Έχω ερωτήσει και παρακαλώ να τις απαντήσετε και όχι απλώς να τις σημειώσετε. Χαίρομαι ιδιαίτερος για την παρουσία σας εδώ και χαίρομαι ιδιαίτερα για τα σχόλια της κυρίας Μπέλτς για την ανάγκη νομοθεσίας για την προάσπιση της ε, ιδιωτικής σφαίρας. Και επίσης χαίρομαι που και οι εταιρείε ε, τεχνολογίας των πληροφοριών ε, συμφωνούν με την ανάγκη μιας τέτοιας νομοθεσίας, όπως και οι νομοθετικοί φορείς της Ηνωμένε Πολιτείε. Θα πρέπει να φροντίσουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε κοινού κανόνες. Άκουσα λοιπόν όλα σας τα σχόλια και τις παρατηρήσεις και Άκουσα ιδιαίτερα από τις κυρίες Λούντμπλαντ και Άλεν το πρόσβαση που να μην καλύπτεται από μια νομότυπη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να υπάρχει άλλος τρόπος πρόσβαση, πρόσβαση στα δεδομένα σας και θα μπορούσε να έχει συμβεί και τέτοιος άλλος τρόπος. Γιατί Απλώς ε, είπατε ότι δεν υπάρχει ε, αδικαιολόγητη πρόσβαση ή μη νομότυπη πρόσβαση. Το θέμα είναι όταν ε, μιλάτε για unwarranted access, σε τι δικαιοδοσία αναφέρεστε, τι νόμους ακολουθείτε όταν εσείς επεξεργάζεστε προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών. Μπορείτε να αρνηθείτε πλήρως ότι παραβιάζετε ενωσιακή νομοθεσία όταν επεξεργάζετε προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης, ε, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι κάποιες αρχές ε, επιτίθεται στο σύστημά σας. Ζητάτε από αρχές ε, στα κράτη-μέλη να διερευνήσουν πιθανότητες παραβιάσεις του του συστήματος ε, της ασφάλειας των διακομιστών σας, ε, η παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Κάνετε δικές σας έρευνες για τέτοιες πιθανές ε, επιθέσεις στην ασφάλεια των δικτύων σας. Είναι ερωτήσεις που πραγματικά και είναι τους πολίτες και γι' αυτό περιμένουμε υπομονησία της απαντήσεις σας, ιδιαίτερα στην πρώτη ερώτηση για το θέμα της δικαιοδοσίας. Επίσης, τι γίνεται με τα clouds, ε, πώς κρίνεται εκεί η αρμόδια δικαιοδοσία. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Ποιος θέλει το λόγο, κυρία Μπέλτς, ο κύριος Ο κύριος Άλμπερχτ μίλησε για την εφαρμοστέα δικαιοδοσία. Ε, και σίγουρα θα πρέπει να αποκλείσουμε σύγκρουση συμφερόντων γιατί στο νέο κόσμο δεν υπάρχει τίποτα σαφές. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε να συμμορφωθούμε με όλες τις νομοθετικές διατάξεις. Και όταν ε, είναι συμβατές οι νομοθετικές διατάξεις, ωραία, αλλά μερικές φορές είναι και αντιφατικές μεταξύ τους. Και τότε είναι δύσκολη η συμμόρφωση. Τώρα, είπατε πώς εφαρμόζουμε τους κανόνες όταν ε, ε, διακομιστής είναι στις ΗΠΑ. ακολουθούμε το Αμερικανικό Δίκαιο και αν τα δεδομένα βρίσκονται στην Ιρλανδία, τηρούμε το Ιρλανδικό δίκαιο. Μέχρι στιγμής ήμασταν τυχεροί και δεν είχαμε πρόβλημα να εφαρμόσουμε τους ε, εθνικούς κανόνες. Σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία και το περίφημο άρθρο 43 για τη νομοθεσία ιδιωτική ε, σφαίρα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί θα δημιουργούσε μια σύγκρουση συμφερόντων και όχι μόνο δεν θα επιλύσει το πρόβλημα ε, ο κορώνας αυτός, αλλά θα μας οδηγήσει και σε μια σύγκρουση που σίγουρα θα ήταν επιθυμητή. Τώρα, όταν γίνεται επίθεση σε ένα διακομιστή μας, σε ένα σερβερ, οποιαδήποτε τέτοια επίθεση βάλει κατά του συστήματος προστασίας μας. Εμείς ε, έχουμε πολύ ε, εκλεπτισμένους και εξεζητημένους μηχανισμούς ε, απόκρουσης τέτοιων κυβερνοεπιθέσεων. Γιατί πολλοί θέλουν να έχουν πρόσβαση στους διακοσμιστές μας. Εμείς ελέγχουμε συνέχεια τα συστήματα ασφαλείας μας και φυσικά συνεργαζόμαστε και με κυβερνητικούς φορείς για να καταπολεμήσουμε το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Σας ευχαριστώ κύριε Σλούντμπλατ. Ευχαριστώ σε ό,τι φορά την δικαιοδοσία πολύ σωστά μίλησε για σύγκρουση εφαρμοστέου δικαίου πολλές φορές ε, η Ντόρθη. Μερικές φορές τα ζητήματα είναι ε, διακυβερνητικά, θα πρέπει να επιληθούν σε επίπεδο κυβερνήσεων. Μερικέ περιπτώσει είναι καθαρή περίπτωση. Ο διακομιστή βρίσκεται στι ΗΠΑ, εφαρμοστέο είναι το Αμερικανικό δίκαιο, αλλά δεν είναι πάντα τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε και εμεί αφήνεια για το εφαρμοστέο δίκαιο και το αρμόδιο το την κατάλληλη δικαιοδοσία. Μιλήσατε για το cloud, την εφοϋπολογιστική. Θα πρέπει να συναυθούν συμφωνίες μεταξύ των κυβερνήσεων. Από αυτές θα κριθεί και το εφαρμοστέο σύστημα. Και εμείς έχουμε διάφορες ομάδες που ελέγχουν το σύστημα για να αποτραπούν επιθέσεις. Θέλουμε να ενισχύσουμε το σύστημα και να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε οποιασδήποτε κυβέρνο επιθέσεις. Εμείς προσπαθούμε να προστατεύσουμε και τους χρήστες μας, αναζητώντας συνέχεια pattern επιθέσεων για να προστατευτούμε. Δυστυχώς συνέχεια γίνονται προσπάθειες ε, εισόδου, διείσδησης στο σύστημα. Προσπαθούμε να τις αποκρούσουμε. Ο κύριος Σάλλαν, ευχαριστώ ε, ε, να συμπληρώσω κάτι για το θέμα αυτό της δικαιοδοσίας. Έχουμε πολλαπλές ευθύνες προφανώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου είναι η υποδομή μας αλλά και στην Ιρλανδία γιατί το Facebook ε, ελέγχεται για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά από την Ιρλανδία και επίσης έχουμε κάθε φορά ευθύνη στην Ελλάδα χώρα που ε, εκδίδει το αίτημα για διαβίβαση δεδομένων και ε, πολλές φορές καταναλώνουμε πολύ χρόνο για να ζογκλάρουμε με όλες αυτές τις ευθύνες και νομοθεσίες για να μην παραβιάσουμε κανέναν στον νόμο. Ε, αυτό που σας ενδιαφέρει εσάς που είστε νομοθέτες είναι να μην αφήσουμε τις ακραίες περιπτώσεις να επηρεάσουν πάρα πολύ τη συνήθη λειτουργία. Ξέρουμε ότι γίνεται μια ακραία συζήτηση για μαζική ε, μεταφορά στοιχείων το αίτημα, το κλασικό που έχουμε είναι για το κλασικό ποινικό δίκαιο. Προσπαθούν να πιάσουν κάποιον στη Γερμανία που έκανε κάτι κακό στη Γαλλία ή στην Ολλανδία ή στη Σουηδία. Ε, έναν εγκληματία. Αυτά ε, μας ζητούν κυρίως οι διεκτικές αρχές και θέλουν τα συστήματα να λειτουργούν απρόσκοπτα έτσι και χωρίς μεγάλες τριβές. Ε, πρόκειται για συνήθεις περιπτώσεις κανονικές του ποινικού δικαίου για τη δικαστική συνδρομή για να μπορούν με τις απαραίτητες εγγυήσεις να λειτουργούν έτσι οι διοκτικές αρχές. Ευχαριστώ. Um, um, Ευχαριστώ πολύ και θα μιλήσω και εξ ονόματος των φιλελευθέρων εγώ. Ποιο άλλος θέλει, θέλεις να επανέλθει ο κύριο Άλμπρεχτ. Ένα μικρό κάτι, γιατί δεν απαντήσατε. Αν ε, κάποια ε, κρατική διοκτική αρχή σα ζητήσει κάτι. Το κάναμε αυτό, ναι. Ε, έχω ε, συμμετάσχε μια περίπτωση hacker που πραγματικά βρήκαμε κάποιον από το Ηνωμένο Βασίλειο που προσπαθούσε να μπει στο σύστημά μας και το διαβιβάσαμε στις ιδιοκτικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και τους βοηθήσαμε να τον πιάσουν. Έτσι λειτουργούμε. Ευχαριστώ. Ε, μιλώ και εγώ λοιπόν ε, ως και όδηση ε, των φιλελευθέρων πριν δώσω το λόγο στα λοιπά μέλη της Επιτροπής. Χαίρομαι πολύ που ήρθατε, αλλά αυτά είναι νομικές δηλώσεις που τις έχετε σχολαστικά προετοιμάσει. Ε, το έχω ξανακάνει αυτό το ανέκδοτο, το έχω ξαναπεί. Ο πρόεδρος Κλίντον όταν είπε στην υπόθεση Λουίσκη ότι δεν είχα ε, σεξουαλικές σχέσεις με αυτή τη γυναίκα. Ε, σχέσεις, σχέσεις, όχι, όχι σεξ. Όχι, όχι στην ουσία, τι είναι αυτά που λες λέει ο Μωράης, όχι σεξουαλικές σχέσεις, ναι, άρα δεν κάνω για δικηγόρος, ε, που ήταν στην κυριολεξία σωστό, αλλά δεν ήταν η αλήθεια. Και ε, πρόκειται για Ευρωπαίους πολίτες εδώ. Ακόμα και αν θέλατε να πείτε την αλήθεια, δεν το λέω προσωπικά αλλά για τις εταιρείε που εκπροσωπείτε. Με συγκινεί, πώς να το πω, ο διακαής σας πόθος ε, να συμμορφώνεστε και να είστε ε, έμπλεοι διαφάνειας. Αλλά είναι πολύ αργά. Για πάρα πολλά χρόνια και ε, ε, off άκουγα πάρα πολλά πράγματα, κανείς δεν τα έλεγε ποτέ δημόσια. Δεν είναι σαν να Ακούω εταιρείε ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται για επιχειρήσει, εταιρείε που συνεργάζονται με κυβερνήσει. Υποπίεση μάλιστα, το αναγνωρίζω. Υποπίεση βεβαίω. Παρ' όλα αυτά συμβαίνει. Εντάξει, ε, οι δικαιοδοσίε συγκρούνται, καμιά φορά είναι δύσκολη να υπάρξει διευθέτηση κτλ. Καταλαβαίνω. Ποιο το είπε, ο Διευθύνων Σύμβουλο τη Γιαχού, που είπε ότι αν πω αυτά που θέλω να πω, μπορεί να καταλήξω φυλακή για καμιά 35 χρόνια. Μα ε, όταν τη, συμμορφώνεσαι με τον Αμερικανικό νόμο παραβιάζεις Ευρωπαϊκό νόμο. Και αν εγώ ήμουν εταιρεία και με πίεζε Αμερικανική κυβέρνηση, καταλαβαίνω τι θα έκανα. Αλλά τελικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι πολίτες και οι χρήστες σας και αναφερθήκατε στην εμπιστοσύνη. Εσείς πια ε, μπορείτε να κατηγορείτε τους πολίτες, τους χρήστες ότι δεν εμπιστεύονται πια τις εταιρείες σας. Μερικές ερωτήσεις για την κρυπτογράφηση. Ωραία, θαυμάσια, σπουδαία. Σε μια προηγούμενη συνεδρίαση ακούσαμε ότι ακόμα και εταιρείε που πιστοποιούν τα πρότυπα κρυπτογράφησης μπορεί να έχουν ε, δωροδοκηθεί, α πούμε, ή ε, πιεστεί από την Αμερικανική κυβέρνηση. Μου λέτε ότι τα δεδομένα μου είναι κρυπτογραφημένα. Ωραία, και αυτό τι σημαίνει. Λέτε ότι δεν υπάρχουν παραθυράκια, ούτε το αυτό το ξέρω. Από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ε, είναι γεμάτη παραθυράκια που τα δημιουργούν, τα φτιάχνουν και μπορεί να μην σας αφήνουν και να μας το πείτε. Πού να τα ξέρω όλα αυτά και ποια εμπιστοσύνη. Άλλο στοιχείο. Ακούμε ιστορίες στα μέσα ενημέρωσης για πληρωμές όχι απλώς ε, να καλύπτεται το, το ε, κόστος της συμμόρφωσης, αλλά για πληρωμή. Μπορείτε να πείτε δημόσια ότι δεν πήρατε λεφτά, δεκάρα τσακιστή πέρα από το κόστος ε, της συμμόρφωσης. Και δηλαδή είστε πρόθυμοι να δώσετε στην Επιτροπή μας μια επισκόπηση των εντολών που έχετε λάβει από τις κυβερνήσεις πέρα από τις άμεσες πληρωμές. Βέβαια υπάρχει και όρος που λέει δεν δαγκώνει το χέρι που σε ταΐζει. Υπάρχει τουλάχιστον μία εταιρεία εδώ πάνω σε αυτό το πάνελ που έχει τεράστιες ε, ε, παραγγελίες από τον αμυντικό τομέα. Εντάξει, καλή διαφάνεια και τα συμφέροντα των εταιρεών Επίσης, ε, τι φρονείτε για τον ασφαλή λιμένα. Τι είναι αυτό το safe harbor. Δίνει ε, οποιαδήποτε ασφάλεια στους χρήστες σας. Αυτές τις ερωτήσεις είχα να κάνω και θα παρακαλούσα τα μέλη του πάνελ να απαντήσουν με τη γνωστή σειρά. Η κυρία Μπέλτς. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Καταλαβαίνω τη σύγχυσή σας. Καταλαβαίνω Καταλαβαίνετε όμω και εσύ ότι δεν μπορείτε να περιμένετε τι δηλώσει από τι εταιρείε να κάνουν δηλώσει ότι παραβιάζουν τον νόμο και να πάνε γενικέ διευθυντέ φυλακή. Κοιτάξτε, κάποιε φορέ μπορείτε να εξαναγκάζεστε να σιωπάτε, αλλά εδώ βρισκόμαστε στην Ευρώπη και στην Ευρώπη υποτίθεται ότι υπάρχει υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για τέτοιου παραβιάσει. παραβιάσεις. Μπορεί λοιπόν στην Αμερική να γεννηθεί κάτι τέτοιο, αλλά... Κοιτάξτε, αν με αφήνατε να ολοκληρώσω για ένα θέμα, θα μπορούσατε να καταλάβετε. Όπως λέγαμε, είμαστε όλοι υπέρ του να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτό θα επιτρέψει καλύτερη ε, συζήτηση, να γίνεται μια συζήτηση βάσει των δεδομένων. Αλλά στον αμερικανικό, στο αμερικανικό δίκαιο δεν προβλέπεται να τα ε, εκθέτουμε τα θέματα αυτά. Και σε κάποιε ευρωπαϊκέ χώρε το ίδιο. Ακολουθούμε λοιπόν του κανόνε. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να κατηγορείτε εμένα ή κάποιον άλλο που ακολουθούν κανόνε που άλλοι προβλέπουν. Το δεύτερο ερώτημα είναι τι κάνουμε και δεν το λέμε. Και αν αυτά που κάνουμε και δεν λέμε παραβιάζουν του ευρωπαϊκού κανόνε. Αυτό είναι τελείω διαφορετικό ερώτημα. Εγώ δεν έχω παραβιάσει κανένα κανόνα σήμερα. Αυτό μπορώ να σα πω. Καταλαβαίνετε όμω και τη δύσκολη θέση στην οποία βρισκόμαστε, γιατί υπάρχουν ε, κατηγορίε και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτές τις κατηγορίες να τις αντικρούσουμε. Αλλά σας ζητώ, μην καταλήγετε σε γρήγορα συμπεράσματα για το τι πραγματικά συμβαίνει ή όχι. Αυτό δεν έχει να κάνει με παρασκήνια ή το τι συμβαίνει στο φως των προβολέων. Επίσης για τα παραθυράκια. Ε, για τα παραθυράκια δεν υπάρχουν. Όχι. Τα προϊόντα μας τα προσφέρουμε στην ε, βιομηχανία της άμυνας, ε, στις κυβερνήσεις, ε, στους χειριστές δεδομένων γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι πελάτες μας ανησυχούν ακριβώς για τα παραθυράκια. Εδώ και χρόνια λοιπόν φροντίζουμε το πρόγραμμά μας που ονομάζεται GSP να επιτρέπει στις κυβερνήσεις να έχουν μια εξονυχιστική εικόνα για το τι συμβαίνει με τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούμε με όλες τις λεπτομέρειες για να είναι ήσυχε ότι δεν υπάρχουν παραθυράκια. Αυτό ήταν για μας ο καταλληλότερος μηχανισμός, προκειμένου να είναι βέβαιοι, αλλά και να καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούμε και δεν θέλουμε βεβαίω να δημοσιοποιούμε το τι γίνεται, εφόσον μιλάμε για απόρριτα στοιχεία. Και σε συμφωνία με μια κυβέρνηση που ε, θα μπορούσε να εξασφαλίσει και τα δικά μας ε, τελικά συμφέροντα και για τις πληρωμές. Δεν αλλάζει κάτι από τις ΗΠΑ στις άλλες χώρες εδώ. Εάν προκύψει εδώ ε, έρευνα, πολλέ φορέ, ε, και δεν μιλάω για την εξάρτητη επιβολή του νόμου, τι δυτικέ αρχέ ή τι αιτήσει ε, από υπηρεσίε, πρέπει να συγκεντρωθούν τα δεδομένα και αυτό απαιτεί κόστο. Υπάρχει κόστο. Ε, το κόστο αυτό ε, καλύπτουμε. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτό μάλλον ζητούμε. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτό είναι και το τρόπο να λειτουργεί το σύστημα. Οι αρχέ πληρώνουν εφόσον θέλουν να συλλέξουν δεδομένα. Εάν νομίζετε ότι εμεί ω εταιρεία παγκόσμια, διεθνή εντορία, δεν, δεν δεχόμαστε αρκετά σε αιτήσει, Τίποτα δεν μπορεί να σα επιτρέψει να καταλήξετε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Το κόστο που ζητάμε δεν σημαίνει ότι. τιμή που ζητάμε δεν σημαίνει ότι κάνουμε κάτι παράνομο. Και για τον ασφαλή λιμένα, ναι, όσο μπορούμε τον εφαρμόζουμε. Τώρα, εάν μπορεί να βελτιωθεί, ναι, ε, εντάξει, συζητιέται αυτό, αλλά. Να προσθέσω κάτι. Ε, από την πλευρά των καταναλωτών επιτυγχάνουμε όλο και περισσότερο τον ασφαλή λιμένα για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπη αλλά από την πλευρά των εταιριών για τους εταιρικούς μας πελάτες εφαρμόζουμε τις ρήτρε που ισχύουν ε, για τα θέματα συναλλαγών ε, για τον ιδιωτικό βίο στην Ευρώπη και τους σχετικούς κανόνες. Δεν μπορούμε τώρα να σας δώσουμε και περισσότερα από αυτά ως αποδεικτικά στοιχεία. Υπάρχουν και όρια, όρια Μπορεί να μην είναι όλα τέλεια, αλλά έχουμε και περιορισμού που δεν του έχουμε επινοήσει εμεί. Κύριε Λόντλαντ, ευχαριστώ. Έχουμε μια μακρά ιστορία του να λαμβάνουμε τέτοια μέτρα. Το 2006 ήμασταν από τι πρώτε εταιρείε που απευθύνθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνη όταν υπήρξε η πρώτη αίτηση για ε, αποκάλυψη στοιχείων. Και υπάρχει ένα νόμο για κράτηση στι ΗΠΑ, ίσω όμω τότε δεν είχε συνδυαστεί με αυτά τα στοιχεία. Πάντω από τότε πιέζουμε για τα θέματα αυτά, γιατί πιστεύουμε ότι οι κυβερνητικέ αιτήσει πρέπει να είναι περιορισμένε, να έχουν συγκεκριμένο στόχο, να είναι πλαισιωμένε και να υπάρχει συγκεκριμένο σκοπό, ε, να είναι επιλογημένε. Η πρώτη έκθεση μα για την διαφάνεια ήταν το 2010, πριν αρχίσουν οι άλλοι. Ήταν σημαντική κίνηση αυτή για εμά ω εταιρεία, για να βεβαιωθούμε ότι οι αποφάσει που λαμβάνονται είναι τεκμηριωμένε, ότι τα μέσα ασφαλεία, ε, η σκοπή ασφαλεία που χρησιμοποιούσε ιδεολογίε η κυβέρνηση είναι βάσιμη. Και να το γνωρίζει αυτό η κοινωνία των πολιτών. Να ξέρει ότι είναι εύστοχε οι αιτήσει και αναλογικέ με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Ε, Ω προ την εμπιστοσύνη. Ε, ναι, εδώ είναι διτό το ερώτημα όμω. Βεβαίω ε, το διαδίκτυο και η κοινωνία των πληροφορία διευρύνει το θέμα τη ε, εμπιστοσύνη. Αλλά το θέμα είναι πώ απευθύνεται κανεί στι κυβερνήσει και ρωτάει του πολίτε μπορούν να τι εμπιστευτούν. Ε, Θα έπρεπε να υπήρχε λοιπόν διαφάνεια. Αυτό ισχύει για τι ΗΠΑ. Θα θέλαμε να υπάρξει και μεταρρύθμιση του συστήματο και στην Ευρώπη, γιατί αυτό το λέει και η θεσμό περί διαφάνεια. Είναι ένα απλό βήματα, βήμα αποκάλυψη στοιχείων. Τι αιτήσει λαμβάνουμε, πόσε ε, συμμορφούνται με του κανόνε για την εθνική ασφάλεια και του επιδικόμενου σκοπού, να γνωρίζουν οι πολίτε το τι αποφασίζουν και να μπορούν να το βασίσουν σε κάποια στοιχεία. Εδώ γίνεται συζήτηση σήμερα για τα θέματα αυτά και συμμετέχουμε. Αυτό είναι μια απόδειξη. Θα συνεχίσουμε να ε, συμμετέχουμε γιατί το ζήτημα αυτό είναι για μα ζήτημα προτεραιότητα. Και για τα παραθυράκια και το θέμα τη αμοιβή θα συμφωνήσω με την Τόροφη. Δεν υπάρχουν παραθυράκια και δεν έχουμε λάβει. Ε, κανένα αντίτιμο για θέματα παρακολούθηση για τον ασφαλή λιμένα, ναι, εντάξει, σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί. Μπορεί να προσαρμοστεί στι ανάγκε που υπάρχουν κάθε φορά για ζητήματα εθνική ασφαλεία, λόγω χάρη αναπερίπτωση, αν πρέπει να τα εξετάσουμε και προσεκτικά, αλλά το σημαντικό μα πάει στο επίπεδο που έλεγα ότι πρέπει να ξεκινάμε, δηλαδή τι κυβερνήσει, το τι αιτήματα ε, υποβάλλουν, το τι πλαίσιο ισχύει για την προστασία τη εθνική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω την άλλη ερώτηση. Θεωρείτε ότι είναι αξιόπιστες ε, οι προδιαγραφές κρυπτογράφησης. Ε, αυτές οι ανοιχτές, ε, ανοιχτές που ελέγχονται είναι σχετικά αξιόπιστες, αλλά δεν είναι ισόβια αξιόπιστες τέτοιες προδιαγραφές κρυπτογράφησης. Θα πρέπει συνεχώς να τις βελτιώνουμε και να ζητούμε όλο και καλύτερες προδιαγραφές κρυπτογράφησης για να βελτιώσουμε την ε, ασφάλεια για το θέμα της κρυπτογράφησης. Σίγουρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αυξήσουμε το κόστος για την παραβίαση της, της ασφάλειας. Και η αντίδραση μερικές φορές στην απειλή της παραβίασης είναι καλύτερα συστήματα κρυπτογράφησης, μεγαλύτερο κόστος, αλλά μεγαλύτερο κόστος και για τον επίδοξο παραβάτη. Και φυσικά διαρευνούμε νέες τεχνολογίες γιατί μας ενδιαφέρει να φτάσουμε στο επόμενο αναβαθμισμένο στάδιο ασφάλειας και προστασίας. Τώρα για τη συζήτηση γενικά. Νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο. Δεν είμαστε εχθροί. Και όλοι πιστεύουμε στην ε, ελευθερία έκφρασης, ε, στο ελεύθερο διαδικτύο. Και όλες αυτές οι αποκαλύψεις, όλα αυτά τα στοιχεία που καθημερινά διαβάζουμε για τις εταιρείες είναι πόδινα και δραματικά και για μας. Και ε, βλάπτουν την εικόνα μας, βλάπτουν τις υπηρεσίες μας και κλονίζουν και την εμπιστοσύνη των ε, χρηστών στις υπηρεσίες μας. Γι' αυτό και πιστεύω θα πρέπει να συνεργαστούμε και είναι προς κοινό μας συμφέρον και όφελος να βελτιωθεί η κατάσταση. ό,τι αφορά τις πληρωμές, Εμεί στο Facebook δεν λαμβάνουμε πληρωμές ε, για τις αιτήσει που λαμβάνουμε από κυβερνήσεις. Βέβαια, κάποιοι ακτιβιστές για την ιδιωτική ασφάλεια έχουν τη λογική ότι αν χρεώνουμε τις κυβερνήσεις θα υποβάλουν λιγότερα αιτήματα. Είναι μια προσέγγιση κι αυτή. Πάντως, μέχρι στιγμής η πολιτική του Facebook είναι να μην δέχεται πληρωμές ε, για τα αιτήματα αυτά. Πάντως, είναι ανοιχτή η συζήτηση. Αν αξίζει να βάλουμε και αυτό το παράγοντα της ε, αμοιβή ή ε, να περιορίσουμε τα αιτήματα. Σε ό,τι αφορά τον ασφαλή λιμένα, εγώ θα προτιμούσα ως ε, πελάτης να έχω συναλλαγές με μια επιχείρηση που έχει προσχωρήσει στον ασφαλή λιμένα. Η ε, είναι σημαντικός ρυθμιστικός φορέας ε, και είναι ένας ρυθμιστικός φορέας πολύ αποτελεσματικός. Το θέμα βέβαια της εθνικής ασφάλειας εξαιρείται, αλλά κανονικά ο ασφαλής ε, λιμένας είναι αμφίδρομος. Και υπάρχει μια αντίστοιχη εξαίρεση και στην ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Είναι, είναι λογικό να μην περιλαμβάνει και την εθνική ασφάλεια ο ασφαλής λιμένας. Γιατί ακόμη και η νομοθεσία για την προστασία δεδομένων εξαιρεί την εθνική ασφάλεια ίσως θα πρέπει να τροποποιηθούν οι νομοθετικές διατάξεις για να περιλαμβάνουν και την εθνική ασφάλεια. Ίσως θα ήταν λογικό βήμα. Πάντως σήμερα η έννοια του ασφαλούς λιμένα δεν την καλύπτει. Γιατί ούτε οι αντίστοιχες κοινοτικέ διατάξεις περιλαμβάνουν την εθνική ασφάλεια στον ασφαλή λιμένα. Όταν μιλάμε για εθνική ασφάλεια, μερικές φορές γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφόρων κρατών. Τώρα, να περάσουμε στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις, στους τρεις τελευταίους παρόντες βουλευτές. Θα τις ακούσουμε όλες μαζί και μετά θα δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας για να απαντήσουν, για να ολοκληρώσουμε μέχρι τις 6.30. Έγκστρομ, Τόρβαλτς και μετά η κυρία Λάτφορτ. Κύριε Έγκστρομ. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση για την κυρία Πέλτς της Microsoft. Επανειλημμένα είπατε ότι δεν έχετε παραθυράκια στα προϊόντα σας και χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι. Τα περισσότερα από τα προγράμματά σας είναι κλειστής πηγής, δεν είναι δωρεάν. Δεν μπορεί κάποιος εξωτερικός, ανεξάρτητος, να ελέγξει ε, τι γίνεται στο ε, κομπιούτερ. Αυτή τη στιγμή τα έχετε εγκαταστήσει εσείς επιτρέπεται σε μερικές κυβερνήσεις να διαβάζουν το κώδικα της πηγής. Εντάξει, και ο κώδικας που τους αφήνεται να διαβάσουν δεν έχει παραθυράκια. Ε, αλλά επειδή είναι κλειστή η πηγή, ε, δεν ε, μπορεί κανείς να το διασταυρώσει. Στην αντίθεση όταν μιλάμε για Linux και τέτοια συστήματα δωρεάν ανοιχτή πηγή στο λογισμικό αυτό, δημοσιεύεται ο κωδικός και ο καθένας ε, που έχει τη δυνατότητα και την πραγματογνωμοσύνη να το ελέγξει, να το επαληθεύσει. Το open source λογισμικό ε, επαληθεύεται, ελέγχεται. Κανένα από τα δικά σας προϊόντα όμως γιατί είναι κλειστή πηγή. Επαναλαμβάνω λοιπόν και ρωτώ. Υποθετικά τελείω συζητάμε τώρα σε περίπτωση που η NSA ή κάποια άλλη υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών σας είχε διατάξει να βάλετε παραθυράκια σε κάποιο προϊόν, θα μπορούσατε τώρα, θα επιτρεπόταν να μας το πείτε μας εδώ σήμερα. <laughs> Τι ανέκδοτα λέτε, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Τόρβαλτς. Ευχαριστώ, Σόφη. Πρώτα απ' όλα, για να ξαναπάμε στη συνουσία. Όπως τα γνωρίζετε, στη Μασαχουσέτη. Υπάρχει μια μικρή πόλη με πολύ ενδιαφέρον όνομα. Υποψιάζομαι ότι όλοι εκεί έχετε κάποια σχέση με σε κάποιες οργανώσεις. Και θα το ρωτήσω λίγο διαφορετικά από τον συνάδελφο. Ο... Στο μεγαλύτερο γιο μου έκαναν την ίδια ερώτηση. Σας πλησίασε η NSA. Για τα παραθυράκια είπε όχι, αλλά δεν την ίδια στιγμή έγινε καταφατικά. Έτσι λειτουργεί το νομικό πλαίσιο. Δεν έδωσε την απάντηση που αναμενόταν και όλοι κατάλαβαν παρόλα αυτά, εάν τον είχαν πλησιάσει ή όχι. Και το τρίτο ερώτημα, το τρίτο πρόβλημα. Ο κύριος Μπέλτερ, Λάντλαντ είπε δεν υπάρχουν παραθυράκια. Ο κύριος Μπέλτς μάλλον είπε ότι δεν υπάρχουν παραθυράκια. Η κυρία Μπέλτς. Ε, τα παραθυράκια. Είναι διαφορετικό πράγμα από του κοριού. Διότι αν υπάρχουν κοριοί και έχετε κοριού στα προγράμματά σα, Αυτή η αυτοί οι παραθυράκια είναι. Και σίγουρα κάποιοι γνω, ε, κερδίζουν χρήματα από όλο αυτό. Χρηματοδοτούν τα παραθυράκια. Υποψιαζόμαστε ότι υπάρχουν εκατοντάδες παραθυράκια σε όλα αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τελευταία ερώτηση, ε, κύριε Λάρπορτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρόμοια γραμμή με αυτή που κι εσείς αναπτύξετε. Βεβαίως θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι ως προς τις κατηγορίες του τύπου για την μαζική συλλογή μεταδεδομένων μέσω του Prism και του Tempora. Αλλά ως προς τις σημερινές σας παρουσιάσεις, σαφώς, για μας είναι δυσχερές, δύσκολο μάλλον, να τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά. Σίγουρα κάποια πράγματα είναι ανακριβή, σίγουρα κάποιες καταχρήσεις έχουν γίνει, είναι απολύτως αδύνατο να το επαληθεύσουμε απλώς. Απλώ αυτό που κάπως με εντριγκάρει είναι τα λόγια που δύο από εσά χρησιμοποίησατε, τη φράση ότι δεν θα επιτρέπατε ε, την άμεση ή ανάρμοστη πρόσβαση στις υπηρεσίες σας. Ποιο είναι το ε, ε, αντίθετο δηλαδή, η έμεση αλλά αρμόζουσα. Τι εννοείται με το άμεση ή ανάρμοστη σαν τη συνουσία. Πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα, κυρία Μπέλτ. Ε, ναι. Αισθάνομαι λες και περνάω τεστ IQ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Τα πάντα έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη, είναι σαφές. Αλλά επίσης σαφές είναι ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Ε, κάτι για τις... Ε, για τα δεδομένα και για τις νομικές απαιτήσεις Για τις ανοιχτές διαδικασίες. Ναι, ανοιχτές είναι οι διαδικασίες εδώ και χρόνια, αλλά είναι ανοιχτές και σε αυτούς που έχουν αναπτύξει τα λογισμικά. Ε, έχουν αναπτύξει τα λογισμικά για να κάνουν ακριβώς αυτά που θέλετε. Είναι λοιπόν περισσότερο επισφαλής οι ανοιχτές πηγές αυτές, το open source, από ότι τα ελεγχόμενα λογισμικά πρώτον. Και δεύτερον, εάν θα μου επέτρεπε ένα σε να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, σας απάντησα. Δεν υπάρχουν παραθυράκια. Τελεία. Δεν μπορείτε να ζητάτε από την NSA. Μα η ερώτησή μου ήταν υποθετικά. Εάν υπήρχαν παραθυράκια, θα είχατε το δικαίωμα να το πείτε. Εάν υπήρχε, υποθέτω ότι δεν θα μπορούσα να το πω είναι μέρος του απορρίτου που πρέπει να τηρώ. Να μην αποκαλύπτω, εάν υπάρχουν παραθυράκια ή όχι. Ενδιαφέρον ερώτημα όμως το τι είναι παραθυράκι. θα έπρεπε εδώ να, είναι, να υπάρξει εντελεχή μελέτη για να το εξακριβώσουμε. Σημαίνει να είναι ευάλωτο ένα λογισμικό που δίνει τη δυνατότητα στην NSA να έχει πρόσβαση σε δεδομένα ή ουδήποτε. Δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Ναι, το λογισμικό μας έχει τα στοιχεία, όπως κάθε λογισμικό παγκοσμίω. Η δική μας όμως προσέγγιση ποια είναι, να προστατεύουμε τους πελάτες μας και όσο μπορούμε ακριβώς να καλύπτουμε αυτά τα ε, κενά. Ε, πολλοί θα προσπαθήσουν να τα εκμεταλλευτούν για να βλάψουν τους πελάτες μας. Βρίσκεται στον πυρήνα, ε, ε, στο είναι το γονότυπο της των εμπορικών μας ε, συμφερόντων να καλύπτουμε τα κενά αυτά για να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λανθασμένους σκοπούς. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα που συζητάμε, διότι κάποιες κυβερνήσεις ανά τον κόσμο θα προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν ε, τα ευάλωτα στοιχεία μιας ε, τεχνολο... ενός τεχνολογικού μέσου για να έχουν πρόσβαση σε πολιτικά δεδομένα. Αυτό όμως από την πολιτική πρόπτικη σας δεν μπορώ να τα απαντήσω εγώ. Εσεί είστε πολιτικοί. Εάν θέλετε να συζητήσετε κάτι σε κυβερνητικό επίπεδο, αν πρέπει να επιτρέπετε ή όχι, μπορείτε να το κάνετε. Αλλά δεν μπορούμε εμεί να το απαντήσουμε. Ούτε τα δεδομένα αυτά τα παράσχουμε, ούτε αυτέ τι τεχνικέ δυνατότητε προσφέρουμε σε άλλου για να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα των πελατών μα σε τέλο πάντων οποιοδήποτε, οποιοδήποτε τα δεδομένα, οποιοδήποτε χρησιμοποιεί τι ε, τεχνολογίες μας, τις υπηρεσίες μας για την άμεση ή ανάρμοστη πρόσβαση. Πρόσβαση προσφέρουμε στα δεδομένα των πελατών μας μόνον εάν υπάρχει σαφές συγκεκριμένο νομικό ευσταθόν και ε, δεδομένο και αν τα δεδομένα, ε, έτοιμα μάλλον και αν τα δεδομένα υπάρχουν τα συγκεντρώνουμε και τα προωθούμε. Εκτός μικροφώνου. Με συγχωρείτε ε, αλλά αυτό ακριβώς κάνουμε. Αυτό επίσης υποχρεώμαστε να κάνουμε βάσει του νόμου. Εδώ είμαστε για να ακολουθούμε και νόμους, όχι μόνο των ΗΠΑ, αλλά τον κόσμο, το, και του υπόλοιπου κόσμου. Ε, η, αν μας έλεγε η NSA, εδώ είναι η σερβερ, η μυστική σερβερ, για πηγαίνετε να δείτε τι θέλετε να δείτε. Αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Καμιά από τι εταιρείε που είναι εδώ δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Η ανάρμοστη πρόσβαση θα ήταν να υπάρχουν κατηγορίες και να βρισκόμαστε εμεί σε αυτή τη δύσκολη θέση που δεν μπορούμε να περασπιστούμε του εαυτού μα. Τη λέξη την ξέρω μόνο στα γερμανικά. Σε περίπτωση αμφιβολιών είναι υπέρ του κατηγορουμένου. Λοιπόν, ε, ε, εγώ ε, με ενδιαφέρει να συζητήσουμε πώς θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα της εμπιστοσύνης αντί να βρεθούμε σε μια κατάσταση πατ, ε, όπως το σκάκι, που δεν πρόκειται να βοηθήσει κανένα. Yes. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει ούτε άμεση ούτε άμεση πρόσβαση, ούτε δικαιολογημένη ούτε αδικαιολόγητη ανάρμοστη. Υπάρχει μόνο νομότυπο αίτημα τη κυβέρνηση που ελέγχεται και εξετάζεται περιπτωσιολογικά. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν υπάρχουν κερκόπορτε, δεν υπάρχουν παραθυράκια και το λέμε καθαρά και εξάστερα. Το ερώτημα όμω είναι εύστοχο γιατί επισημαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Εμεί λέμε κάτι, εσεί το ε, αφισβητείτε, αλλά δεν ε, μπορούμε να έχουμε πραγματική εικόνα για το τι συνέβη πραγματικά. Εμείς προσπαθούμε να σας πούμε την αλήθεια. Γι' αυτό θέλουμε περισσότερη διαφάνεια, κοινοβουλευτική εποπτεία, έλεγχο και φυσικά και δικαστική ε, εντολή, μια νομότυπη διαδικασία. Για να μπορούμε να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι όντως ε, σας λέμε την αλήθεια όταν δηλώνουμε ότι σας λέμε την αλήθεια. Κατά τη γνώμη σας, ε, προγράμματα σαν το πρίσμα και το τέμπρα δεν υπάρχουν. Εμείς δεν ακούσαμε κανένα τέτοιο πρόγραμμα, ε, δεν ακούσαμε τη λέξη πρίσμα πριν την αναφέρετε εσείς. Αλλά τα γενικά του χαρακτηριστικά τα διαβάσατε στον τύπο. Δεν σας λέει τίποτα ένα τέτοιο πρόγραμμα, σαν το πρίσμα. Δεν συμμετείχαμε σε κανένα τέτοιο πρόγραμμα, δεν έχουμε χορηγήσει. Ναι, αλλά δεν είχατε καμία ιδέα, δεν είχατε καν ιδέα ότι τέτοιου είδους προγράμματα υπάρχουν και ότι υπήρχε μαζική μεταφορά δεδομένων. Τέτοιου ίδιου ε, προγράμματα δεν υπάρχουν κατά τη γνώμη σας. Σε λάθος ε, άνθρωπο θέτετε την ερώτηση. Θα πρέπει να αποταθείτε στις ε, υπηρεσίες ασφάλειας των διαφόρων κυβερνήσεων. Ο κύριος Άλλαν, συμφωνώ με τον κύριο Λάντμπλαντ Τώρα, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Νομίζω ε, Δύο και δύο, αντί να καταλήγουν συμπέρασμα ότι κάνουν τέσσερα, κάνουν 25. Υπήρχε ένας, ε, μια πληροφορία για μαζική μεταφορά δεδομένων κάπου στι ΗΠΑ, Αυτό πριν τι αποκαλύψει του Edward Snowden Μετά έγινε μια συμπίληση όλων αυτών των ε, νομιογενών πληροφοριών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το, τον όρο που χρησιμοποίησα, το άμεση και ανάρμοστη, ε, δεν ήταν τυχαία η επιλογή αυτών των λέξεων, γιατί ε, ο τύπος διατηνόταν το αντίθετο. Εμείς χρησιμοποίησαμε ακριβώ την αντίθετη ορολογία από αυτή που χρησιμοποιούσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το άμεσα και ανάρμοστη. Το θέμα είναι ότι πόσε ε, ελάχιστες πληροφορίες θα δημοσιεύονται. Γιατί εμείς ε, το κάνουμε από δικής μας πλευράς και μερικές εταιρείε με πιο αργούς ρυθμούς, άλλοι με πιο αργούς ρυθμούς. Αλλά εμείς ξοδεύουμε χρόνο και χρήμα ε, δίνοντας στοιχεία για το πόσες αιτήσει λαμβάνουμε αυτοί που θέτουν τις αιτήσει, ε, οι δημόσιες διοικήσεις, ε, δεν ε, μπαίνουν στον κόπο να δημοσιεύσουν τέτοιες πληροφορίες για να δημιουργήσουν μια τεκμηριωμένη εικόνα οι πολίτες για το ποιος είναι την αλήθεια. Εμείς δίνουμε πληροφορίες για το τι αιτήσεις έχουμε λάβει, αλλά το θέμα είναι οι ίδιοι οι αιτούντες θα πρέπει να δίνουν στοιχεία για το πόσες αιτήσει μας έχουν καταθέσει. Τότε θα μπορούμε να κάνουμε μια αντιπαραβολή των στοιχείων και να μπορέσουμε να βάλουμε όλες τις ψηφίδες στο μοσαϊκό και να δημιουργήσουμε μια εικόνα για να δούμε αν οι ισχυρισμοί ήταν ακριβή ή όχι. Σα σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ε, αυτό μας φέρνει στο τέλο τη σημερινή συνεδρίασης. Ευχαριστώ όλα τα μέλη του πάνελ που ήρθαν και εκτέθηκαν ε, στην αγανάκτηση και στη ματέωση και απογοήτευσή μας, αλλά είναι προς αναζήτηση της αληθείας όλα αυτά. Ψάχνουμε να βρούμε και εμείς την αλήθεια. Ευχαριστώ όλους σας και τους διερμηνείς. Η επόμενη συνεδρίαση, 5η, 14 του μηνός το απόγευμα 3 με 6.30. Ελπίζω να σας ξαναδώ όλους τότε και ευχαριστώ.